Uh, so, um, και κύριοι, είμαστε αρκετοί παρόντε. Διάφοροι έφτασαν τα τελευταία λεπτά. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Θα ήθελα να πάρετε όλοι θέση, να λάβετε θέση. Γιατί έχουμε πολλά σημεία τα οποία πρέπει να διεκπαιρεώσουμε. Θα ήθελα να υιοθετήσουμε το σχέδιο μερίσιας διάταξη. επίσημα. Έχετε να προτείνετε αλλαγέ. Όχι, υιοθετείτε. Μεταδιδόμαστε από το ίντερνετ, όπως όλες οι συνεδριάσεις μας, βέβαια. Οποιοςδήποτε είναι συνδεμένος online τον καλωσορίζω. Έχουμε ένα νέο τεύχος του newsletter, ε, εσείς έχετε λάβει τα αντίτυπα και όσοι είναι συνδεδεμένοι μαζί μας ε, μέσω ίντερνετ μπορούν να το βρουν στο ίντερνετ, αν το επιθυμούν, και να παρακολουθούν τις εργασίες της ΙΜΚΟ. Έχουμε πρακτικά. Έχουμε τα πρακτικά της 1ης Φεβρουαρίου 2011, τα οποία έχουν υποβληθεί. Αν έχετε σχόλια να προτείνετε αλλαγές ή οτιδήποτε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης αύριο μπορείτε να το κάνετε. Προχωρούμε. Ε, επειδή τα δύο επόμενα θέματα είναι δικά μου, θα ήθελα η Μπερναντέτ να λάβει τη θέση του Προέδρου, παρακαλώ. Θα ήθελα τα δύο επόμενα σημεία να τα παρουσιάσει, να, σε αυτά να προεδρεύσει η Μπερναντέτ για να παρουσιάσω τις δύο μου εκθέσεις. Θέλετε να αλλάξουμε και θέση για να παρουσιάσω τις δύο μου γνωμοδοτήσεις. Ναι. Voilà, donc la mise en place est en fait. Πολύ ωραία, πήραμε θέση. Αντικαθιστώ προσωρινά τον Πρόεδρο για τις δύο του εκθέσεις και θα περάσουμε στην πρώτη από αυτές για τα ευρωπαϊκά δίκτυα ευρυζωνικότητας επένδυσης στην ψηφιακά τροφοδοτούμενη ανάπτυξη. Ο Πρόεδρός μας είναι ο εισηγητής του αφιών των λόγων. Λοιπόν, του λόγων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν όλους τους κοιόδης εισηγητές που συνσέφεραν στο πρώτο σχέδιο της έκθεσης. Ε, είχαμε μια καλή συνεδρίαση όπου κυκλοφόρησαν διάφορες ιδέες και νομίζω ότι ήμασταν στο ίδιο μήκος κύματος γενικά. Έχω κάποιες προτάσεις να σας κάνω σήμερα το απόγευμα. Οι γνωμοδοτήσεις όλος ιδιαίτερος εποφελούνται νομίζω πολύ από επιπρόσθετες τροπολογίες, γιατί όπως ξέρετε οι προϋποθέσεις είναι αυστηρές για τις νομοδοτήσεις. Οι προϋποθέσεις ε, οι χρονικές. Σε αυτή τη γνωμοδότηση για την ε, ανάπτυξη των νέων ε, δικτύων ευρυζωνικότητας και πρόσβαση σε δίκτυα οπτικών ινών, ήθελα να μιλήσω για τα δικαιώματα των χρηστών. Νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο έχουμε συνεισφέρει ως Επιτροπή και θέλω να τονίσω ένα-δύο θέματα ε, συνεχεία για αυτά τα δικαιώματα. Καταρχάς όμως, σε ό,τι αφορά την ενιαία αγορά, είναι σαφές ότι μία ανταγωνιστική υποδομή για τις επικοινωνίες, το οποίο σημαίνει υποδομή ευρεία ζώνης που θα βασίζεται κυρίω σε ένα δίκτυο οπτικών ινών αλλά και όπου οι ασύρματες συνδέσεις θα είναι πολύ σημαντικές νομίζω ότι θα βοηθήσουν πολύ να λειτουργήσει καλύτερα η ενιαία αγορά και να αυξηθεί η διασυνοριακή δραστηριότητα. Αυτά τα στοιχεία τα αναφέρω στην πρώτη τροπολογία και επίση για να, για να τονώσουμε τις επενδύσεις χρειαζόμαστε μια πλήρω λειτουργούσα και ανταγωνιστική αγορά. Αυτή τη στιγμή, μια και οι προπολογισμοί πιέζονται, θα πρέπει να μεγιστοποιήσουμε την αξία των επενδυτικών ευκαιριών, ούτω ώστε να επενδύσουμε οι δυνατόν σε συνδέσεις ευρεία ζώνη. Μιλάω λοιπόν για τι επενδύσει. για το άνοιγμα των δικτύων κυρίω. Ε, σε μια μεγάλη ζήτηση και ζητώ από τις κυβερνήσεις και τις δημόσιες αρχές να λειτουργήσουν, να συνεργαστούν με τους παρόχους ε, διαδικτυακών υπηρεσιών, ούτω ώστε να βελτιώσουμε την, ε, το δυναμικό ενός δικτύου. Ούτως ώστε να έχουμε, ας πούμε, έξυπνα δίκτυα, ε, να έχουμε ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας ή δημόσιες προμήθειες ηλεκτρονικώς Όλα αυτά νομίζω θα κάνουν τις επενδύσεις πιο ελκυστικές. Και αν τα συνδυάσετε με άλλα πράγματα που μας ενδιαφέρουν, σε διάφορες άλλες μορφές υποδομών, νομίζω ότι θα μειωθεί το κόστος για τους χρήστες. Γιατί το σημαντικό ε, για την ευρεία ζώνη είναι πόσο κοστίζει στον συντρομητή. Όταν έχουμε λοιπόν ε, μείωση των ε, επενδύσεων, όπου δεν κάνουμε επενδύσεις ειδικά σε περιοχές της υπαίθρου, νομίζω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε ένα ελκυστικό πακέτο επενδύσεων. Παράλληλα, θα χρειαστούμε φυσικά κάποια δημόσια στήριξη. Αυτό συμβαίνει σε πολλές χώρες, αλλά το πλαίσιο, δηλαδή τα κριτήρια για τις κρατικές ε, ενισχύσεις και θα πρέπει αυτά όλα να ανοίξουν στον ανταγωνισμό, δηλαδή να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των παρόχων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το τελευταίο θέμα αφορά τα δικαιώματα ακριβώ των χρηστών. Νομίζω ότι θα πρέπει να, να προσπαθήσουμε να ενδιαφερθούν οι καταναλωτές ε, στις υπηρεσίες ε, ευρυζωνικότητας. Το πρώτο από τα που πρέπει να κάνουμε είναι να τους δώσουμε περισσότερες πληροφορίες, πιο ακριβείς πληροφορίες για το είδος της υπηρεσίας που λαμβάνουν αυτή τη στιγμή. Ε, οι ρυθμιστικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, η Ofcom, ε, συνέγραψαν μία μελέτη α, που δείχνει ότι οι καταναλωτές μειώνονται, α, μειώνεται η ταχύτητά τους, ταχύτητα σύνδεσής τους και αυτό είναι απαράδεκτο. Ε, και υπάρχει στα δικαιώματα των ε, καταναλωτών ε, στα πλαίσια της μεταρρύθμισης που εσείς περάσατε και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες για τις συνδέσεις, για τις υπηρεσίες οι καταναλωτές, οι συνδρομητές. Η ταχύτητα της ευρεία ζώνης είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και ζήτησα τις ρυθμιστικές αρχές την τις Ευρωπαϊκές Ρυθμιστικές Αρχές για τις τηλεπικοινωνίες στην ΠΕΡΕΚ, ε, την οποία υποστηρίζουμε εμείς ως Επιτροπή και ως Κοινοβούλιο, να, κάνουν κάποιους, ε, να βγάλουν κάποιους κανόνες για την ε, ταχύτητα της ευρείας ζώνης, ούτως ώστε να καταλαβαίνουν οι καταναλωτές, οι χρήστες, την ταχύτητα που τους δίνουν γιατί με αυτόν τον τρόπο θα ενδιαφερθούν πιο πολύ για ένα ελκυστικό ε, πακέτο που να βασίζεται σε οπτικές σύνες. Οι διαφημιζόμενες ταχύτητες ε, σε ένα δίκτυο οπτικών ινών είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που στην πραγματικότητα υπάρχει. Και αυτό είναι πρόβλημα. Η διαφημιζόμενη λοιπόν ταχύτητα είναι πολύ μεγαλύτερη από την πραγματική. Επίσης, ε, κάποια θέματα για την ε, ουδετερότητα και, την, ε, και το άνοιγμα του ίντερνετ. Έχω κάνει κάποια σχόλια. Θα πρέπει να έχουμε υψηλότερο δυναμικό βριζονικότητα, ούτω ώστε οι πάροχοι να μην χρησιμοποιούν μέτρα κατά του ανταγωνισμού, Τώρα οι διατάξεις που υπάρχουν στην οδηγία για τις τηλεπικοινωνίες και που αρχίζουν οι ρυθμιστικές αρχές να εφαρμόζουν είναι κατάλληλες προς το παρόν, αλλά θα πρέπει να εξακολουθούμε να, να παρακολουθούμε όλη την κατάσταση. Σε πολλές χώρες λοιπόν τώρα οι πάροχοι υπηρεσιών ε, δίδουν πολύ περισσότερες πληροφορίες για το πώ διαχειρίζονται τα δίκτυα στου ε, καταναλωτέ. Υπάρχει μια πρόσφατη ε, συμφωνία στον Ηνωμένο γιατί είναι η πρώτη χώρα που μετέφερε στην εσωτερική τη νομοθεσία αυτό, για πιο ανοιχτό ε, στυλ και είδο πληροφοριών στου καταναλωτέ, για το τι δηλαδή του δίνουμε σε επίπεδο ευρυζωνικότητα και το, τι κάνουμε, πώ παρέχονται υπηρεσίε σε περίπτωση που υπάρχει συμφόρηση. Πάρτε λίγο, σε παρακαλώ. very good report. Thank you. Ελπίζω ότι εν τέλει με τη δική σας συνεργασία η έκθεση θα είναι εξαιρετική. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Μάλκολμ και για τα σχόλια που μας παρουσιάσατε αλλά και για όλη την εργασία. Θα δώσω τον λόγο τώρα στους διαφορούς σκιώδης εισηγητές και πρώτα η κυρία Κοράτσα Μπίλτ η οποία αντικαστά την κυρία Κόρχολα. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που μπορώ να σας παρουσιάσω τις απόψεις της φίλης ε, κυρίας Κόρχολα η οποία υποστηρίζει απολύτως την θαυμάσια εργασία του κ. Χάρμπορ που δείχνει ότι κατανοεί τα θέματα των επενδύσεων των δικτύων μεγάλης ταχύτητας και ευρυζωνικότητας που πρέπει να αναπτυχθούν για να αυξηθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και να δημιουργηθεί απασχόληση. Η κυρία Κορχόλα τονίζει την σημασία του ανταγωνισμού στην αγορά ώστε να υπάρξει, να είναι αρκετά ευθυνές οι τιμές για τους καταναλωτές και ταχύ εφαρμογή από πλευράς ε, κρατών μελών και των σχετικών αρχών των ε, πλαισίων που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης αναμένει ένα πρόγραμμα πλαίσιο πολιτικής και υπενθυμίζει σε όλους ότι αποτελεί σημαντικό μέρος της προώθησης της ε, ψηφιακής ατζέντα στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει η Προεδρεύουσα κυρία Βερνιού. Ο κύριος Κορέι Κάμπος. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Μάκομ Χάρμπορ για τη δουλειά που έκανε στη συνεισφορά αυτής της γνωμοδότησης που είναι πολύ πλούσια και σημαντική και θέλω να τον ευχαριστήσω κυρίως για το ότι έλαβε υπόψη τις προτάσεις που έκαναν οι σκιώδεις εισηγητές στην συνάντηση που είχαν για το e-commerce, το ηλεκτρονικό εμπόριο και για την πολυμορφία των πολυμέσων στην τεχνολογία και για τις πιο υπερπεριφερειακές περιοχές. Αυτή η ανακοίνωση είναι πολύ καλοδεχούμενη στο μέτρο που αναγνωρίζει τα ωφέλη της ευρυζωνίας και έχει έτσι και τους στόχους μιας στρατηγικής. Η ευρυζωνική επικοινωνία θα είναι μία από τις, ένας από τους αυτοκινητοδρόμους της επικοινωνίας που θα προωθήσει φυσικά, θα πρέπει να προωθηθεί και η υποδομή που θα αυξήσει αυτή την τάση και θα αυξήσει και την απασχόληση. Και έτσι θα μειωθούν οι δαπάνες φυσικά, δαπάνες συναλλαγών σε σχέση με αυτό το δίκτυο. Και θα γίνει φυσικά χρήση των τεχνολογικών προτεραιμάτων. Η επικοινωνία αυτή, η ανακοίνωση αυτή σε σχέση με το δυναμικό και τις ε, ελλείψεις στην αγορά θα πρέπει να καλύψει τις προϋποθέσεις για να μπορούν να συναλλάσσονται οι, ε, όσοι εμπλέκονται. Επίσης η ανακοίνωση ή καλύτερα είναι αναγκαίο να βελτιώσουμε την προσπελασιμότητα στα κονδύλια των υποδομών για αυτές τις υποδομές ε, ώστε να μπορέσουμε να πάμε πέρα από τις ε, προσδοκίες και πρέπει να ταυτοποιήσουμε και να άρουμε τα εμπόδια ο τομέας, ο δημόσιος τομέας έχει ρόλο να διαδραματίσει για την προώθηση των υποδομών που πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη ζήτηση και την προσφορά και να ρυθμίζει την ισορροπία. Και θα πρέπει να έχει τεράστια επίπτωση και στην ε, εκπαίδευση και στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στην ε, διασυνδεσιμότητα ώστε να υπάρξουν κίνητρα για τις ε, αγορές και να μπορέσει να ανακάμψει η οικονομική ανάπτυξη. Αυτά είναι θεμελιώδεις στόχοι. Με τον ίδιο τρόπο όσον αφορά τη διασύνδεση σε ευρυζωνικά με τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τα, τις δημόσιες υπηρεσίες και μέσω των δημόσιων προμηθειών θα πρέπει με καινοτόμο τρόπο να δράσουμε μέσω του e-help, e-education, ηλεκτρονική εκπαίδευση και κατάρτιση μπορούν να δώσουν πολύ θετικά αποτελέσματα τεχνολογικά στην αναζήτηση υπηρεσιών ευρυζωνικά. Θα υποβάλουμε τροπολογίες και επενούμε και συγχαίρουμε τον συντάκτη γνωμοδότησης για το έργο του. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Μάντερς είναι απόν. Α, εσείς κύριε Κρότσμαν. Κυρία Πρόεδρε, λυπούμε πολύ. Είχε πει ότι θα έλθει. Δεν μου έχει αναθέσει να πω τίποτε. Λυπούμε. Δεν πειράζει. Όταν έλθει θα του δώσουμε το λόγο έστω και αν έλθει αργότερα. Και αν δεν έλθει θα σας δώσω εσάς το λόγο. Τώρα, εκ μέρους, των Πρασίνων, ο κ. Έγκστρομ δεν είναι παρόν. Α, εσείς, κυρία Μπίλε Ευχαριστώ, κύριε Χάρμπορ, που θέσατε για παράδειγμα το ζήτημα της ουδετερότητας του δικτύου που ήταν μέγα θέμα στην συζήτηση που είχε γίνει για τις καθολικές υπηρεσίες. Θέσατε και το θέμα των κρατικών ενισχύσεων που ακόμα αποτελούν πρόβλημα για ορισμένες χώρες μέλη και όπου η σχετική ενημέρωση δεν είναι σαφής. Έχουμε κενά στην Ήπεθρο σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην ευρυζωνική επικοινωνία και ούτε έχουν ακόμη ολοκληρωθεί τα σχετικά μέτρα. Χαίρομαι που μπαίνουν στο παιχνίδι και τα, οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί χρηματοδοτήσεων. Α, βλέπω τον κύριο Μάντερ που καταφθάνει, Αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο για μα. το συνόλο λοιπόν υποστηρίζουμε την έκθεσή σα, του κύριου Χάρμπορ δηλαδή, είναι καλή, θέτει σωστά τα θέματα και θα δούμε ίσως στις λεπτομέρειες αν χρειαστεί να υποβάλουμε κάποιε τροπολογίες. Αλλά πάντως στις γενικές γραμμές ε, μας ικανοποιεί και τον ευχαριστούμε. Καλά λοιπόν, ο κύριος Μάντερς ήλθε, θα του δώσω λίγο χρόνο να ε, εγκατασταθεί στο έδρανό του και το λόγο θα βάλει λάβει πρώτα ο κύριος Ντεγιούγκ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ τον Μάλκολμ Χάρμπορ για την γνωμοδότησή του που περιλαμβάνει ορθά πράγματα. Έχω και λίγες ερωτήσεις και κάποιες προσθήκες ερωτήσεις ως εξή. Αφενός χρειάζεται ανταγωνισμός, βέβαια, και ως καταναλωτής έχω καμιά φορά την εντύπωση ότι δεν μου προσφέρονται αρκετές επιλογές. Γνωρίζω την κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου καμιά φορά ο πάροχος της υπηρεσίας έχει τόσο μεγάλο μερίδιο της αγοράς, που είναι και δύσκολο να βρει κανείς άλλον. Και δεν είναι και πολύ διαφορετικά τα πράγματα και στην Ολλανδία. σε αυτό εννοείται στην πρώτη σας παράγραφο και εάν, εάν είναι όντω αυτό θα συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά έχουμε και μέρη της χώρας, κυρίως σε μεγαλύτερες χώρες, με απομακρυσμένες περιοχές ή νησιωτικές περιοχές, όπου ίσως να μην είναι κερδοφόρα η υπόθεση αυτή ε, για να επενδύσουν οι επιχειρήσεις. Και εκεί νομίζω πρέπει να παρέμβει το κράτος. Διότι όλο και περισσότερο βλέπουμε την πρόσβαση στην ευρυζωνικότητα ως θεμελιώδης δικαίωμα. Όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση όπου και αν κατοικούν. Δεν βλέπω πολλά σχετικά με, τη, αυτό στη γνωμοδότηση ότι υπάρχει απέτηση, αξίωση α, ε, από τον, κατά των χωρών μελών δηλαδή για να προσφέρουν τις επενδύσεις αυτές, την, την στήριξη αυτή. Καθώς επίσης και κοινοπραξίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την λειτουργία των δικτύων. Δεύτερη ερώτηση ταχύτητα του διαδικτύου. Όντως στην πράξη δεν νιώθει κανείς, δεν βλέπει την ίδια ταχύτητα όπως αυτή που διαφημίζεται. Ταυτόχρονα ποικίλει από ιστοσελίδα σε ιστοσελίδα. Εγώ έχω διαδίκτυο οπτικών ινών ε, στο σπίτι μου με πολλά μεγαμπάιτα ένα δευτερόλεπτο με ναι, πολύ καλή δηλαδή ποιότητα πρόσβασης. Όταν επισκέπτομαι όμω ορισμένε ιστοσελίδε. βλέπω ότι η ιστοσελίδα είναι συμφορημένη, όχι τόσο το κέντρο του παρόχου της υπηρεσίας. Διερωτώ με πώς μπορεί να ισχύσουν οι γενικοί κανόνες αφού υπάρχει διαφορά από ιστοσελίδα σε ιστοσελίδα. Δεν ξέρω πώς ίσως μπορούμε να το καταστήσουμε σαφέ αυτό στην ε, αντίστοιχη παράγραφο. Τώρα, για το ηλεκτρονικό εμπόριο και όπου η Επιτροπή μας έχει συμφωνήσει ξανά στο παρελθόν για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις χρειάζεται ιδιαίτερη μνήμα γιατί για αυτές δεν είναι πάντα εύκολο να ξεκινήσουν δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου και βεβαίως αυτό είναι προς το συμφέρον το δικό μας και γενικότερα της ενιαίας αγοράς να μπορούν να το κάνουν. Άρα χρειάζονται διευκόλυνση. Ξέρω ότι η Επίτροπος Κρούς εξετάζει το θέμα αυτό. Χρειάζονται λοιπόν στήριξη με προσφορά λογισμικού ε, με τρόπους για να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου και νομίζω ότι τα όσα ήδη έχουμε συμφωνήσει μπορούν να προσθεθούν και στο κείμενο της έκθεσής σας. Και τέλος, υπάρχουν ορισμένε ομάδες ανθρώπων, όπως οι ηλικιωμένοι, που έχουν ανάγκες που χρειάζονται ειδική κάλυψη. διότι ίσως οι ίδιοι δυναμοί δεν αντιλαμβάνονται αμέσως ε, την ανάγκη, αλλά η ηλεκτρονική υγεία για παράδειγμα. Ιδιαίτερα για ειδικευμένους ανθρώπους η ευρυζωνικότητα έχει μεγάλη σημασία και θα έχει μεγαλύτερη στο μέλλον. Αυτές λοιπόν οι λίγες ερωτήσεις νομίζω όμως ότι συνολικά είναι ε, καλή η γνωμοδότησή σας. Η Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Μάντας. Ναι, ευχαριστώ. Η ευρυζωνικότητα είναι και θα είναι σημαντική. Διότι πρόκειται για επικοινωνία. Πολύ σημαντικό βέβαια θέμα. Ο μάλκον Μίδη έχει μεταφέρει μερικές από τις ιδέες μου στην γνωμοθέτησή του και τον ευχαριστώ. Είναι γνωμοδότηση βέβαια και ελπίζω η Επιτροπή Βιομηχανίας να μεταφέρει, να αντιγράψει τις δικές μας ιδέες στο κείμενό της. Γιατί θέλουμε μια ενιαία αγορά που να λειτουργεί. Και βλέπω συχνά να συντάσσονται μεν γνωμοδοτήσεις, αλλά οι αρμόδιες επί της επιτροπές δεν τις υιοθετούν. Ελπίζω τούτη τη φορά να γίνει. Διότι όπως είπα είναι πολύ σημαντικό θέμα, ενημέρωση δηλαδή όλων των καταναλωτών, πρόσβαση στην πληροφορική όλων των καταναλωτών, όλων των πολιτών. Λίγο πολύ αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ. Άρα μίλησαν όλοι οι Σάντου, η κυρία Σίτλερ, Στίλερ. Ευχαριστώ, ε, κυρία μου, ευχαριστώ και τον εισηγητή. Καλή δουλειά κάνατε, Μάλκολμ και ιδίως από τη σκοπιά της Επιτροπής μας το ζήτημα της, του ανταγωνισμού στην αγορά και κυρίως όταν έχει μέγα μερίδιο αγοράς ένας πάροχος υπηρεσιών δεν είναι υγιές αυτό για τους καταναλωτές για τις ίνες, για τις οπτικές ίνες αυτό που χρειάζεται να είναι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να είναι ανοιχτά προσβάσιμο. Είναι σημαντικό αυτό. Το ζήτημα της ουδετερότητας με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη Υπάρχουν και, ζήτημα μιας και, και ζητήματα μιας και μιλάμε για πρόσβαση καταναλωτών γιατί υπάρχουν ε, πολλές ε, προκλήσεις περιφερειακές και άλλες. Η ιδέα αυτή λοιπόν όπου θα έχει σε ένα σημείο το χωριό ένα ψηφιακό κέντρο ανά 2.000 κατοίκους δηλαδή Αυτό θα πρέπει να το προωθήσουμε όσοι εξημών εκπροσωπούμε καταναλωτές εν τέλει, για να έχουν πρόσβαση, γιατί δεν θέλουμε να υπάρχει ψηφιακό χάσμα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ψηφιακό σχίσμα. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ώστε οι πολίτες που εκπροσωπούμε να έχουν πρόσβαση. Αυτό λοιπόν το ψηφιακό πηγάδι του χωριού είναι σημαντικό για να βοηθήσει ανθρώπους σε περιφέρειες ώστε να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε αυτή την ψηφιακή επανάσταση. Κανένας από εμά δεν είναι στη γενιά που αποκαλείται στα αγγλικά digitally native, αυτοί που γεννήθηκαν μέσα στο διαδίκτυο. Αλλά αντιλαμβανόμαστε ποια είναι η σημασία. Τώρα για την ηλεκτρονικές, για τις ηλεκτρονικές προμήθειες επίσης είναι πολύ σημαντικό. Τώρα στα Highlands και Islands η, τα σχολεία έχουν πρόσβαση στην ευρωζωνικότητα. Αλλά οι κοινότητες όταν είναι κλειστά τα σχολεία δεν έχουν πρόσβαση στον πόρο αυτό. Βρισκόμαστε τώρα σε ε, ψηφιακή εποχή και μιλούμε για περιφερειακές. Όταν ε, λοιπόν γίνονται διαγωνισμοί δεν έχουν πρόσβαση. Πρέπει να μπει αυτό μέσα. Τέλος πάντων ευχαριστώ εν τέλει τον Μάλκον για το κείμενό του, έχει καλύψει πάρα πολλά θέματα και τα σχόλια των συναδέλφων επίσης, επίσης εμπλούτησαν την ε, συζήτηση. Ευχαριστώ. Όλοι οι βουλευτές που πήραν το λόγο Μάλκομ νομίζω ότι είπαν ότι ήταν θαυμάσια η δουλειά σου. Ο κύριος Φρανκ Μάσερ είναι ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Εύκολα, εύκολη δουλειά μου, δεν έχω να πω πολλά. Και η γνωμοδότηση του Μάλκομ και τα σχόλια που άκουσα μας βρίσκουν απολύτω σύμφωνους. Όχι μόνο εντοπίσατε τα τμήματα της ανακοίνωσης που θεωρούμε ότι είναι σημαντικά, αλλά τονίσατε και τι γίνεται τώρα και τι θα γίνει μετά στην ψηφιακή ατζέντα. Από πού ξεκινήσαμε. Αυτή η ανακοίνωση είναι τμήμα της ψηφιακής ατζέντα, που είναι μία από τις πρωτοβουλίες της ε, Ευρώπης 2020. Ο βασικός στόχος της δουλειάς μας είναι θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Και ξέρω ότι πολλοί από εσά ε, τονίσατε τη σημασία αυτού του πράγματος και τη σημασία μιας ε, πλήρως λειτουργούσας και ανταγωνιστικής αγοράς που μπορεί να δημιουργεί Θέσει απασχόληση και πραγματικά λειτουργεί με ενιαίο τρόπο στην Ευρώπη. Να τονίσω και εγώ κάτι που είπατε και εσείς με διαφορετικό τρόπο μεταξύ σας. Το να χαμηλώσουμε, το να μειώσουμε το κόστος των επενδύσεων. Εκτιμούμε ότι θα χρειαστούμε 250 δισεκατομμύρια ευρώ για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Ξέρουμε πολύ καλά τις δημοσιονομικές πιέσεις και τη λιτότητα που αντιμετωπίζουν περισσότερες ευρωπαϊκές ε, κυβερνήσεις. Ε, η μείωση του κόστου των επενδύσεων είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει και η γνωμοδότηση να το τονίζει και αυτό είναι θετικό που το αναφέρει. Τώρα τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Η Κομισιόν έκανε μια δημόσια διαβούλευση για την ουδετερότητα του δικτύου και για τις καθολικές υπηρεσίες. Και περιμένουμε να προκύψει κάποια δήλωση στο εγγύς μέλλον μετά τη δημόσια διαβούλευση. Οι συνάδελφοί μου στη Γενική Διευθύνση Ανταγωνισμού δουλεύουν για την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις. Θα τις έχουμε το 2012, τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές. Αυτά τα λέω για να ενημερώσω την Επιτροπή σας. Τέλος, θέλω να σχολιάσω αυτό το ψηφιακό πηγάδι. Η Κομισιόν σχεδίασε τους στόχους στην ανακοίνωση για την ευρυζωνικότητα, ειδικά για να αποφύγουμε αυτό το ψηφιακό πηγάδι. Θέλουμε 30 ε, MB το δευτερόλεπτο για όλους στην Ευρώπη μέχρι το 2020 και 50% των οικοκυριών να έχουν 100 MB το δευτερόλεπτο. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη είναι μεταξύ των καλύτερων, ότι έχουμε ανταγωνιστική υποδομή που θα ανταγωνίζεται στην παγκόσμια αγορά και ότι κανένα δεν θα μείνει πίσω. 30 Mbit για όλους και τα νησιά και τα Highland της Ιρλανδίας και όλη την Ευρώπη γενικά, όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά κυρίε και κύριοι και ευχαριστώ. Να μιλήσω για το χρονοδιάγραμμα πριν δώσω το λόγο στο Μάλκομ για να ολοκληρώσει. 24 Μαρτίου είναι καταληκτική ημερομηνία για τις τροπολογίες. Πλησιάζει. Θα εξετάσουμε τις τροπολογίες στις 13 Απριλίου και θα ψηφίσουμε στην ΙΜΚΟ επίσης στις 13 Απριλίου, την ίδια μέρα δηλαδή. Θα ψηφίσει η Ήτρε στις 5 Μαΐου και θα συζητηθεί το θέμα στην Ολομέλεια κατά πάσα πιθανότητα του Ιουνίου. Μάλκομ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την υποστήριξή τους, αλλά και για κάποιες πρόσθετες ιδέες που υπέβαλα. Και σίγουρα μέχρι την Πέμπτη θα υπάρξουν και κάποιες τροπολογίες που θα είναι ενδιαφέρουσες. Υπήρξε πολύ καλή ανταπόκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σημειώνω την παρατήρηση και ρωτήθηκαν και ερωτήσεις σχετικά. Οι στόχοι θα έλεγα όσον αφορά το ευρυζωνικό φάσμα ε, αφορούν τα κράτη-μέλη. Τώρα, αν χρειαζόμαστε νομοθετικό έργο, αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστή πρόταση που θα υποβληθεί στην Κοινοβουλευτική μα Επιτροπή. Και έχουμε και συνάδελφο που έχει αναλάβει την πτυχή αυτή. Το θέμα του ανταγωνισμού είναι σημαντικό θέμα, θα έλεγα, επειδή είναι σαφέ ότι από την μεταρρύθμιση, το πλαίσιο μεταρρύθμισης των τηλεπικοινωνιών, ότι σε τομεί όπου υπάρχει ένα πάροχο ινών πρέπει παρόλα αυτά να είναι διαθέσιμο και σε άλλους ε, που εμπλέκονται στην ε, αγορά και σε σχέση με την μη διακριτική μεταχείριση. Εκεί ακριβώς ε, ο ανταγωνισμός, οι συμφωνίες για τον ανταγωνισμό θα διαδραματίσουν τον ρόλο τους διαμορφώνοντας αυτό το πλαίσιο και θα πρέπει εδώ να υπάρξει και προσέλκυση και των επενδύσεων κάποιες χώρες ε, υπάρχει ήδη κάποιο πρότυπο γι' αυτό. Αυτή είναι η βάση με την οποία πρέπει να προχωρήσουμε προς το μέλλον. Και σε σχέση και με τις δημόσιες αρχές ε, όπως ε, επενδύουν, θα έπρεπε να είναι διαθέσιμο αυτό το πλαίσιο σε ανταγωνιζόμενους παρόχους. Και σε πολλές χώρες και στο Ηνωμένο Βασίλειο μία από τις πιο ανταγωνιστικές επιλογές σας σε σχέση με τους παρόχους, ακόμα και καλωδιακά που μπορούν να ανταγωνιστούν τις ε, οπτικές ε, ίνες. Ε, και αυτό το πλαίσιο ανταγωνισμού ανοίγει και η επόμενη γενεά πάλι στο ευρυζωνικό θα προχωρήσει. Και ένας συνδυασμός είναι κοινό, αυτό ήταν η παρατηρήσή μου χρειαζόμαστε μια τεχνολογική προσέγγιση, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχουν συνδυασμοί τεχνολογιών που θα είναι διαθέσιμοι και στις πιο απόμακρες περιοχές της Ένωσης θα είναι προσπελάσιμη η δορυφορική μετάδοση. Να το θυμόμαστε αυτό. Καλό θα είναι να μου αποστείλουν κάτι τις τροπολογίες τους οι συνάδελφοι. Και αναλαμβάνοντας, δίνοντας συνέχεια στην πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπάρξει κάποια πίεση όσον αφορά τον Επίτροπο για τον Ανταγωνισμό να υποβληθούν οι προτάσεις του σχετικά γοργά. Διότι χρειαζόμαστε αυτό το πράγμα, όπως και η κυρία Βερνιό το παρατήρησε επίσης και τα άλλα θέματα. Ελπίζω ότι θα καλυφθούν και από τις τροπολογίες σας ή και από τις δικές μου και ολοκληρώνοντας σε σχέση με αυτό που είπε η κυρία Κόρολα και η κυρία Κοράτσα θα έπρεπε να έχουμε μία ή δύο τροπολογίες για το ραδιοφάσμα που θα προσπαθήσουμε να είναι συμβατές και με τη δική της τροπολογία, διότι οι μεγάλες αποφάσεις για την απελευθέρωση του ραδιοφάσματος θα έχουν κέρια σημασία για την ευρυζωνικότητα και υπό τους όρους ε, της τέταρτης ε, γενεάς δικτύων και τεχνολογίας, αλλά και για τις τοπικές σύνδεσεις Wi-Fi. Να το λάβουμε υπόψη. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις σας, τις προτάσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα δουλέψετε πολύ σήμερα, γι' αυτό λοιπόν θα σας ξαναδώσω το λόγο για την δεύτερη έκθεση, είναι πολύ σημαντική, για την νέα εμπορική πολιτική για την Ευρώπη, στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρώπη 2020, πολύ σημαντικό θέμα. Μάλκομ, ξανά εσύ. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε και με μια διαφορετική τώρα εδώ προσέγγιση. Δίνω κάνω ένα πρόλογο πρώτα απ' όλα λέγοντας ότι με μεγάλη χαρά είδα ότι συμφώνησαν οι συντονιστές να υπάρξει έκθεση γιατί όπως όλοι γνωρίζετε, η δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή απομίζεται τις ευθύνες της στην παγκόσμια σκηνή με ιδιαίτερη σοβαρότητα και είναι σαφές ότι οι εξελίξεις στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά δεν τεκταίνονται ε, σε ένα στεγανό πλαίσιο και σε απομόνωση, αλλά βρισκόμαστε σε ένα δίκτυο εμπορικών ε, πλεγμάτων και σχέσεων. Και είχαμε πάει σε αποστολές ε, στην Κίνα, Ινδία, στη ΣΥΠΑ, και για να συζητήσουμε κάποια από αυτά τα πράγματα. Και πάλι εδώ επικεντρώθηκα σε αυτό που είναι μια πολύ καλή και ευρία έκθεση σε τομείς που θεώρησα ότι ήταν σημαντικές σε συνεισφορές ε, στα θέματα της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής. Πρώτον, δεν θα εκπλαγείτε να δείτε ότι η τυποποίηση και ότι η ανάπτυξη των ε, τυποποιήσεων ε, προχωρούν. Και από πλευρά τη τυποποίηση και των προδιαγραφών πρέπει να είναι σαφέ ότι οι προδιαγραφέ και η τυποποίηση, ιδιαίτερα για τι παγκόσμιε αυτέ διατάξει, έχουν κέρια σημασία για το παγκόσμιο εμπόριο. Επιπλέον όμως ιδιαίτερα σε σχέση με την, ε, το έργο μας με τις ανεπτυγμένες αγορές ε, και τους εταίρους, ε, οι προδιαγραφές γίνονται όλο και πιο σημαντικές. Διότι πολλές φορές, ιδιαίτερα σε σχέση με τις ΙΠΑ και την Ιαπωνία, βλέπουμε πολλές περιπτώσεις όπου απογοητεύονται σε σχέση με τους εμπλεκόμενους. Υπάρχει απογοήτευση για τις διαφορετικές προδιαγραφές και τυποποίησεις που ισχύουν σε σχέση για παράδειγμα και με το περιβάλλον ιστορικά σε σχέση με τη διαφορετική υιοθέτηση ε, και διαφορετικές απόψεις που διέπουν αυτά τα πλέγματα. Χρειάζεται όμως ε, μια πολιτική πίεση και μια πολιτική ευαισθητοποίηση για να προχωρήσουν αυτά τα πράγματα συνολικά. Διότι διαφορετικές προδιαγραφές και διατάξεις ε, να που προσπαθούν να επιτύχουν τον ίδιο στόχο προκαλούν αυξημένες δαπάνες. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα για ένα τομέα που γνωρίζω καλύτερα, αν δει κανεί, ε, για παράδειγμα, σε σχέση με το, ε, την, τη, τις, ε, δοκιμές αντοχής υλικών για τα αυτοκίνητα σε περίπτωση συγκρούσεων για παράδειγμα. Αν δει κανεί το κόστος και επαναλάβει τον υπολογισμό αυτό σε σχέση με το τι κοστίζουν αυτές οι δοκιμές, ενώ θα πρέπει να ε, αναλώνουμε, να δαπανούμε τα κονδύλια που έχουμε για τα ε, καλύτερα αποτελέσματα που μπορούν να επιτευχθούν και όχι απλά για δοκιμές που δεν είναι ιδιαίτερα παραγωγικές. Με ιδιαίτερη χαρά ε, είδα ότι ξαναξεκίνησε το Διατλαντικό Συμβούλιο για τα εμπορικά θέματα και που επικεντρώνονται στις προδιαγραφές της επόμενης γενεάς, νανοτεχνολογία, ηλεκτρική, ηλεκτρονική ε, υγεία, ευφυή, αυτοκίνητα. Αυτά είναι πάρα πολύ λογικά πράγματα ως πρωτοβουλίες. Γιατί δεν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δουλέψουμε ευθύ εξ αρχή με του εταίρου μα, ε, τον είπα, και να καταλήξουμε σε κοινού στόχους Και να καταλήξουμε, για παράδειγμα, και σε σχέση και με την Κίνα και την Ιαπωνία προ την ίδια κατεύθυνση. Ανέφερα αυτά τα θέματα επειδή γνωρίζετε ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή έχει θεσπίσει μια στενή σχέση συνεργασίας και με τη ΣΥΠΑ και σε σχέση και με την αποστολή στην Κίνα εξ ονόματός σας για την, για την υπογραφή μιας πολύ σημαντικής ε, συμφωνίας για τα θέματα αυτά τυποποίησης και προδιαγραφών μεταξύ Κίνας, ΣΥΠΑ, Ευρώπης. Έκανα λόγο για τις ε, υπηρεσίες, γιατί για το ενιαίο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών αυτό είναι σημαντικό για να δούμε πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε την ε, οικοδόμηση του εμπορίου και την δόμηση εμπορικών και υπηρεσιακών σχέσεων. Δεν θα σας εκπλήξει οι δημόσιες ε, ε, αγορές και τα δημόσια συμβόλαια στην περίπτωση προμηθειών. Αυτό και πάλι είναι ένας άλλος τομέας. Συνεργαζόμενοι με τους εταίρους μας θα πρέπει να μπορέσουμε να ανοίξουμε νέες αγορές και ολοκληρώνοντας ε, στην παράγραφό μου συμπερασματικά σε αυτή την έκθεση, όπως είπα και πιο πριν, προσβλέπω στις τροπολογίες που θα καταθέσετε για την καινοτομία για παράδειγμα και τη σημασία που έχει να ανοίξουμε αυτή την αγορά σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες και συγκεκριμένα τώρα για τις νέες τεχνολογίες. Αυτό πάλι διασυνδέεται με την παρατήρησή μου για τις κοινέ προδιαγραφές και όσον αφορά και την τυποποίηση, αλλά και την ενθάρρυνση έρευνας και ανάπτυξης να ανοίξουν ευκαιρίες για μεγαλύτερη συνεργασία με χώρες όσον αφορά αυτή την κονίστρα αυτό το στίβο. Ενδιαφέρομαι να ακούσω τις απόψεις των σκιωδών εισηγητών. Και πάλι είναι απαραίτητε θέλω να πω οι τροπολογίες σας για να εμπλουτιστεί αυτή η γνωμοδότηση, για να μπορέσει να διευρυθεί το ε, φάσμα της και να συμπεριληφθούν οι δικές σας παρατηρήσεις έτσι. Ευχαριστώ. Merci, Malcolm. Ευχαριστώ, Μάλκομ. Θα δώσω το λόγο στους σκιώδες εισηγητές. Η κυρία Λουγκρίπ, πρώτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον πρόεδρε, τον Μάλκολμ Χάρμπορ, για το σχέδιο γνωμοδότησής του. Να τον ευχαριστήσω για τη θέληση που δείχνει από την αρχή να εμπλέξει τους σκιώδεις ε, εισηγητές στην εκπόνηση της ε, γνωμοδότησής του. Ήδη έχει ενσωματώσει κάποιες από τις προτάσεις και τις συστάσεις που εκφράσαμε. Όχι όλες, σίγουρα, αλλά Γι' αυτό ακριβώς κάνουμε και αυτή τη συζήτηση. Η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας απασχολεί τα μάλα, γιατί είναι βασική λόγω της επίπτωσης που μπορεί να έχει, μέσω του προσανατολισμού που της δίνουμε, μέσω των αποφάσεων που παίρνουμε, ε, επηρεάζει άμεσα την ανάπτυξη, την οικονομική μας ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητά μας, την εσωτερική αγορά, την αγορά εργασίας, ε, το σύνολο των προϊόντων που παρουσιάζουμε στους καταναλωτές. Επομένως, επηρεάζει άμεσα και τον τρόπο λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Είναι αυτονόητο και αυτό ακριβώς λέει και η Κομισιόν στην ανακοίνωσή της, ότι η πρώτη προτεραιότητα της Κομισιόν θα πρέπει να είναι να ολοκληρωθεί ο κύκλος της ΔΟΧΑ, αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα η κατάληξη του κύκλου της Ντόχα θα πρέπει να είναι και φιλόδοξη αλλά και ισορροπημένη και παγκόσμια. Για όλα τα μεγάλα, για όλα τα μείζωνα θέματα που είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, φυσικά υπάρχουν και όλες οι συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών που η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να διαπραγματεύεται. Αλλά και εκεί. Αλλά μην ξεχάσουμε σε ποια εποχή και σε ποιο κόσμο ζούμε οι εμπορικοί μας εταίροι είναι και ανταγωνιστές μας παράλληλα. Ακριβώς για αυτό το λόγο και έχοντας συνέστηση αυτής της παγκόσμιας πραγματικότητας, οι συζητήσεις που γίνονται στα πλαίσια του ΠΟΕ και στα πλαίσια των διμερών διαπραγματεύσεων για την ετοιμασία συμφωνιών ελευθέρων ανταλλαγών είναι έμπλες ρεαλισμού. Αλλά στερούνται και στερούνται βεβαίως οποιαδήποτε αφέλεια Θα ήθελα λοιπόν να κάνω κάποιες ε, σκέψεις, τις οποίες θα τις διατυπώσω μέσω τροπολογιών στο σχέδιο του Μάλκολ. Βεβαίως, τα περισσότερα θέματα που είναι αντικείμενο της Επιτροπής μας τα έχει θίξει. Θέλω να επανέλθω απλώς αυτή τη στιγμή σε τρία θέματα. Καταρχάς, η αρχή της αμοιβαιότητας μου φαίνεται σημαντική και της συμμετρίας Νομίζω ότι θα πρέπει να τονίσουμε στη διατύπωση της γνωμοδότησης της Επιτροπής μας αυτές τις δύο αρχές. Αμοιβαιότητα και συμμετρία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το έκτακτο που έγινε το Σεπτέμβριο του 2010, που μίλησε για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους στρατηγικούς της εταίρους, για πρώτη φορά ανέφερε αυτή την έννοια της αμοιβαιότητας και είπε, παραθέτω, ότι η ανεπτυγμένες χώρες και οι αναπτυσσόμενες χώρες, οι εταίροι μας, θα πρέπει να λειτουργούν σε ένα, σε μια, σε ένα πνεύμα αμοιβαιότητας. Υπάρχει αυτό στην ανακοίνωση του φθινοπόρου. Και σε ορισμένε εκθέσεις που ψηφίστηκαν στο τέλος του 2010 αναφέρονται αυτές ε, οι αρχές. Νομίζω ότι και εμείς είναι σημαντικό να ξαναμιλήσουμε για αυτή την αρχή και να την αναπτύξουμε αυτή την ιδέα στο σχέδιο γνωμοδότησή μα. Όλε οι συμφωνίε ελευθέρων συναλλαγών που είναι σε φάση προετοιμασία θα πρέπει να συναυθούν με, με διάφορε απαιτήσει, με φιλοδοξίε και χωρί αφέλεια. Δηλαδή να υπάρχει μια ισορροπία. Να λάβουμε υπόψη τι ιδιαιτερότητε και των δύο μερών, τι οικονομικέ, κοινωνικέ και περιβαλλοντικέ ιδιαιτερότητε και να φτιάξουμε ένα ισορροπημένο όλο. Ιδίω ό,τι αφορά το άνοιγμα των δημοσίων συμβάσεων. Ε, αυτό το είπατε όμως, Πρόεδρε, μάλλον σα το προτείναμε και το έχετε εντάξει στην ε, γνωμοδότησή σας. Επίσης, η επίπτωση που έχουν οι συμφωνίες ελευθερών συναλλαγών σε ορισμένου τομεί της ε, εσωτερικής αγοράς. Γεωργία, αλλά όχι μόνο. μιλάμε για τομεί όπου ε, οι εταίροι μας τους αντιμετωπίζουμε με λιγότερους κανόνες, πολύ λιγότερο δεσμευτικούς κανόνες και αυτό έχει καταστρεπτικές συνέπειες για την ανάπτυξη των δικών μας των μέων που είναι ευαίσθητοι. Στα πλαίσια λοιπόν των διαπραγματεύσεων, πριν από τις, ε, τη σύναψη των συμφωνιών, ε, ελευθέρων συναλλαγών, υπάρχει μια ανάλυση των επιπτώσεων από τη σύναψη αυτών των συμφωνιών στην εσωτερική αγορά. Τελευταίο θέμα. Ένα θέμα που μπήκε επιτάπητος ε, πρόσφατα από τον Επίτροπο Μπάρνιε και τον Επίτροπο Ταγιάννη. Η αξιολόγηση των ε, εξοκοινοτικών επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να υπάρξει ένας προσανατολισμός της ε, στρατηγικής μας της εμπορικής ε, πολιτικής μας στο εξωτερικό που αποφεύγει το σκόπελο της ε, αφέλειας, θα πρέπει οπωσδήποτε να αξιολογήσουμε τις επενδύσεις που κάνουν οι ξένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να δούμε την επίπτωση που έχουν στις επιχειρήσεις μας, στην ε, βιωσιμότητα των πιο οικονομικών μας τομέων. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον αυτό. Συμπερασματικά, ευχαριστώ τον πρόεδρο Χάρμπορ για την δουλειά του για τη δουλειά που έκανε ήδη για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης ε, και εμείς με χαρά θα προσπαθήσουμε να το εμπλουτίσουμε. Ε, λέω αυτά που λέω για να συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτών των ιδεών. Θα δώσω το λόγο στις επόμενες σκιώδους και θα ήθελα να του ζητήσω να είναι λίγο πιο λακωνικοί γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Περνάει ο χρόνος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, λέει η κυρία Στήλερ, ευχαριστώ τον εισηγητή. Θα είμαι σύντομη γιατί πολλά από τα, από τα σας αμεκάλυψαν. Ο εισηγητής μιλάει για τις δημόσιες προμήθειες, για τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα που είναι σημαντικό. Επίσης, ιδέες για τους ηλικιωμένους, και προϊόντα για αυτούς. Η ασφάλεια των προϊόντων για τους καταναλωτές είναι πολύ σημαντικό και χαίρομαι που το έβαλε ο, ο εισηγητής. Στο σημείο 6 μιλάμε για το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή συγκριτικό πλεονέκτημα ε, και τι σημασία έχει στην καινοτομία. Επίσης πρέπει να δούμε τους πόρους και το, δυναμικό ούτως, και να τα κάνουμε αυτά ε, κλειδιά της επιτυχίας ε, της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που υπόθηκε ήδη είναι ε, θέματα, εταιρικής, θέματα εταιρικής ευθύνης. ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον. Όλα αυτά μπορούμε να τα αναπτύξουμε λίγο περισσότερο. Αλλά συνολικά τα στοιχεία που χρειάζονται υπάρχουν. Ε, επίσης, ε, τη δουλειά που έχουμε κάνει ήδη στην Επιτροπή ε, για την τυποποίηση, το αναγνωρίζουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να συγκεράσουμε σε αυτή την έκθεση διάφορες, την εργασία που κάναμε σε διάφορους τομείς πολιτικής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα Ρίτα, για άλλη μία φορά να επιβεβαιώσω ή να ενδυναμώσω στην επιλογή των κυριότερων σημείων τον κύριο για την τυποποίηση και τις προδιαγραφές. Είναι κέριος τομέας αυτός και πολλές φορές πρέπει να τον τονίζουμε και να τον αναφέρουμε για να υπάρχουν αυτές οι προδιαγραφές και να είναι η βάση της εργασίας μας. Θέλω να κρούσω κόδωνα κινδύνου, να μην υπερτιμήσουμε το, τη σημασία του θέματος των δημόσιων προμηθειών. Θέλω να επισημάνω ένα πράγμα, ότι η συζήτηση για το πράσινο βιβλίο και για τις δημόσιες ε, αγορές και προμήθειες θα θέσει το θέμα των συμφωνιών μέσα στο πλαίσιο του ΠΟΕ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και ποιες επιπτώσεις υπάρχουν και στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σε σχέση με την ε, κινητοποίηση που πρέπει να διασφαλιστεί. Θα πρέπει όμως ε, να συντονιστούμε είναι σημαντικό το άνοιγμα των αγορών, αλλά όταν έρχεται αυτό το επιχείρημα ότι βλέπουμε ότι έχουμε δυσκολίες όταν προσπαθούμε με καινοτόμο τρόπο να δραστηριοποιηθούμε, αυτό είναι λιγότερο καλό. Και ένα παράδειγμα είναι ο τομέας του Fairtrade όπου θα έπρεπε να έχουμε τη δυνατότητα οι προμήθειες και οι αγορές ε, να γίνονται σε αυτό το πλαίσιο. Θέλω να χαιρετήσω αυτό που αναφέρε ο προλαλής σας ή προλαλή σας ε, για τις ε, επιπτώσεις. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη μελέτη επιπτώσεων προτού καταλήξουμε σε κάποιες αποφάσεις, ιδιαίτερα για τους ευαίσθητους τομείς. Πρέπει να γνωρίζουμε περισσότερα προτού λαμβάνουμε τέτοιες αποφάσεις. Ευχαριστώ. Monsieur Crossman, Θέλει να, θέλει να μιλήσετε στη θέση της κυρίας Οντήλ Σμιτ. Ο σκιώδης εισηγητής κυρίας Όλε Σμιτ θα ήθελε να ευχαριστήσει τον ε, συντάκτη γνωμοδότησης για τη συνεργασία και τις προτάσεις. Όπως και στη συνάντηση που είχαν προηγούμενα το Μάρτιο, θεωρεί ο κύριος Σμίτ ότι καλύπτονται οι περισσότεροι τομείς. Ωστόσο, θεωρεί ο κύριος Σμίτ ότι η γνωμοδότηση επίσης πρέπει να έχει κάποιες αναφορές για τη σημασία του ελευθέρου εμπορίου όσον αφορά και τα πολιτισμικά θέματα και σε σχέση με την ε, κάλυψη από τον ε, των ε, τιμών. Τα γεωργικά προϊόντα είναι σημαντικό ε, ποσοστό της, ε, των εισαγόμενων και θα πρέπει να μπορούμε να διασφαλίσουμε την καλή λειτουργία της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Σε σχέση με τους συναδέφους ε, ΑΚΕ, ο κύριος Σμιτ μέσα στο πλαίσιο των ΑΚΕ πάντα υπογράμμιζε τη σημασία που έχει η πρόσβαση στην ενιαία εσωτερική αγορά γεωργικών προϊόντων που είναι ένα σημαντικό μέρος ε, του ε, εισοδήματος των αναπτυσσόμενων χωρών ε, τα γεωργικά προϊόντα. Μεγαλύτερο ελεύθερο εμπόριο θα έκανε μεγάλη τεράστια διαφορά για αυτές τις χώρες και για την ενιαία εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εισαγωγή αυτών των προϊόντων, γεωργικών προϊόντων έχει μεγάλη επίπτωση στην ενιαία εσωτερική αγορά και στους καταναλωτές και αυτό θα πρέπει να αναφέρεται σε σχέση με την γνωμοδότηση της ΙΜΚΟ. Ευχαριστώ. Λαπαγόλ Ευχαριστώ. Ο κύριος Τρασκόφσκι και ζητώ συγγνώμη αν διαλύω το όνομά σας. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο για το διατλαντικό οικονομικό Συμβούλιο και σε σχέση με την αντιπροσωπή, σχέση με τις είπα, συμφωνώ για τις σχέσεις, τη σημασία που έχουν αυτές οι σχέσεις και για την αναζωογόνηση του Διατλαντικού ε, Συμβουλίου. Θα πρέπει να το αναφέρουμε αυτό όμως και για το Ευρωκοινοβούλιο, γιατί αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε ε, για τον διάλογο νομοθετών με το Κογκρέσο και για την αλλαγή των προτεραιοτήτων όταν συζητάμε αυτά τα θέματα με τους Αμερικανούς εταίρους. Όχι μόνο να συζητάμε θέματα ε, εξωτερικής πολιτικής αλλά και θέματα ρυθμιστικά όσον αφορά και τις προδιαγραφές και το e-commerce και που θα πρέπει μετά την συνθήκη της Λισαβόνας και κάποιες δυσκολίες που είχαμε να μπορέσουν να ενταχθούν στο σωστό πλαίσιο. Ενδιαφέρον θα ήταν να το αναγνωρίσουμε και αυτό και να το λάβουμε υπόψη σε αυτή τη γνωμοδότηση. Όχι μόνο να κάνουμε λόγο για τα εμπορικά θέματα, αλλά για το τι γίνεται και σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο. Ευχαριστώ. σας ευχαριστώ. Υποστηρίζω απόλυτα την προσέγγιση του Μάκομ διατυπώνοντας σαφώς ότι το ελεύθερο εμπόριο είναι η η πορεία προς το μέλλον και για την ανταγωνιστικότητα και για την ε, ε, ανάπτυξη και για την σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη που δεν μπορούν να, δεν μπορούν να λειτουργήσουν στην παγκόσμια αγορά με τις ίδιες προδιαγραφές όπως άλλες ε, εταιρείες και θα πρέπει να μπορέσουμε να επικεντρωθούμε και στην σύγκληση όσον αφορά και την ασφάλεια των προϊόντων για τους καταναλωτές και το ενδιαφέρον θέμα των, της ασφάλειας των παιχνιδιών. Ενδιαφέρον θέμα με και τα περισσότερα παιχνίδια εισάγονται στην Ευρώπη και πρέπει εδώ να μπορούν να ελέγχονται οι προδιαγραφές, να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και τα παιχνίδια που παράγονται και πολλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια σημαντική παρατήρηση εδώ. Αν θέλουμε να είμαστε συνεκτικοί για τα όσα συμβαίνουν τώρα στην Μεσόγειο και στην όχθη της Βόρειας Αφρικής πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι σε μια, για μια νέα πολιτική εμπορίου για την Ευρώπη να μπορέσουμε να ανοίξουμε αυτή την, αυτές τις πύλες ή αυτές τις χώρες. Δεν μπορούμε μόνο να ζητάμε να προαθεί ο, ε, ο εκδημοκρατισμός αυτών των χωρών και να μένουν τα προϊόντα τους ή να μην είναι ελεύθερα τα προϊόντα τους και οι συναλλαγές. Υπέρ της ειρήνης και της δημοκρατίας πρέπει να γίνει αυτό και θα καταθέσω μια τροπολογία σχετικά με αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν ζητάει κανένα άλλο το λόγο. Τώρα θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Μιγγέλ Σεβάιρος Μπαρόν. Ευχαριστώ για τις συνεισφορές σας ε, σε αυτή την έκθεση. Η ανακοίνωση της Επιτροπής για την ε, ανάπτυξη, το εμπόριο και την ανάπτυξη ε, εντάσσεται στα πλαίσια της ε, ατζέντα για την Ευρώπη 2020. Είναι μια μακρόπνοη στρατηγική. Προσπαθούμε να σπείρουμε τώρα για να ε, κόψουμε τους καρπούς αργότερα. Θέλουμε να εντοπίσουμε τις προτεραιότητες και τους στόχους ε, στην ατζέντα και το εμπόριο και στα πλαίσια του πολυμερούς, των πολυμερών μάλλον διαπραγματεύσεων στα πλαίσια του ΠΟΕ γύρω στις Ντόχα κτλ. Ε, εντοπίζουμε τους στόχους και τις προτεραιότητες που θα πρέπει να διαπραγματευτούμε, αλλά και σε διμερές επίπεδο. Και μόνο μετά το, την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων θα υπάρξει η εφαρμογή. Και μακρο, πιο μακροπρόθεσμα θα υπάρξουν και οικονομικά ωφέλη από όλες αυτές τις πολιτικές. Με μεγάλη χαρά βλέπουμε ότι οι βουλευτές αναφέρθηκαν στους βασικούς στόχους και στις προτεραιότητες αυτής της ανακοίνωσης, κυρίως τη σημασία που δίνει η Κομισιόν να, αντιμετωπιστεί, να αντιμετωπιστούν τα τεχνικά και ρυθμιστικά εμπόδια, όχι μόνο με τους μεγάλους εταίρους όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η νέα ατζέντα με τη ΣΥΠΑ ε, στα πλαίσια του ΤΕΚ έχει δώσει ήδη κάποια αποτελέσματα, αλλά και με άλλους εταίρους. Η Ιαπωνία, Κίνα, με τους οποίους, με τους οποίους έχουμε συνεχή διάλογο. Κάποιες από τις ανησυχίες που αναφέρατε, όπως οι δημόσιες προμήθειες, είναι ψηλά στις προτεραιότητες της Κομισιόν. Επίσης, η αναφορά στις αρχές της συμμετρίας και αμοιβαιότητας, το λαμβάνω υπόψη μου. Στα πλαίσια των δημοσίων προμηθειών θα εφαρμόσουμε αυτές τις αρχές για μεγαλύτερη διαφάνεια και για δυνατότητα ξένων επενδυτών να λάβουν μέρος ε, σε αυτές τις δημόσιες προμήθειες. Ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστώ. Πριν ξαναδώσω το λόγο στο Μάλκομ, θέλω να σε υπενθυμίσω το χρονοδιάγραμμα. Καταθέτουμε τις τροπολογίες μέχρι τις 24 Μαρτίου 12 το μεσημέρι, εξέταση των τροπολογιών στις 12 Απριλίου, ψηφίζουμε στην ΙΜΚΟ στις 13 Απριλίου, ψηφίζουν στην ΙΝΤΑ στις 23 Μαΐου και στην Ολομέλεια τον Ιούνιο. Δίνω το λόγο τώρα στο Μάλκον για να μας πει τα τελικά του σχόλια. Και οι δύο εκθέσεις ε, ήταν πάρα πολύ σημαντικές και τον ευχαριστώ εκ των προτέρων. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε ως εισηγητής ε, να ε, αναφέρομαι στην Επιτροπή και υπό την Προεδρία σας. Δεν έχω να προσθέσω πολλά. Όλα αυτά έχουν πάρα πολύ ε, σημαντική πρόσθετη αξία. Προσβλέπω στις τροπολογίες σας ένα πράγμα που θα ήθελα να δώσω συνέχεια σε σχέση με τον κύριο Τρασκόφσκι. Ένα σημαντικό σημείο. Έχει δίκιο φυσικά ότι θα έπρεπε να το αναφέρουμε αυτό σε σχέση με τον νομοθετικό διάλογο διατλαντικά. Θα ήθελα να προσθέσουμε όμως κάτι εδώ σε αυτό ότι και άλλες κοινοβουλευτικές ε, επιτροπές πρέπει να εμπλέκονται πολύ περισσότερο σε αυτό το πλαίσιο από ότι μέχρι σήμερα έχει δίκιο που λέει ότι προχωρεί η νομοθεσία διατλαντικά και σε σχέση με τον διάλογο πρέπει να προαχθεί ακόμα πιο πολύ. Αλλά χρειάζεται και πραγματογνωμοσύνη ε, πραγματογνωμόνων όπως ε, της δικής μας ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και πρέπει να υπάρχει εμπλοκή σε αυτό το διάλογο σε σχέση με την αντιπροσωπεία για τη ΣΥΠΑ και για το Κογκρέσο μέσα στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου. Δεν γίνεται αυτό και δεν γίνεται συχνά. Πρέπει να γίνεται όμως. Λοιπόν, μια ευκαιρία είναι αυτό που υπάρχει να προσθέσουμε αυτό το σημείο με την υποστήριξή σας θα το συζητήσω να δούμε πώς θα υπάρξει μια τακτική μορφή τροπολογία που θα μπορέσει να κατατεθεί και να υποστηριχθεί ώστε και από πλευρά του κυρίου Μπρόκ να διασφαλιστεί ως πρόεδρος που είναι αυτής της Επιτροπής ε, να εμπλέκονται περισσότερο οι ενδιαφερόμενοι. Ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο η πρόεδρος. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να εργαστώ ε, από αυτών των δύο θεμάτων που μου κινούν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον. Και τώρα έχουμε έκθεση του κύριου Ρέπο επί της τροποποίησεως του κανονισμού για τη συνεργασία μεταξύ εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνε για την επιβολή των, ε, του δικαίου προστασίας των καταναλωτών. Αρχικά, η αρχική νομοθεσία είχε, την είχε επεξεργαστεί η κυρία Γκέπχαρτ στην πρώτη φάση της ζωής της Επιτροπής ΙΜΚΟ το Έξι και τέσσερα μάλλον. Θα δώσω το λόγο λοιπόν τον, στον κύριο Ρέπο για να αναπτύξει την, ε, αναθεωρημένη, τον αναθεωρημένο αυτόν κανονισμό. Μετά ο σκιώδης ηγητής είναι παρόν ο Σάιμον Μπούσουτιλ, τον οποίο καλωσορίζω και άλλα πρόσωπα. Και θα ήθελα να λάβω και εγώ το λόγο εξ ονόματος της δικής μου πολιτικής ομάδας και έχουμε και τον κύριο Μόλνερ που τον γνωρίζει καλά η Επιτροπή Ενίας Αγοράς και έχουμε και εκπρόσωπο της Ουγγρικής Προεδρίας που επίσης θα κληθεί να λάβει το λόγο εφόσον το επιθυμεί. Ρέπο λοιπόν πρώτος λαμβάνει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ για πρώτη φορά συζητάμε μια πρόταση για κανονισμό όσον αφορά την συνεργασία για την προστασία καταναλωτών και συναφή θέματα και πώς θα πρέπει να διαμορφωθούν αυτά. Σε αυτή τη φάση ενδιαφέρομαι περισσότερο να ακούσω τις απόψεις των άλλων σκιωδών εισηγητών και άλλων συναδέλφων και σε σχέση και με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που συναντήσαμε και εκπροσώπους της Ουγγαρίας και που συζητήσαμε με αυτούς ε, τα θέματα, θα συναντηθούμε και με άλλους ε, αυτή την εβδομάδα. Από το 2004 έχουμε έναν κανονισμό πλέον που καλύπτει την ευρωπαϊκή, πανευρωπαϊκή επιβολή των προδιαγραφών προστασίας καταναλωτών και θεμάτων συνεργασίας μεταξύ εθνικών αρχών και για το πώς θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα δίκτυο επικοινωνίας. Θέλουμε επίσης να εναρμονιστούν τα ε, δικαιώματα και τα θέματα εφαρμογής ε, και μέσω μηχανισμών ε, ανταλλαγής πληροφοριών και όταν λαμβάνονται αποφάσεις και μέτρα για την κύρωση παραβάσεων όταν συμβαίνουν αυτές οι παραβάσεις ε, διασυνοριακά. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ένα υψηλότατο επίπεδο πανευρωπαϊκά και να βελτιωθεί και να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Έχει υποβληθεί μια τροπολογία σε, αυτόν τον, σε αυτήν την πρόταση κανονισμού. Αφορά όμως ε, μόνο τις νομοθετικές πτυχές ε, και τις τεχνικές πτυχές χωρίς να επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής. Πράγμα το οποίο θα σημαίνει ότι θα σημαίνει ότι θα επικαιροποιηθεί το παράρτημα. συζήτησα τα θέματα με του εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατέστησα σαφέ ότι ο πιο σημαντικό ρόλο, λόγο για την αναθεώρηση του κειμένου είναι το θέμα τη ε, ε, εμπιστοσύνη των καταναλωτών, οδηγία ε, για την αύξηση αυτής της εμπιστοσύνης. Εκεί το θέμα της νομικής βεβαιότητας και ασφάλειας θέτει ένα θέμα ιδιαίτερα όταν αφορά αυτό την προστασία των καταναλωτών, αλλά και όταν το βλέπουμε και υπό το πρίσμα των κρατών μελών. Είναι ε, ε, ένα θέμα το οποίο δημιουργεί κάποια προβλήματα. Δεν αμφιβάλλουμε για τις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ταυτόχρονα υπευλήθηκε η πρόταση των παρατημάτων που θα επικαιροποιηθούν και θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε σχέση με τις ε, ε, παρεμβάσεις που γίνονται σε αυτό το πλαίσιο και που θα πρέπει να αντικατασταθούν από το κείμενο της νέας οδηγίας. Ε, επίσης σε σχέση και με το παράρτημα τα δικαιώματα των ε, επιβατών για παράδειγμα σε σχέση με τις μεταφορές από το 2004 αυτά όλα έχουν ενταχθεί σε διαφορετικές διατάξεις αυτού του κανονισμού. Άλλες αλλαγές από την άλλη πλευρά αφορούν την διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής ε, και σε σχέση με το παράδειγμα. Αυτό όμως δεν ανήκει σε αυτό το, στο πλαίσιο αυτής της πρότασης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι για πολύ μικρό διάστημα υπάρχει αυτό το πλαίσιο και δεν έχουμε αρκετές, ε, αρκετή ε, πείρα για το τι μπορεί να γίνει. Ούτε έχουμε από την άλλη πλευρά επαρκή στοιχεία και σε σχέση με την, τις επαφές μου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δίκτυο CPC και η αξιολόγηση που βρίσκεται καθοδόν υπό εκπώνηση κατά το δεύτερο τμήμα του, το τελευταίο τμήμα του 2011 θα αρχίσει ε, αξιολόγηση σε σχέση με τα αποτελέσματα και θα δημοσιευθούν τα αποτελέσματα του χρόνου το 2012. Στη συνέχεια θα υπάρξει δημόσια διαβούλευση και μόνο όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η διαβούλευση δηλαδή κάπου το 2014, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι έτοιμη να εξετάσει την ε, μεταρρύθμιση, την αναθεώρηση του συστήματος. Κατά τη διάρκεια της Βελγικής Προεδρίας συζητήθηκε το θέμα, πρότεινε το Βέλγιο να υπάρξει μια τροποποίηση του κειμένου, ώστε να υπάρχει υποχρέωση πλέον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάζει την διεύρυνση του, φάσμα, του πεδίου εφαρμογής και σε άλλες οδηγίες για την προστασία των καταναλωτών και ταυτόχρονα να εξετάζεται πώς θα μπορέσει να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του δικτύου CPC και να υποβάλει σχετική πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποφασίστηκε όμως σε σχέση με την ομάδα εργασίας να υιοθετηθεί μόνο η τεχνική μορφή τροποποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μην υπάρξουν άλλες αλλαγές σε σχέση με το κείμενο για τον κανονισμό. Τι θα έπρεπε στη συνέχεια τώρα να κάνει το Ευρωκοινοβούλιο. Όπως προανέφερα, σε αυτή τη φάση θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ να ακούσω τις δικές σας, τις ίδιες τις δικές σας απόψεις επί του θέματος. Προσωπικά βλέπω τρεις εναλλακτικέ λύσεις εδώ. Η πρώτη θα ήταν μια μινιμαλιστική λύση. Να δεχθούμε δηλαδή με άλλα λόγια την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια τεχνική τροποποίηση δεν θα άλλαζε ο κανονισμός, η άλλη όμως εναλλακτική λύση είναι μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα θα προσθέταμε την πρόταση της Βελγικής Προεδρίας την Βελγική πρόταση για μια αναθεώρηση του κειμένου λαμβάνοντας υπόψη και τις ε, προθεσμίες όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι έχει ήδη ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μέτρα για την αξιολόγηση του συστήματος και τρίτη εναλλακτική λύση μαξιμαλιστικής προσέγγισης αλλαγές στο κείμενο για να διευρυνθεί το φάσμα του κανονισμού. Υπό το φως των, ε, της πείρας μας ε, θα ήθελα να κάνουμε μόνο πολύ μικρές αλλαγές γιατί δεν έχουμε αρκετά στοιχεία ή τεκμήρια με βάση τα οποία θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στην υιοθέτηση ευρύτερων αλλαγών σε αυτή τη φάση. Αλλά επίσης ε, και η μεσοπρόθεσμη λύση θα ήταν εφικτή. Μια και όμως ξεκινάμε διαπραγματεύσεις και συζητήσεις σε αυτή τη φάση δεν θα ήθελα να προδικάσουμε την έκβαση αυτών των συζητήσεων με οδήποτε τρόπο. Όμως πιστεύω ότι η προστασία των καταναλωτών και η νομοθεσία σχετικά με την προστασία των καταναλωτών θα πρέπει να, να γίνεται σε ένα, ολοκληρωμένο θα έλεγα ε, βάθρο για να μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί και για προτάσεις που θα διασφαλίζουν την θέση των, των, τα δικαιώματα των καταναλωτών και στο μέλλον και αυτό θα μπορούσε να συγκριθεί με τις, ε, την προσέγγιση συλλογικής δράσης ε, που θα μπορούσε να αναλυθεί. Και η συνεργασία μεταξύ των ε, αρχών έχει και η συνεργασία αυτή έχει και τη σημασία της για μια πρόταση σχετικά που θα έπρεπε να οδηγήσει σε μια ε, εκκίνηση των συζητήσεων σχετικά σύντομα ώστε να έχουμε το επόμενο φθινόπωρο κάποιες προτάσεις ε, προς λήψη απόφαση. Ανάλογα με το ποια προσέγγιση θα υιοθετηθεί, ποια εναλλακτική λύση θα υιοθετηθεί, θα εξαρτηθεί η ταχύτητα με την οποία θα προοδεύσει αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τα στοιχεία που βάζετε στην, πρόταση, σας. Συμφωνώ ότι πρέπει να δουλέψουμε πολύ γρήγορα. Οι βασικές αρχές του κανονισμού, όπως βλέπω και από την έκθεσή σας και τις εξηγήσεις σας, ε, δεν τίθεται να αμφιβόλω, είναι απλώς ε, θέμα αναθεώρησης του. Ε, επίσης, το θέμα της κανονικής πίστης, ε, η σχετική πράξη δηλαδή, πρέπει να συμπεριληφθεί. Ε, μας έχει απασχολήσει και μας αυτήν την Επιτροπή αυτό το κείμενο για την κανονική πίστη. Τώρα ας ακούσουμε τους σκιώδεις εισηγητές, ο κύριος Πουσουτήλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή για τη σαφή παρουσίασή του. Αν κατάλαβα καλά, προτείνει μία από τις τρεις επιλογές. Η πρώτη είναι απλώς να επικυρώσουμε την πρόταση, μια και είναι ουσιαστικά τεχνική πρόταση. Δεύτερον, ε, να βάλουμε μια ρήτρα αναθεώρησης είναι μια ενδιάμεση λύση και η τρίτη λύση είναι να μπούμε σε βαθιές αλλαγές. Εγώ συμφωνώ μαζί του ότι θα πρέπει να επιλέξουμε τη δεύτερη επιλογή, δηλαδή να βάλουμε μια ρήτρα αναθεώρησης. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει αυτή την τεχνική πρόταση να τη χρησιμοποιήσουμε για να επιφέρουμε ουσιαστικέ αλλαγέ στον κανονισμό, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Συμφωνώ όμω ότι χρειάζεται μια αναθεώρηση για γιατί αυτό το κείμενο δεν μας έδωσε ούτε σε εμά ούτε στους καταναλωτές αυτό που θέλαμε. Υπάρχουν όλο και περισσότερες περιπτώσεις στην καθημερινή μας ζωή, στην καθημερινή ζωή των καταναλωτών, ε, διασυνοριακών αγορών, και η προστασία των καταναλωτών και οι σχετικές αρχές που προστατεύουν τους καταναλωτές δεν συνεργάζονται μεταξύ τους επαρκώς για να εξασφαλίσουν αυτή την προστασία των καταναλωτών όταν αγοράζουν σε μια άλλη χώρα, διασυνοριακά λοιπόν. Επομένως χρειάζεται μια αναθεώρηση. Ε, είναι σαφές ότι οι υπηρεσίες ε, προστασίας των καταναλωτών πρέπει να συνεργάζονται καλύτερα και να επανορθώνουν ε, τι ζημίε που υφίστανται οι καταναλωτέ όταν αγοράζουν σε άλλη χώρα. Ναι, χρειάζεται βελτίωση, αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει ε, να αναθεωρήσουμε ε, άρδιν μέσω μιας τεχνικής πρότασης. Έτσι λοιπόν ε, θερμό, θέλω να υποστηρίξω τη δεύτερη εναλλακτική του λύση. <coughs> Ευχαριστώ κύριε Μπουσουτήλ. Για το θέμα της εφαρμογής ε, είναι ένα θέμα χωριστό που το συζητήσαμε με την Επιτροπή. Υπήρχε και μια προφορική ερώτηση για την αποτελεσματικότητα του κειμένου. Ε, έχουν γίνει διάφορες αλλαγές. Έχουμε τώρα κάποια στοιχεία συγκριτικά. Καλό είναι να έχουμε το νομικό πλαίσιο, αλλά πρέπει να εφαρμόζεται κιόλας καλό θα ήταν και τα κράτη-μέλη να αφιερώνουν τους απαραίτητους πόρους για την εφαρμογή αυτού του κειμένου. Κύριο Στροσφόρ, ευχαριστώ τον κύριο Ρέπο για την ε, παρουσίασή του που ήταν πολύ σαφής. Θέλω να πω σε όλους τους συναδέλφους ότι παρότι αυτό το κείμενο είναι πολύ τεχνικό, έρχεται την κατάλληλη χρονική στιγμή. Μόλις τελειώσαμε στην Επιτροπή την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Αυτά τα πράγματα είναι συμπληρωματικά μεταξύ του. Υπάρχει το πλαίσιο τη οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Προστίθεται ο κατάλογο των οδηγιών που αφορούν του καταναλωτέ και από την άλλη υπάρχει το δυναμικό πραγματική εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη αυτού του μηχανισμού. Νομίζω ότι για όλους, αλλά και για την ομάδα μας κυρίως, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια αποτελεσματική εφαρμογή αυτών που ψηφίζουμε, ούτως ώστε να εξυπηρετήσουμε όχι μόνο τον καταναλωτή, αλλά και τις επιχειρήσεις και τις μικρές επιχειρήσεις που εξυπηρετούν τους ε, πολίτες σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα είναι πολύ ε, συγκεκριμένο. Κυρίως να δούμε ποιες είναι οι παράνομες και αθέμητες πρακτικές. Θα πρέπει δηλαδή αυτοί που δεν είναι ε, τίμοι έμποροι να εντοπίζονται, να στυλιτεύονται, ειδικά όταν δρουν διασυνοριακά. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι στον κανονισμό του 2004 αναφέρεται ότι η Κομισιόν κάθε δύο χρόνια θα πρέπει να εκπονεί μια έκθεση που να κάνει έναν απολογισμό για την εφαρμογή αυτού του κανονισμού. Το κάνει. Αν κοιτάξουμε το, την τελευταία αυτή έκθεση της Κομισιόν για την εφαρμογή του κανονισμού, ε, είναι πολύ διαφωτιστική. Αποδεικνύεται ότι είναι πολύ χρήσιμο αν δούμε ότι, ας πούμε, 87 άτομα ε, συνελήφθησαν τον Απρίλιο του 2008 γιατί ε, είχαν μπλεχτεί εκεί σε μία απάτη. Αυτό αποδεικνύει ότι λειτουργεί το πλαίσιο. Ε, ζητάμε περίπου, τα κράτη μάλλον, υποβάλλουν περίπου 100 αιτήσει αμοιβαίας συνδρομή για να εντοπίσουν έτσι, προβληματικές και ύποπτες καταστάσεις. Όταν κοιτάξουμε πιο προσεκτικά, βλέπουμε ότι τα αιτήματα που λαμβάνονται κατανέμονται δίκαια, ας πούμε, ισορροπημένα στα κράτη-μέλη. Δηλαδή καλύπτουμε όλη την επικράτεια, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα τα κράτη-μέλη. Αλλά για τα αιτήματα τα οποία φεύγουν από ένα κρατός μέλος, εκεί έχουμε διαφορές. Δηλαδή, σε ορισμένα κράτη-μέλη ζητούμε πολλές πληροφορίες ή ζητάμε πολλά αιτήματα συνδρομής χάρη στο δικτυο εδω ενώ υπάρχουν άλλα κράτη-μέλη τα οποία δεν ζητάνε τίποτα. Δεν ε, υποβάλλουν καμία αίτηση. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτά τα κράτη-μέλη είναι απόλυτα θωρακισμένα οποιαδήποτε αθέμητη πρακτική. Απλώς δεν υπάρχουν τα μέσα, δεν κινητοποιούνται τα κράτη-μέλη ούτως ώστε να γίνονται όλα όσα προβλέπει ο, όλα προβλέπει ο κανονισμός. Από όλα αυτά λοιπόν τι συνάγω. Ότι αν πρέπει να γίνει κάπου μια προσπάθεια, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν με την ίδια αποτελεσματικότητα αυτόν τον κανονισμό, ούτω ώστε να έχει νόημα αυτή η ιστορία. Να μην υπάρχουν δηλαδή κράτη κράτη-καταφύγια, αν θέλετε, για ορισμένους ε, εμπόρους οι οποίοι είναι παράνομοι, παρά, παράτυποι και που δεν εκτίθενται και που δεν τους ζητάμε να λογοδοτήσουν σε αυτά τα κράτη-μέλη, καταφύγια. Είναι η μοναδική ε, απέτηση που διατυπώνω. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε τον κύριο Ρέπο. Θα συζητήσουμε τις τρεις εναλλακτικέ λύσεις που μας προτείνει. Όπως και αυτός και όπως ο εισηγητής του ΕΛΚ ε, θεωρώ ότι πρέπει να δείξουμε ρεαλισμό. Δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να προσαρμόσουμε να προσαρμοστούμε, να υπάρχει αποτελεσματικότητα, ταχύτητα, αλλά μην κάνουμε υπερβολικές προσπάθειες προσαρμογής, όσο χρειάζεται. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογής. Θέλω λοιπόν να εφαρμοστεί απλώς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το κείμενο όσο έχει σήμερα. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν επίσης τις ε, ευθύνες της Κομισιόν ε, και να την υποστηρίξουμε απέναντι στις ε, προσπάθειες που κάνει σε σχέση με τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Και εγώ επιθυμώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή, ο οποίος έκανε μια θαυμάσια εισαγωγή στο θέμα. Υποστηρίζω την πρότασή του. Ας μην το εξής. Έχουμε την έκθεση Charles για την οδηγία GBST για θέματα εποπτείας των αγορών και για μια ευρωπαϊκή τυποποίηση στο θέμα αυτό. Εάν επανέλθει πρέπει να ξανασυζητηθεί. Γι' αυτό και δεν έχει νόημα εδώ να, κάνουμε, να επιφέρουμε μεγάλες διαφορές, μεγάλες αλλαγές. Μόνο εφόσον επανεξεταστεί η οδηγία για την ασφάλεια των τροφίμων, τότε θα πρέπει να επανεξεταστεί. καθώς επίσης και για την καταναλωτική πίστη. Εφόσον επανέλθουν αυτά, ούτως ή άλλως νομίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει σχέδιο αναθεώρησης. Καθώς επίσης εδώ εντάσσεται και η έκθεση του κ. Σβάμπ για τα, δικαιώματα των καταναλωτών. Αυτά θα έρθουν και τότε δεν χρειάζεται να τα ζητήσουμε. Εγώ προτιμώ λοιπόν αυτές τις αλλαγές με μικρά βήματα που προτείνει ο κύριος Ρέπο. Σας ευχαριστώ. Εδώ ολοκλήρωσα τον κατάλογο των εγγεγραμμένων. Τώρα θα απολαύσετε τα δικά μου σχόλια. Αλλά ήδη το απολαύσατε. Θα δοσοσυγήσω ζητήσω από τον κύριο Μολιέ τώρα να απαντήσει σε ενδεχόμενα ερωτήματα που τέθηκαν. Μετά θα επιστρέψω τον λόγο στον κύριο Ρέπο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε για συζήτηση αυτή τη πρόταση τόσο γοργά. Το εκτιμούμε ιδιαίτερα αυτό και τονίζει πραγματικά τις ανησυχίες, τα μελήματα των σκιωδών εισηγητών που πρέπει το δυνατόν ευρύτερα να ληφθούν υπόψη και να δράσουμε όσο γίνεται ταχύτερα. Όπως επεσήμανε ο κύριος Ρέπος στην εξαιρετική του παρουσίαση, είναι καθαρά τεχνικού χαρακτήρα πρόταση αυτή. Είναι τεχνικού χαρακτήρα επειδή όλες αυτές οι αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί από το Συμβούλιο, από το Ευρωκοινοβούλιο και έχουν ήδη νομοθετηθεί αυτές οι προσεγγίσεις. Θέλουμε να αποφύγουμε τη νομική αβεβαιότητα. Θέλουμε να υπάρξει μια, ένα σαφές πλαίσιο και σε αυτή τη φάση δεν στοχεύουμε στο να αλλάξει το φάσμα το εύρος ή να αλλάξουν οποιαδήποτε άρθρα νομοθετικά άρθρα. Τα επιχειρήματα έχουν ήδη αναφερθεί. Θα ήθελα απλά να επαναλάβω κάποια πράγματα. Έχει λειτουργήσει επί τέσσερα χρόνια αυτός ο κανονισμός μόνο και όπως ε, επισημάθηκε τα πρώτα δύο χρόνια επικεντρώθηκαν σε τεχνικού χαρακτήρα θέματα. Αυτή είναι τώρα η τεχνική η ε, συγκυρία για την ε, σύνταξη της αξιολόγησης σε σχέση με τις προτάσεις που θα υποβληθούν στο Κοινοβουλίο που θα κάνουμε και λόγο για την εφαρμογή. Αλλά σε σχέση με τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής. Πρέπει να κατανοήσουμε λοιπόν την αναγκαιότητα των αλλαγών, αλλά νομοθετικού χαρακτήρα χωρίς να πειράξουμε τον κανονισμό ή μήπω θα πρέπει σε σχέση με την εφαρμογή να προχωρήσουμε με την κοινή προσέγγιση για τις πρακτικές και προτεραιότητες για να κατανοήσουμε αυτά τα πράγματα κατά τη διάρκεια αυτού του έτους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διοργανώσει ημερίδες και ε, σεμινάρια μελετών. Σήμερα ήμουν επικεφαλής ε, ενός ε, σεμιναρίου για την προστασία προσωπικών δεδομένων και θα δούμε και άλλα θέματα τα οποία προήχθησαν από την Βελγική Προεδρία πέρσι. Όπως προαναφέρθηκε θα κάνουμε μια εξωτερική αξιολόγηση για την εφαρμογή του κανονισμού και θα είναι τότε η χρονική στιγμή κατά την οποία θα έχουμε την τρίτη διετή έκθεση που θα παρουσιαστεί για την επόμενη περίοδο και αυτό συμπίπτει ιδιαίτερα με τον χρονορίζοντα όπως είχε αρχικά υπό την Βελγική Προεδρία στις συναντήσεις ε, της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου. Η τρίτη λοιπόν φορά, για τρίτη φορά θα συνέρθουμε και θα προσέλθουμε στο Ευρωκοινοβούλιο και τότε θα είναι η χρονική στιγμή όπου θα μπορέσουμε να σας εκθέσουμε το τι τεκταίνεται, ποια θα πρέπει να αλλάξουν και πού πιστεύουμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Και πάλι σε σχέση με ένα πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης που πρέπει να γίνει, θα πρέπει οι 300 τόσες ε, ε, αρχές που συνεργάζονται μαζί μας ε, να μπορέσουν ε, να εμπλακούν. Εκείνες γνωρίζουν καλύτερα τι πρέπει να αλλάξει. Σήμερα δεν έχει κανένας άλλος αυτές τις γνώσεις. Και για να καταφέρουμε να έχουμε αξιόπιστες ισχυρές προτάσεις θα πρέπει να τις αναλύσουμε και θα πρέπει να υπάρχει και γνώση όσον αφορά τις αρμοδιότητες των αρχών αυτών. Θα γίνει λοιπόν μια σε βάθος αξιολόγηση για να δούμε τι θα πρέπει να γίνει με αυτόν τον κανονισμό. Για όλους αυτούς τους λόγους πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να περιοριστούν οι φιλοδοξίες σε αυτή τη φάση και να αναφέρονται μόνο στις, ε, στο ελάχιστο αναγκαίο, στο ελάχιστο ε, αναγκαίο ως πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη οποιασδήποτε καλές ε, προτάσεις ε, που μπορούν να διατυπωθούν και θα εξεταστούν αργότερα και έτσι μέχρι το 2014 θα είμαστε σε θέση με αυτή τη διαδικασία να υιοθετήσουμε μια αναθεωρημένη διατύπωση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν χρειαστεί αυτό, ακόμα δεν ξέρουμε αν θα είναι αναγκαίο και αν θα χρειαστεί ή όχι. Η διαδικασία προβλέπει όμω ε, και την δυνατότητα αυτή. Θέλω και πάλι να ευχαριστήσω όλου όσου παρενέβησαν διότι πραγματικά αυτό δίνει τη δυνατότητα να προβληματιστούμε σοβαρά για τα θέματα προστασίας ε, των καταναλωτών. Θα πρέπει να ενδυναμωθεί αυτή η συνιστόσα για την ενιαία εσωτερική αγορά και να αποβεί προς όφελος των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Ευχαριστώ για την υποστήριξη όλων εκείνων που εξέφρασαν τις απόψεις τους. Ευχαριστώ όλους εκείνους ε, και τον Πρόεδρο φυσικά. Ευχαριστώ. Uh, Σας ευχαριστώ. Έχουν γίνει συζητήσεις μεταξύ των αρχών επιβολής και είναι αποφασισμένες να επιτρέψουν στα συστήματα να λειτουργήσουν καλύτερα. Από, την, από το Συμβούλιο τώρα, η εκπρόσωπος του Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εξ ονόματος της Ουγγλικής Προεδρίας θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω και χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι ανάμεσά σας και πάλι στη δική σας Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Η Ουγγρική Προεδρία θα προσπαθήσει να συνεργαστεί με τον καλύτερο τρόπο μαζί σας, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ευρύτερα. Είναι μια προτεραιότητα αυτή για μας κατά τη διάρκεια των έξι αυτών μηνών της Προεδρίας μας. Με βάση τα όσα άκουσα είναι σαφές πλέον για μένα ότι αυτό το χαρτοφυλάκιο είναι ένα υπόδειγμα αυτής της στενής συνεργασίας. Η, τα σημεία αφετηρίας βρίσκονται πολύ κοντά το ένα στο άλλο από πλευρά Προεδρία και Ευρωκοινοβουλίου. Τρεις παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω, τρία σχόλια. Αυτό το σχέδιο αφορά την αναβάθμιση ενός νομοθετικού πλαισίου, ε, ενός νομοθετικού ε, έργου. Πρόκειται εδώ για την ακριβώς την προσπάθεια και συμφωνώ ότι μια μινιμαλιστική προσέγγιση είναι ευκταία. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ από την άλλη πλευρά ότι αυτό, αυτή η προσέγγιση δεν αποκλείει από την άλλη πλευρά την αναγκαιότητα, την ανάγκη μιας ευρύτερης αναθεώρησης ύστερότερα, μιας πιο εξειδικευμένης αναθεώρησης σε υστερότερη φάση αν αυτό καταστεί αναγκαίο. Έχει επιτευχθεί συμφωνία σε σχέση με το Συμβούλιο σε επίπεδο ομάδας εργασίας ε, που ευθυγραμμίζεται με αυτά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προανέφερε και εξέθεσε. Δηλαδή η ομάδα εργασίας συμφώνησε με άλλα λόγια ότι θα ακολουθηθεί μια μινιμαλιστική προσέγγιση και θα προσαρμοστεί η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεχόμαστε ότι θα περιοριστούμε έτσι στην επικαιροποίηση μόνο και ενημέρωση αυτών των ε, εδαφείων Προσβλέπουμε στις προτάσεις ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις τροπολογίες ε, των Ευρωβουλευτών και με ιδιαίτερη ικανοποίηση θα συνεργαστούμε στενά μαζί σας. Ε, είμαστε μια φιλική προς το Ευρωκοινοβούλιο Προεδρία και έτσι θέλουμε να εξελιχθούν τα πράγματα και να συνεχίσουν να εξελίσσονται. Θα καταβάλουμε, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Έχουμε ήδη έρθει σε επαφή με τον εισηγητή και δεν υπάρχουν διαφωνίες μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ και εσάς και τους συναδέλφους σας για την στενή συνεργασία σε θέματα προστασίας καταναλωτών. Κύριε Ρέπο, επιθυμείτε να ολοκληρώσετε και να μας προτείνετε και χρονοδιάγραμμα. διάγραμμα. ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Μάκομ Χάμπορ, τον πρόεδρο, του συναδέλφους, τους κοιότητες συζητητές, τους εκπροσώπους της Προεδρίας. Σας ευχαριστώ όλους σας. Και εγώ ως Φινλανδός πρέπει να πω ευχαριστώ για όλες τις προτάσεις και ιδέες. Θα συνεχίσω τη δουλειά αυτή με την ομάδα μου και όσους συνεργάζονται, μαζί μας. Η ιδέα είναι να διατηρηθεί η όθηση αυτή και με ταχύς ρυθμούς να προχωρήσουμε. Θα έχουμε σύντομα το σχέδιο του κειμένου και θα ε, μεταφραστεί και κατά τα μέσα Απριλίου θα είναι ελπίζουμε στα χέρια μας και θα μπορέσουμε έτσι να συζητήσουμε πιο εξειδικευμένα αυτά τα θέματα στην επόμενη συνάντησή μας. Η ψήφιση θα πρέπει να προβλέπεται ήδη κατά τα τέλη Μαΐου στην Επιτροπή ΙΝΚΟ αν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο αυτό. Ευχαριστώ. Yes, I think that's... Ναι, νομίζω ότι είναι εύλογο το χρονοδιάγραμμα. Είναι προφανές άλλωστε ότι η Επιτροπή ΙΜΚΟ το υποστηρίζει. «28 Μαρτίου θα σταλεί η έκθεση στην μετάφραση 12-13 Απριλίου θα την συζητήσουμε και 20 Απριλίου οι ε, τροπολογίες για να ψηφιστεί στην, ε, πριν τα τέλη Μαΐου και στην Ολομέλεια τον Ιούνιο. Υπό την δική σας Ουγγρική Προεδρία πάντως, κυρία Κέρτες. Ευχαριστώ λοιπόν. Θα προχωρήσουμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έκθεση Myers, έκθεση Mayer μάλλον, επιλογές πολιτικής. Από ό,τι έμαθα όμως ο κύριος Μάιερ δεν ε, είναι σε καλή υγεία σήμερα. Θα λάβει το λόγο ο κύριος Σβάπ λοιπόν εις αντικατάστασή του και είναι και παρούσες οι παρόντες οι σκιώδεις Σφάμπ και μετά οι υπόλοιποι ισχυώδεις ηγητές, μάλλον οι οποίοι είναι όλοι μαζί μια ισχυρή ομάδα. Για την έκθεση λοιπόν του κ. Hans Πέτερ Μάιερ, ο κ. Σφάμπ, ευχαριστώ. Ο κ. Μάιερ δυστυχώς ασθενεί σήμερα και μου παρακάλεσε να τον αντικαταστήσω. Το θέμα του σχετίζεται και με το θέμα που προωθώ εγώ, που ε, συντάσσω δηλαδή έκθεση από αυτού, πράσινη βίβλος για Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων και για τις 89 κατατεθήσεις τροπολογίες, τις οποίες έχει συζητήσει με τους σκιώδεις συζητητές. Νομίζω πρώτα συμφωνούμε όλοι ότι οφείλουμε να προστατεύσουμε και να διατηρήσουμε το υψηλό επίπεδο προστασίας των Ευρωπαίων καταναλωτών. Αυτό ήδη αποτελεί αντικείμενο της εκθέσεως, αλλά και αντικείμενο των τροπολογιών. Συμφωνούν επίσης όλοι για την μελέτη επιπτώσεων. Το ερώτημα που τίθεται είναι με ποια μορφή και ποιες θα είναι λεπτομέρειες θα δοθούν. Εδώ υπάρχουν πολλές και διάφορες τροπολογίες από ολόκληρο αριθμό συναδέλφων, αμφωτέρων των φίλων. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα προτιμά τις τροπολογίες 24, 27 και 56 που ζητούν σε βάθος εξέταση. Εγώ θα παρακαλέσω τον εισηγητή να υποστηρίξει τις τροπολογίες αυτές, ώστε να διασφαλιστεί στην τελική ψηφοφορία επαρκής πλειοψηφία για την μελέτη των επιπτώσεων. Πέραν αυτών, συμφωνούμε επίσης ότι είναι σημαντικό να αναμένουμε τα αποτελέσματα που θα δώσει η Οδηγία Προστασίας Δικαιωμάτων Καταναλωτών και μετά να συνδυάσουμε τα δύο κείμενα. Τέλος, πρέπει να έχουμε την δυνατότητα ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσουμε να εξετάσουμε τα πορίσματα της ομάδας εμπειρογνωμόνων πριν να προχωρήσουμε σε υιοθέτηση κάποιου μηχανισμού εναλλακτικού για το ε, δίκαιο συμβάσεων. Είμαι βέβαιος ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τα λάβει αυτά υπόψη και ως αποτέλεσμα της διαδικασίας διαβουλεύσεων. Τώρα, ως Επιτροπή αγοράς και προστασίας καταναλωτών με αποκλειστική αρμοδιότητα για το θέμα αυτό, οφείλουμε να πούμε τη γνώμη μας για τις διάφορες επιλογές. Για το λόγο αυτό δεν κατανοώ την θέση των σοσιαλιστών καθώς και άλλων πολιτικών ομάδων που δεν θέλουν να ληφθεί θέση. Εμείς έχουμε προτείνει τρεις συμβαστικές τροπολογίες που αποτελούν συμβιβασμό μεταξύ ενός άριστου ε, δικαίου συμβάσεων και του λεγόμενου toolbox όπου οι συμβάσει ηλεκτρονικού εμπορίου θα υπόκειται στο εναλλακτικό αυτό μηχανισμό, ενώ όλα τα υπόλοιπα θα πηγαίνουν στο toolbox. Στις συμβαστικές τροπολογίες αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην παράγραφο 9 οι συμβαστικές τροπολογίες διαβάστηκαν λίγο πριν από τη συνεδρίαση σε όλους τους κοιόδης ηγητές. Εγώ πάντως θα χαρώ εάν υπάρξει σημαντική υποστήριξη υπέρ της εκθέσεως του κ. Μάιερ και θέλω να ευχαριστήσω έξω ονοματός του όλες και όλους τους κοιόδης ηγητές και ελπίζω η προσπάθεια αυτή για να θεσπιστεί ευρωπαϊκό ε, δίκαιο συμβάσεων να επιτύχει. Σε ευχαριστούμε πολύ κύριε Σουβά. Η κυρία Στάιλερ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ τον Ανδρέα Σουβάμπα για το ότι αντικατέστησε στον συνάδελφο και για την παρουσίασή του. Νομίζω εύγλωτα υπεγράμισε το τι συμβαίνει και ποιες διαφορές υπάρχουν σε σχέση με την προσέγγιση. Πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι για τις εναλλακτικέ δυνατότητες και πολλοί από εμά που θα ήθελαν μελέτη επιπτώσεων όλων των εναλλακτικών δυνατοτήτων πριν από την λήψη απόφασης Προσπαθήσαμε να υποβάλουμε κάποιες τέτοιες προτάσεις, ε, όμως ε, η θεμελιώδης ε, θέση στην οποία βρισκόμαστε. Θα ήθελε ο κύριος Μάγιας να υιοθετήσουμε μια ανάποψη ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση των διαφορετικών προτάσεων διότι δεν έχει γίνει μια μελέτη επιπτώσεων. Μέχρι την επίλυση αυτού του θέματος, ε, το θέμα της μελέτης επιπτώσεων θα πρέπει να αναλύει όλες τις εναλλακτικέ λύσεις που βρίσκονται στο τραπέζι και θα πρέπει να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις και γνωρίζοντας ε, το τι θα συνεπάγονται αυτά. Λοιπόν, σε σχέση με τις διαφορετικές απόψεις αυτό είναι σημαντικό. Προφανώς ε, θα πρέπει να συνεχίσει η συζήτηση, να συνεχίσει η συζήτηση των διαφορετικών θεμάτων. <coughs> Αν δεν επιληθεί όμως αυτό το θέμα, δεν είναι δυνατόν να θεωρήσουμε ότι επιλύεται το θέμα της ε, ε μελέτης επιπτώσεων. Και έτσι δύσκολα θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε την ε, συμβαστική τροπολογία όπως προτάθηκε από τον κύριο Μάης. Τώρα επαρκούμε σε αυτό, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Από πλευρά Κρόισμαν, νομίζω εκείνος θέλει να παρέμβει τώρα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σμιτ θα ήθελε ω σκιώδη εισηγητή τη ομάδα Άντε να ευχαριστήσει τον εισηγητή και του άλλου σκιώδη για καλή δουλειά που έγινε. Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό είναι ένα αρκετά καλοσυζητημένο θέμα σε σχέση με τις επιπτώσεις όσον αφορά την νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο σήμερα. <clears throat> Από πλευρά Άντε υποστηρίζεται η πρόταση του κυρίου Μάιες που ευθυγραμμίζεται ως θέση με τον εισηγητή της Επιτροπής Γιούρη. Εδώ σε σχέση με το συμβατικό δίκαιο και για την περαιτέρω ανάπτυξη του toolbox αυτό είναι αρκετά προβληματικό για κάποιες ομάδες. Όμως ο κύριος Σμιτ και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή θα πρέπει να εξεύρουμε μια λύση, λέει, που θα δώσει στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων να γνωρίζει τα στοιχεία, να γνωρίζει ποια είναι η άποψή μας και ποια συνέχεια πρέπει να δοθεί σε αυτό το εγχείρημα. Επίσης, από την Άντε, από το σκιώδη σητή της ΑΝΤΕ υπογραμμίζεται η σημασία της μελέτης επιπτώσεων σε σχέση με τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η επίπτωση του Ευρωπαϊκού Συμβατικού Πλαισίου στο Εθνικό Συμβατικό Πλαίσιο. Θεωρεί ο κύριος Σμιτ ότι είναι αναγκαίο να θίγονται αυτά τα θέματα σε σχέση με την ε, Διεθνή Σύμβαση για την ε, ε, Πώληση Αγαθών είναι πολύ σημαντικό να ληφθούν αυτά τα πράγματα υπόψη και να λαμβάνονται υπόψη σε σχέση με τη μελέτη επιπτώσεων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Um, Κυρία Ρούλα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να συμφωνήσω σε μεγάλο βαθμό και εγώ με αυτά και εμείς δίνουμε ιδιαίτερη σημασία να γίνει αξιολόγηση επιπτώσεων. Θέλουμε μια ανοιχτή διαδικασία γι' αυτό. Θέλουμε και τις δύο δυνατότητες να σα αφήσουμε ανοιχτές και το εθελοντικό, εθελούσιο πλαίσιο και το toolbox και τα δύο πρέπει να παραμένουν ανοιχτές δυνατότητες και είναι σημαντικό στην μελέτη επιπτώσεων να δούμε και τις επιπτώσεις στο εθνικό δίκαιο που θα συνεπάγεται κάτι το πρωτού απόφαση. Από την άλλη πλευρά Πρέπει να δούμε ότι έχει προηγηθεί εργασία ήδη σε αυτό το επίπεδο. Δεν θέλουμε να ολοκληρώσουμε τελεσίδικα τώρα αυτή τη ε, διαδικασία, αλλά θέλουμε να μείνει ανοιχτή αυτή η διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη και τις δύο εναλλακτικέ δυνατότητες. Και οι δύο δυνατότητες πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές. Ζητούμε να γίνει μελέτη επιπτώσεων και να δούμε μετά στη συνέχεια τα αποτελέσματα ιδιαίτερα προσεκτικά. Αν υπάρχει εθελοντικό πλαίσιο συμβάσεων, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και τη θέση της ε, Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, αυτά θα πρέπει να συνάδουν με τα όσα είναι δεδομένα ήδη σήμερα όσον αφορά το κεκτημένο για την προστασία καταναλωτών επί του οποίου εργάζεται ο κύριος Σβάμπ. Πρέπει να αναμείνουμε να υπάρξει μια ε, μετεξέλιξη και συγχώνευση όλων των διαφορετικών τομέων ώστε να υπάρχει μια σωστή επισκόπηση ώστε μέσα στο συμβατικό δίκαιο να συμπεριλαμβάνονται όλα αυτά τα στοιχεία και να μπορούμε να δούμε ποια θα είναι η συνολική επίπτωση αυτών. Ευχαριστώ. Thank you very much. Mr. Fox. Ευχαριστώ. Fox παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω μεγάλους δισταγμούς για τα ωφέλη αυτής της ε, εθελοντικής προσέγγισης, διότι στην υλοποίηση, στην εφαρμογή, καθότι βλέπω, θα υπάρξουν επιζήμες επιπτώσεις για τους καταναλωτές. Ένα εθελοντικό τέτοιο μέσο δεν θα μπορεί να είναι εθελοντικού χαρακτήρα για τους ε, καταναλωτές και θα πρέπει οι συναλλασσόμενοι να αποφασίσουν τελεσίδικα ποιο θα είναι το ε, κύριο στοιχείο το οποίο θα πριτανεύει. Διότι στα κράτη-μέλη όπου υπάρχει ε, χαμηλό επίπεδο προστασίας καταναλωτών αυτό θα παραμείνει έτσι με αυτό σε αυτό το πλαίσιο. Όμως σε άλλα κράτη όπου υπάρχει υψηλό επίπεδο προστασίας καταναλωτών όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και στη Σκανδιναβία θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί περισσότερο για να διασφαλιστεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας καταναλωτών. Είναι πολύ δύσκολο να δω πώς θα μπορέσει αυτό το εθελοντικό μέσο να ωφελήσει τους καταναλωτές. Κατά τα άλλα συμφωνώ με σχεδόν όλα όσα προανέφερε η κυρία Στάιλερ. Με ενθάρρυναν όμω τα σχόλια που έκανε η κυρία Ρούλε για την ανάγκη να υπάρξει σφαιρική πλήρη μελέτη επιπτώσεων και για τι δύο αυτέ εναλλακτικέ δυνατότητε. Και ελπίζω ότι παρακολουθεί και προσέχει ο κύριο Σβάμπ εξ ονόματο του συναδέρφου. Διότι <clears throat> γνωστοποιούνται οι προτιμήσεις όσον αφορά τις απόψεις του. Όμως και οι δύο αυτές ε, εναλλακτικές δυνατότητες θα πρέπει να έχουν πλήρη μελέτη επιπτώσεων. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να λάβουμε κάποια απόφαση. Να μην αποκομίσει την εντύπωση ο εισηγητής ότι υπάρχει κάποια προτίμηση για το εθελοντικού χαρακτήρα μέσω προτού γίνει μια πλήρης μελέτη επιπτώσεων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Okay. Um, thank you very much. I think I don't see else. Δεν θέλει κανένας να ζητάει το λόγο. Δεν θέλει να ζητήσει το λόγο ο κύριος Μάιερ από την Επιτροπή να σχολιάσει. Καταλαβαίνω ότι αυτά που είπε ο κύριος Φόξ για τους καταναλωτές ε, συζητήθηκαν την περασμένη Παρασκευή, την ε, Ευρωπαϊκή Μέρα για τους καταναλωτές. Εγώ δυστυχώς δεν μπόρεσα να πάω. Και επίσης, με βάση τις δεσμεύσεις που, που πήρε η Κομισιόν, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μια ε, μελέτη αντικτύπου και για τις δύο εναλλακτικέ λύσεις. Αλλιώς όλη αυτή η διαδικασία για την έξυπνη νομοθεσία θα, δεν θα έχει κανένα νόημα. Λοιπόν, ο εκπρόσωπο Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, για αυτή την ευκαιρία. Θα είμαι και πολύ σύντομο Καταρχήν, από σχεδόν όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες και όλους τους προλαλήσαντες ε, ζητήθηκε να υπάρξει μια πλήρης μελέτη επιπτώσεων. Είναι φυσικό θα το κάνουμε αυτό και θα ανταποκριθούμε έτσι σύμφωνα με τις οδηγίες ε, που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση αυτού του έργου. Στην μελέτη επιπτώσεων θα λαμβάνει υπόψη όλες τις εναλλακτικές λύσεις αυτό το πλαίσιο μελετών επιπτώσεων. Κατά τούτο λοιπόν αυτό το σημείο θα ληφθεί υπόψη και έτσι θα ενταχθεί. Ένα άλλο σημείο που ήθελα να αναφέρω, το οποίο έθιξε ο κύριος Σβάμπ. Ο κύριος Σβάμπ είπε ότι το κοινοβούλιο, λέει το Ευρωκοινοβούλιο <clears throat> και άλλοι εμπλεκόμενοι φυσικά, θα ήθελαν το αποτέλεσμα της ομάδας επαϊόντων να δουν ποιο είναι το ε, αποτέλεσμα των εργασιών τους. Είναι απόλυτα κατανοητό αυτό και πολύ σημαντικό σημείο. Κάτι που στην ε, διαβούλευση έχει πολυσυζητηθεί διότι τα εμπλεκόμενα ε, μέρη που έχουν τοποθετηθεί αντίστοιχα είπαν θα, θέλαμε να δούμε το κείμενο πρώτα και τα στοιχεία προτού λυθεί τελεσίδικη απόφαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έχει δημοσιεύσει κάποια κεφάλαια των ε, αποτελεσμάτων των εργασιών των ε, πραγματογνωμόνων και μετά το τέλος της εργασίας ε, της ομάδας των εμπειρογνωμόνων θα δημοσιευθεί το σύνολο του κειμένου ώστε έτσι φυσικά να είναι διαθέσιμο στο Ευρωκοινοβούλιο και στα κράτη-μέλη που θέλουν να δουν το σύνολο του κειμένου και να αποκρισταλώσουν απόψεις λαμβάνοντας υπόψη υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία. Όπως όμως η κυρία Ρούιλε πολύ σωστά προανέφερε, η όλη αυτή η διαδικασία για τη συζήτηση και την επεξεργασία διαρκεί σχεδόν πάνω από 10 χρόνια ήδη. Και πραγματικά θα είχε νόημα εδώ να, ε, ε, όχι να σταματήσουμε αυτή τη διαδικασία, αλλά να ολοκληρωθεί, να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί, ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα και σε αρκετό βάθος για την αξιολόγηση των μελετών επιπτώσεων. Μια τελευταία παρατήρηση, επειδή σχεδόν όλοι οι προλαλήσαντες τόνισαν ποια, άσχετα από το ποια αποτελέσματα θα πρέπει να έχουμε, θέλουμε να διασφαλίσουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας καταναλωτών με οποιοδήποτε κείμενο θα έχουμε. Και έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακριβώς έτσι το αντιμετωπίζει και η ίδια. Πράγματι, όταν θα έχουμε ένα μέσο συμβατικό σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, όχι μόνο θα πρέπει να έχουν ε, οι καταναλωτές τα ωφέλη ενός οικονομικού πλαισίου που θα μεγεθυνθεί, διασυνοριακά, δηλαδή θα πολλούνται αγαθά και θα συναλλασσόμεθα με τέτοια αγαθά ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη επιλογή διασυνοριακά από αυτή την προσφορά αλλά και αυτά τα προϊόντα να μπορούν να τα αγοράζουν οι καταναλωτές σε πιο προσιτές τιμές, πιο φθηνά. Αλλά επίσης σημαντικό, οποιοδήποτε μέσο του Ευρωπαϊκού Συμβατικού Πλαισίου πρέπει να διασφαλίζει ότι η πλειοψηφία των Ευρωπαίων καταναλωτών θα έχουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας. Δηλαδή νομικά υψηλότερο επίπεδο προστασίας σε σχέση με το σημερινό κεκτημένο. Και αυτό είναι ένα θεμελιώδες στοιχείο στον στόχο που προσπαθεί να υλοποιήσει η ομάδα επαϊόντων, η ομάδα πραγματογνωμόνων και μπορώ να σας διασφαλίσω ότι στην ήδη εργασία αυτής της ομάδας πραγματογνωμόνων διασφαλίζεται ένα σαφώς υψηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Θα το δείτε αυτό με τη δημοσιοποίηση, με τη δημοσίευση του κειμένου. Και για να πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα μόνο, το σημερινό κείμενο των πραγματογνωμόνων ε, σε σχέση με το συμβατικό ε, πλαίσιο ξεπερνά κατά πολύ τα εσκαμένα. Δημιουργεί λοιπόν, ε, διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας καταναλωτών. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως στόχο και έτσι και για τους πραγματογνώμονες της ομάδας εργασίας. Ευχαριστώ για την προσοχή. Well, Ευχαριστώ την Επιτροπή. Θα ψηφίσουμε αύριο. Ε, ο κύριος Μάιερ δεν θα είναι εδώ αύριο, ε, οπότε κύριε Σβάμπ, αν θέλετε να κάνετε τα τελικά σας σχόλια σήμερα. Κύριε Σβάμπ, ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους που παρενέβησαν. Ο συνάδελφος Μάιερ προτιμά όσον αφορά <clears throat> την μελέτη επιπτώσεων της τροπολογίας 24 και 26 <clears throat> και σε σχέση με τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί. Πρόκειται για το θέμα, αν επιτρέπετε την αναφορά στον συνάδελφο Φόξο, παρατήρησα, άκουσα πολύ προσεκτικά τα όσα είπε. Στην τροπολογία 26 που έχει τεθεί, πρόκειται για το θέμα αν θα εξεταστεί στη μελέτη επιπτώσεων ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει τροποποίηση του νομικού πλαισίου, ότι δηλαδή δεν θα ληφθούν κάποια άλλα μέτρα. Πιστεύω ότι όμως όταν έχουμε μπροστά μας την κατάσταση για τις εγγυήσεις, τα εχέγγυα που δίνονται και έχουμε διαφορετικά πλαίσια εγγυήσεων, εγγυητικά πλαίσια στην Ευρώπη, είναι προφανές ότι πανευρωπαϊκά χρειάζεται μία ε, ενιαία προσέγγιση, ένα θα έλεγα πλαίσιο δημιουργίας εγγυήσεων. Και έτσι δεν θα πρέπει από τις διαφορετικές δυνατότητες να αποκλείσουμε μεν κάτι, αλλά θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάτι κοινό και σε σχέση με την τροπολογία 26 ο κύριος Μάγες είναι πρόθυμος να συζητήσει αυτά τα θέματα. Θα δούμε κατά πόσο θα μπορέσει να παραστεί αύριο. Η κυρία Στάιλερ προς παρόμοια κατεύθυνση τοποθετήθηκε. Βρίσκω ότι όλοι οι συνάδελφοι ζητούν μια ενιαία τέτοια κοινή προσέγγιση, διότι αναγνωρίζεται πόσο δύσκολη είναι αυτή η πορεία βέβαια όμως παρόλα αυτά πρέπει να διαπιστώσουμε και να πούμε ότι ο κατακαιρματισμός, ο νομικός κατακαιρματισμός για την ενιαία εσωτερική αγορά δημιουργεί προβλήματα και δημιουργεί προβλήματα και για τους καταναλωτές. Κάτι πρέπει να κάνουμε μακροπρόθεσμα και για τις μελέτες επιπτώσεων για να καταλήξουμε σε ένα πιο κοινό πλαίσιο. Καλό θα ήταν λοιπόν αν μπορούσαμε έτσι να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κύριε Σβάμπ, που αντικαταστήσατε τον κύριο Μάγερ. Στις 10 ε, και 4 από το αύριο ψηφίζουμε αυτή την έκθεση και άλλες. Σας ε, παρακαλώ να φέρετε τις ε, ηλεκτρονικές σας κάρτες. Ούτως ή άλλως σας στείλω και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το επενθυμίσω. Περνάμε τώρα σε ένα νέο φάκελο. Ο κύριος Ταραμπέλα είναι ο εισηγητής μας. Είναι μια άλλη νομοθετική γνωμοδότηση για μια πρόταση κανονισμού για την ε, χρήση των φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορούχων ενώσεων σε οικιακά απορριπαντικά πλυντηρίων ρούχων. Πολύ ενδιαφέρον θέμα για την Επιτροπή. Θα δούμε, κύριε Ταραμπέλα, ποια είναι η διάσταση της ενίας αγοράς. Θα ήθελα παρακαλώ να παρουσιάσετε την έκθεσή σας. Μετά θα ακούσαμε την κυρία Κόμη που αντικαθιστά την κυρία Σαρτόρτ, Κρόιτσμαν, Ρούλερ, Φόξ, Σαβίνη που δεν έχει επιστρέψει, αλλά αυτά μετά τον κύριο Ταραμπέλα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω, καθώς και, το... και τους, εισηγη... τους συντονιστές και το Προεδρείο που επιτρέψατε να διατυπώσουμε μια γνωμοδότηση, κάτι που δεν προβλεπόταν. Αυτή η πρόταση ε, κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκινάει από δύο διαπιστώσεις ότι τα φωσφορικά άλατα στα απορριπαντικά είναι υπεύθυνα εν μέρη για, τον ευτροφισμό. Δηλαδή ε, δημιουργούνται όλο και περισσότερα ε, φύκια και αυτό ε, δημιουργεί ανισορροπία. Ε, επίσης δεν υπάρχει, ε, υπάρχει στρέβλωση του, της εσωτερικής αγοράς. Αυτό σημαίνει και πρόβλημα στο κόστος για τους καταναλωτές και για να ρυθμιστούν αυτά τα προβλήματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, λέει ότι θα πρέπει να μειώσουμε κατά 0,5% την, τις φωσφορικές ενώσεις ε, στα απορριπαντικά. Το 2014 θα δούμε τι γίνεται με τις φωσφορικές ενώσεις σε άλλα απορριπαντικά που χρησιμοποιούνται στα πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων. Λοιπόν, βασίζομαι στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά από τι ε, διαβουλεύσει με τα διάφορα μέρη διαπιστώνω ότι η πιο ισορροπημένη προσέγγιση είναι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, συνοψίζοντα σε τέσσερα σημεία ποια είναι η πρόταση. Καταρχά, θα πρέπει ε, στα απορριπαντικά ε, για τα ρούχα να μειώσουμε τα, φωσφορικά άλατα λόγω του ευτροφισμού. Τα απορριπαντικά δεν είναι ο βασικός ένοχος για τον ευτροφισμό με βάση ένα ε, Ισπανικό Ινστιτούτο ε, που έκανε μια μελέτη από ε, τη ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι υπεύθυνα τα απορριπαντικά αυτά για το 6% του ευτροφισμού στην Ευρώπη. Με διάφορες διαφορές ανάλογα με τις ροές των, των υδάτινων οδών. Ανάλογα με το αν οξυγονώνεται περισσότερο το νερό ή όχι. Αλλά γενικά κατά μέσο όρο 6% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, επομένως, τα απορριπαντικά ε, με φωσφορικά άλατα δεν ε, συμμετέχουν κυρίω στον ευτροφισμό, αλλά κυρίως τα ανθρώπινα και ζωικά α, απόβλητα. Ε, επομένως, θα πρέπει να εστιάσουμε κυρίω στον καθαρισμό των, α, λιμάτων. Των λιμάτων. Ε, θα πρέπει να περιορίσουμε λοιπόν τα φωσφορικά αλλά στα απορριπαντικά. Υπάρχουν οι φωσφονάτες, το κυτρικό άλας. Αυτές είναι διάφορες εναλλακτικέ λύσεις. Αλλά μερικές φορές δεν μπορούμε να απαλλαγούμε τελείως από τα φωσφορικά άλατα και τις φωσφορούχες ενώσεις. εξού και να περιοριστούμε στο 0,5%. Ορισμένε φορέ λέμε 0,5% ε, γραμμάρια αναδόση απορριπαντικού. Ε, καλό είναι λοιπόν να βάλουμε ένα όριο αριθμητικό και όχι ποσοστό. Για να μην βρούνε οι βιομηχανίες ε, παραθυράκια για να αποφύγουν αυτή την διάταξη. Αυτό που συμβαίνει στο Βέλγιο, ας πούμε, που έχουμε μειώσει την, το την περιεκτικότητα από το 2004 σε φωσφορικά άλατα στο 0,5% δεν ε, είδαμε μια αρέωση το, σε φωσφορικά άλατα και στην πραγματικότητα έχουμε πολύ πιο συμπυκνωμένα απορριπαντικά και τελικά ξεπερνάμε αυτό το 0,5%. Ε, η Γερμανία έχει αυτό το όριο το 0,5%. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Ε, υπάρχει μείωση αλλάζει η συμπεριφορά της βιομηχανίας, μήπως ε, ε, τι κάνει, αραιώνει τα απορριπαντικά ή τα συγκεντρώνει περισσότερο. Τώρα, για τα πλυντήρια πιάτων. οι καταναλωτές δεν θέλουν ε, απορριπαντικά τα οποία δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους που δεν, δεν πλένουν στην πραγματικότητα. Ε, έχουμε ένα Ινστιτούτο που έκανε κάποιες μελέτες που δείχνουν ότι καμία διαφορετική λύση δεν υπάρχει ακόμα αποτελεσματική. Παραδείγματο χάρη, ε, όταν παίρνουμε τα πιάτα με απορριπαντικά χωρί φωσφορικέ ε, ενώσει, ε, στην πραγματικότητα πρέπει να τα ξαναπλύνουμε γιατί υπάρχουν κάτι ε, υπολείμματα άσπρα ή θα πρέπει να αυξήσουμε τη θερμοκρασία. Οπότε δεν κάνουμε τίποτα για το περιβάλλον. Επίση, έχουμε ένα πολύ σκληρό νερό με πάρα πολύ, πολύ ας πούμε ασβέστιο μέσα ε, επομένως θα πρέπει να χρησιμοποιούμε μεγαλύτερα προγράμματα, μεγαλύτερης διάρκειας δηλαδή, αν δεν χρησιμοποιούμε απορριπαντικά με φωσφορικές ενώσεις. Ε, προφανώς Κομισιόν έχετε δίκιο ότι μέχρι το 2014 πρέπει να κάνουμε μια αξιολόγηση για την ε, χρήση των φωσφορικών ενώσεων ε, στα πλυντήρια πιάτων. Επίση, θα πρέπει να δούμε τον κύκλο ζωής αυτών των προϊόντων. Από την αρχή μέχρι το τέλος, μέχρι την εξάλληψη, την εξαφάνιση του προϊόντος από τον καταναλωτή. Ε, έχει, έχουν γίνει μελέτες για τις εναλλακτικά, τα εναλλακτικά διαλύματα. Ε, και πρέπει να δούμε, ε, εποφελεί το περιβάλλον, εποφελεί το καταναλωτή. Κάτι άλλο. Μέχρι στιγμή θα πρέπει να ενημερώνουμε τον καταναλωτή. Στην πραγματικότητα δεν ενημερώνεται καλά. Οι καταναλωτέ θα πρέπει να ενημερώνονται ε, με κείμενα, ε, με λογότυπου, να λέμε παραδείγματο χάρη ότι αν βάζετε περισσότερο ας πούμε, απορριπαντικό δεν σημαίνει ότι είναι πιο αποτελεσματική η πλήση. Ε, είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε ε, ανακυκλώσιμες συσκευασίε κτλ. Ή να χρησιμοποιείτε αυτά τα απορριπαντικά που πολλούνται σε εναλλακτικέ συσκευασίε και τα μεταγγίζετε ε, στα αρχικά μπουκάλια. Επίσης, μερικές φορές ε, υπάρχουν βιομηχανίες οι οποίες κάνουν διαφήμιση και λένε «Α, εμείς έχουμε ε, απορριπαντικά τα οποία έχουν φωσφορικές ενώσεις κάτω από το 0,5%. Ε, με αυτό είναι Υποχρέωση ούτως ή άλλως. Απλώς κάποιοι το διαφημίζουν, κάποιοι όλοι. Δεν θέλ, κάποιοι όχι. Ε, δεν θέλω να γίνεται κάτι τέτοιο. Ε, θα πρέπει να ακούσουμε τους πάντες, θα πρέπει να δούμε ε, από τη μία την προστασία των καταναλωτών, από την άλλη το περιβάλλον και από την άλλη τη διάσταση της εσωτερικής αγοράς. Δεν θα πρέπει να προτάξουμε κάποια συμφέροντα ει βάρο κάποιων άλλων. Θα πρέπει να φτιάξουμε ένα κανονισμό το οποίο είναι, ο οποίο είναι ισορροπημένο. θα σέβεται το περιβάλλον, προστατεύει καλύτερα του καταναλωτέ και να βρούμε τελικά ισορροπημένες λύσεις. Δεν θέλω να έρθουμε σε αντιπαράθεση, δεν θέλω να βγάλουμε τα μαχαίρια, παρότι μου αρέσει η συζήτηση επί ε, συγκεκριμένων προτάσεων, επιχειρημάτων και ιδεών. Thank you very much indeed. Ευχαριστούμε πολύ και για την ε, επεξεργασία αυτών των ε, λεπτομερικών θεμάτων και για τους σκιώδεις εισηγητές. Εσείς κυρία έχετε τον λόγο πρώτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, μιλώ εξ ονόματος του κυρίου Σαρτόρη, που λόγω προβλήματος με τις εναέριες μεταφορές δεν μπορούσε να έρθει εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ταραμπέλα για το άνοιγμα και τη διαθεσιμότητά του που έδειξε από την αρχή αυτής της νομοδότησης. Καλό είναι να εμπλακούμε κι εμείς, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε αυτή την εναρμόνιση και σε αυτόν τον τομέα που χρειάζεται. Η εθνική νομοθεσία σε ό,τι αφορά τις ενώσεις αυτές ε, δείχνει ε, μεγάλες διαφορές. Στην Ισπανία δεν υπάρχει καμία ανώτατη οριακή τιμή ε, στην περιεκτικότητα των φωσφορικών ενώσεων. Από το 2012 στην Γαλλία δεν θα υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης φωσφορικών ενώσεων, ενώ εμείς θα έχουμε κάποιες ανώτατες οριακές τιμές στην Ιταλία. Χρειάζεται λοιπόν μία εναρμόνιση. Όχι μόνο για την παραγωγή και τη θέση στην εμπορία αυτών των προϊόντων, κάτι που χρειάζεται παρόλα αυτά, αλλά κυρίως για να αντιμετωπίσουμε ε, τη χρησιμοποίηση και την διάθεση αυτών των προϊόντων. Να δούμε πώς ε, αντιμετωπίζουμε μάλλον την διάθεση αυτών των προϊόντων. Η μείωση των φωσφορικών αλάτων στα απορριπαντικά είναι δεδομένο, όπως είπε και ο κύριος Ταραμπέλα πια. Ε, οι βασικοί λόγοι, παρότι δεν είναι οι μόνοι που ανάγκασαν τη βιομηχανία προς αυτήν την κατεύθυνση, συνδέονται κυρίως με τον κίνδυνο του ευτροφισμού των υδάτων ε, είναι ε, από τους κύριους υπεύθυνους του εθνοφισμού ε, οι φωσφορικές ενώσεις. Όχι λόγω της χρησιμοποίησης του φωσφόρου, αλλά των φωσφορικών αλάτων. Ο φωσφόρος σε μικρές ποσότητες δεν δημιουργεί ευτροφισμό, αλλά μόνο τα φωσφορικά άλατα. Επίσης, για να μην υπάρξουν επικαλύψεις, καλό θα ήταν να ξεκινήσουμε ένα προβληματισμό για τον τρόπο που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ε, θα να ρυθμίσουμε μάλλον ε, τις φωσφορικές ενώσεις, τα φωσφορικά άλατα. Νομίζω ότι πρέπει να τροποποιήσουμε την ε, πρόταση της Κομισιόν, να βάλουμε ε, ανώτατες οριακές τιμές, ε, δηλαδή ποσοτικά όρια και όχι ποσοστά, τα οποία μας παραπλανούν. Αν αποφασίσουμε να περιοριστούμε στη ρύθμιση των ορίων των φωσφορικών αλάτων, τότε καλό θα ήταν να βρούμε και εναλλακτικέ λύσεις ελάχιστη δηλαδή, ε, ελάχιστα ποσότητα φωσφόρου και φωσφονάτες. Νομίζω ότι οι συζητήσεις με τους άλλους κοιόδης εισηγητές θα γίνουν με αποτελεσματικό τρόπο, ε, όπως ακριβώς ξεκίνησαν και ελπίζω να συνεργαστούμε για να βελτιώσουμε κάποια σημεία ευαίσθητα του κειμένου της Κομισιόν. Ευχαριστώ ακόμα μια φορά τον κύριο Ταραμπέλα για τη δέσμευσή του και σας ε, δηλώνουμε και εμείς διατεθειμένοι από πλευράς μας να συνεργαστούμε απόλυτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Κρόιτσμαν. Ο κατακαιρματισμός της αγοράς απορριπαντικών προκαλεί περιτά έξοδα και για τις επιχειρήσεις και για την διοίκηση. Και αυτό μου φαίνεται καλή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εναρμονιστούν οι εθνικές διατάξεις για την ε, χρήση φωσφορικών αλάτων και συγχαίρω τον κ. Ταραμπέλα. Συμφωνώ ότι μια ενδεχόμενη νομοθετική πρόταση και για απορριπαντικά πλυντηρίων αλλά και πλυντηρίων πιάτων Χρειάζεται μια ρύθμιση λοιπόν μέχρι το 2014. Η ερώτηση είναι μήπως πρέπει να γίνει και νωρίτερα. Ίσως το 2012 ή 2013 εάν είναι σε θέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας υποβάλει τη σχετική αξιολόγηση ώστε να μπορέσουμε να αντιδράσουμε στα γεγονότα τα οποία θα μας υποβάλει. Το ίδιο ισχύει για ενδεχόμενους περιορισμούς για την χρήση απορριπαντικών στον βιομηχανικό τομέα. Όπως διαβάσαμε στη μελέτη επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέχρι τώρα δεν υπάρχουν όριμα, όριμες τεχνολογικά λύσεις για τον βιομηχανικό τομέα. Στα απορριπαντικά πλυντηρίων πιάτων υπάρχουν ακόμα προβλήματα για την ε, αποδόμησή τους. Χρειάζεται λοιπόν περαιτέρω έρευνα και αυτό βέβαια αποβαίνει για την ώρα σε βάρος των μικρών και μισών επιχειρήσεων. Ενδιαφέρουσες είναι οι δηλώσεις της Κομισιόν σχετικά με τη μελέτη για ενδεχόμενη απόλυτη απαγόρευση των φωσφορικών αλάτων. Οπότε θα έπρεπε να κλείσουν πολλές εκατοντάδες επιχειρήσεις και να χαθούν 3 με 5 χιλιάδες θέσεις εργασίας. Άρα χρειάζεται να αναζητηθούν Εναλλακτικέ επιλογές και χρειάζεται προσεκτική προσέγγιση του θέματος, διότι δεν έχει κανένα νόημα να προσπαθούμε αφενός να δημιουργήσουμε θέσει απασχόλησης στην ενιαία αγορά και από την άλλη μεριά με βιαστικέ και απρόσεκτε κινήσεις να συμβάλλουμε στην μεγάλη απώλεια θέσεων εργασία. Γι' αυτό και εκφράζουμε την ικανοποίησή μα και πάλι για τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής και εδώ χρειάζεται να συζητηθούν εάν θα πρέπει οι περιορισμοί αυτοί να είναι ποσοστιαίοι, αναλογικοί ή απόλυτοι, ή θα μείνουμε σε αυτό 0,5%. Κατά τα άλλα είμαστε ανοιχτοί για κάθε είδους συζήτηση και τροπολογίες, αλλά θεωρούμε ότι το πρόβλημα, το οποίο παρουσιάζεται βέβαια και στο impact assessment, είναι ότι πολλές χώρες δεν έχουν εγκαταστάσεις καθαρισμού και εκεί βεβαίως πλήττονται περισσότερο από τις δυσμενείς επιπτώσεις από ότι άλλες χώρες. Άρα θα έπρεπε να φροντίσουμε ώστε και στις χώρες που έχουν τέτοιες ελλείψεις να δημιουργηθούν οι κατάλληλες ε, εγκαταστάσεις καθαρισμού των υδάτων. Σας ευχαριστώ. Uh, thank Σας ευχαριστώ κυρία Ρούλε. Συμφωνώ, βεβαίως είμαι υπέρ των εγκαταστάσεων καθαρισμού. Αυτά όμως επίσης κοστίζουν λεφτά. Πρέπει λοιπόν να γίνει σωστός υπολογισμός. Λέμε ότι θα υπάρξει απώλεια θέσεων απασχολήσεως από τις απαγορεύσεις, αλλά πρέπει να εξετάσουμε και ποιο είναι το κόστος σε βάρος του περιβάλλοντος. Στην Σουηδία υπάρχει απαγόρευση. Η Γαλλία επίσης, στην Γαλλία επίσης επίκειται να ε, θεσπιστεί απαγόρευση. Έχει λοιπόν νόημα να γίνει μια προσπάθεια εναρμόνισης στο ευρωπαϊκό επίπεδο και γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να επεκταθεί η ε, απαγόρευση και στις εγκαταστάσεις πλήσεως πιατικών με τις απαραίτητες μελέτες βέβαια, αλλά πρέπει να περιληφθούν και αυτές οι εγκαταστάσεις πλήσεως πιάτων. Ευχαριστώ και τον εισηγητή αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις προτάσεις της, διότι δεν έχει νόημα τα πράγματα να, μείνουν μονάχα στο επίπεδο των χωρών μελών, διότι έτσι προκαλείται στρέβλωση στην αγορά. Πρέπει να εναρμονιστεί. Άλλωστε και το νερό δεν περιορίζεται, το, το νερό κυκλοφορεί παντού και επιβαρύνεται και αυτό είναι σε βάρος όλων μας εν τέλει. Ευχαριστώ. Φόξ. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ταραμπέλα για την δουλειά που έκανε και για τη συνεργασία και θέλω να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το αίσθημα της ε, πειθαρχίας που κατέδειξαν και το ότι δεν ε, επεκτάθηκε το θέμα των, ε, των καθαριστικών των πιατικών και για την απώλεια των θέσεων απασχόλησης σε σχέση με την απαγόρευση των φωσφατούχων και για τη διαφοροποίηση μεταξύ φωσφορούχων και φωσφατούχων θα έπρεπε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μελετήσει προσεκτικά τις επιπτώσεις που θα είχε μια απλή απαγόρευση και να δούμε κατά πόσο θα υπήρχε ένα θετικό πλαίσιο. Προτού ληφθεί μια τέτοια απόφαση, θα ήθελα να δω ποιο είναι το κόστος σε σχέση με τις δαπάνε που θα προκληθούν για τις βιομηχανίες. Δεν έχω καμία αντίρρηση σε σχέση με μια τέτοια απαγόρευση για τα φωσφατούχα. Υπό τον όρο ως προϋπόθεση ότι θα συνέχιζε η βιομηχανία να χρησιμοποιεί λιγότερο ζημιογόνες ε, ουσίες ε, φωσφατούχων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω σε σχέση με την συνενετική προσέγγιση και ευχαριστώ και πάλι για τη συνεργασία. Σα ευχαριστούμε πολύ. Δεν βλέπω κάποιοι άλλοι να θέλουν να παρέμβουν σε αυτή τη συζήτηση. Έχουμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ. Έχασα τα χαρτιά μου. Μπορείτε να μας πείτε ποιο είναι το όνομά σας και να μας απαντήσετε, να ανταποκριθείτε σε σχέση με τις παρατηρήσεις που έγιναν. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κλάους Μπέρεντ είναι το όνομά μου επικεφαλής μονάδας ε, στην ε, μονάδα ε, επιχειρήσεων Enterprise, καθώς επίσης και για τον κανονισμό για τις, τα αντιρρυπαντικά. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ταραμπέλα και τους χειώδεις εισηγητές για τα πολύ θετικά σχόλια που ακούσαμε και την υποστήριξη της πρότασης που έχουμε υποβάλει πράγματι απέρευσε από μια πολύ σοβαρή σε βάθος ανάλυση των επιπτώσεων και των στοιχείων που χρησιμοποιήσαμε σε σχέση με αυτές τις ουσίες και για τις ε, πιθανές εναλλακτικέ λύσεις και τις επιπτώσεις είτε στην ανθρώπινη υγεία είτε στο περιβάλλον είτε και την τεχνική δυνατότητα μελέτης επιπτώσεων και εφικτότητας. Θα ήθελα να ανταποκριθώ στα σχόλια του κυρίου Ταραμπέλα ότι δεν είναι μόνο η μόνη πηγή των φωσφατούχων αυτές οι ουσίες. Η σκέψη μας καθορίστηκε από την αρχή της αναλογικότητας. Γι' αυτό περιορίσαμε την πρόταση αρχικά στην ε, πραγματική απαγόρευση αυτών των ε, φωσφατούχων όσον αφορά τα ε, καθαριστικά, αλλά επίσης και σε σχέση με την δυνατότητα όπου υπάρχουν εναλλακτικέ ε, ε, άλλες ε, ύλες ή ουσίες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Και για το γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθούν άλλες φωσφορούχες ή φωσφατούχες ουσίες. Ένας από τους λόγους είναι υπό διαφορετική σύνθεση με χαμηλή συμπίκνωση η αξιολόγηση που έγινε από την ΣΕΡ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα μπορούσαν να αποτελούν ένα κίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον. Εξού και θεωρήσαμε ότι ήταν αναγκαίο να αποφύγουμε την ε, ε, αύξηση τέτοιου, ε, της χρήσης τέτοιου είδους ουσιών, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθετικές ουσίες. Ο κύριος Ταραμπέλα ζήτησε να δούμε αν θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε διαφορετικά την διατύπωση αυτή αντί να έχουμε ένα ανώτατο όριο για παράδειγμα ε, γραμμαρίων αναδόση. Πρέπει να πω ότι μια παρατήρηση ήταν αυτή που έγινε σε μας μετά την ε, υποβολή της πρότασής μας. Καθορίζοντας ένα ποσοστό θα μπορούσε να ε, διευκολύνει την προσέγγιση αυτή. Όπως ανέλαβε, ανέφερε ο κύριος Ταραμπέλα, δεν είδαμε αύξηση αλλά το αντίθετο και αληθεύει το ότι αν παραμείνουμε σε ένα ε, τέτοιο ποσοστό θα μπορούσε ίσως ε, να δημιουργήσει κάποιο ε, εμπόδιο στη συνέχεια είμαστε πρόθυμοι να δούμε πώς θα μπορέσει να προσεγγιστεί αυτή η δυνατότητα. Αν θα μπορούσε η προσέγγιση του κυρίου Ταραμπέλα να υιοθετηθεί ή μια άλλη ε, διαφορετική προσέγγιση. Έχουμε την εντύπωση ότι το 0,5% στις ε, σημερινές ας το πω, συμπυκνώσεις θα ήταν το 0,5% ε, ως γραμμάρια ως όριο. Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και το είδος των ε, ρήπων. Και αν δει κανείς ε, ε, τις οδηγίες στο πακέτο υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες χρήσης διαφορετικής ποσότητας αυτών των αντιρρυπαντικών δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή όμως να αντικατασταθούν πανευρωπαϊκά αυτές οι ουσίες. Η ουσία, η είναι ότι στην Σουηδία μπορεί να αντικατασταθεί ευκολότερα αυτή ε, από τις άλλες ε, χώρες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, η ε, χωρίς φωσφατούχα χρήση στα, στις μηχανές που ε, πλένουν τα ε, πιάτα δεν θα ήταν δυνατόν να έχουν την ίδια ε, θετική απόδοση. Γι' αυτό δεν θα μπορούσα αμέσω ε, να πω ότι θα το κάναμε άμεσα. Είναι πρώιμη αυτή η φάση τώρα να ληφθεί μια τέτοια απόφαση. Πρέπει να αναμείνουμε μελέτη επιπτώσεων. Αν γίνει η αναθεώρηση σε πρώιμη φάση θα ε, ήταν αντιπαραγωγική. Γι' αυτό προτείναμε κατά τα τέλη του 2014 να γίνει αυτό. Και τέλος εξίσου σημαντικό η πρόταση του κυρίου Ταραμπέλα να υπάρξουν και άλλες ε, οδηγίες στην συσκευασία για την χρήση αυτών των ουσιών λαμβάνοντας υπόψη αυτή αυτές τις ε, προτάσεις ήδη εφαρμόζονται στις ε, συσκευασίες ε, των <clears throat> ουσιών αυτών με την εθελοντική αυτή προσέγγιση των εταιριών που έχουν δείξει μια θετική προσέγγιση του προβλήματος σε σχέση με την αντιμετώπιση ως νομική υποχρέωση. Θα θέλαμε φυσικά στην αναθεώρηση για τα στοιχεία αυτά να δούμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο τι μπορεί να γίνει σε σχέση με τα όσα ανέφερε ο κύριος Ταραμπέλα για τον, την αξιολόγηση κύκλου ζωής και σίγουρα θα εξετάσουμε τις εναλλακτικέ δυνατότητες και τις επιπτώσεις και στην υγεία και στο περιβάλλον αλλά και την, ε, το εφικτό του εγχειρήματο από πλευράς ε, τεχνικής ε, τεχνολογίας. Σας ευχαριστώ. Thank you Ευχαριστώ. Νομίζω ότι τα σημείωσε αυτά που είπατε ο κύριο Ταραμπέλα. Τώρα για το χρονοδιάγραμμα, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Ταραμπέλα για να συνοψίσει. Ε, 24 Μαρτίου, ε, 5η, 23 Απριλίου, α, Συγγνώμη, 15 Ιουνίου θα ψηφίσει η 23 απριλιου συγγνωμη Αρμόδια η καθηγητη αρμοδια επιτροπη και θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Ε, Πολύς χρόνος, δίνουμε, ε, πρώτος χρόνος δίνεται, αλλά δεν πειράζει. Κύριε Ταραμπέρα, θέλετε να σχολιάσετε αυτά που ακούσατε ή να πείτε οτιδήποτε άλλο πολύ σύντομα, γιατί υπενθυμίσατε τις, χρονο... τις ημερομηνίες. Ευχαριστώ τους ε, συναδέλφους για την ε, συνεργασία και επαναλαμβάνω ότι με, τη βοήθη... με την... εγώ και η βοηθός μου θα είμαστε στη διάθεσή σας για να εξετάσουμε τις τροπολογίες. Ευχαριστώ για τις καλές προθέσεις και για την καλή συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την ε, Κομισιόν. Ο κύριος Μπένες είναι ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Ζητώ συγγνώμη που ξέχασα το όνομά του. Πάμε τώρα στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Πριν κάνουμε, ακούσουμε μια σημαντική παρουσίαση για το σύστημα ενημέρωση για την εσωτερική αφορά ε, θα ήθελα να παραμείνατε και να την ακούσετε, γιατί θα ακούσετε ενδιαφέρουσε πληροφορίε για το πώ λειτουργεί αυτό το σύστημα. Μα ενδιαφέρει πάρα πολύ εμά ε, ο, ο ΣΥΜΚΟ. Ο κύριος Δεκάμπος είναι ο υπεύθυνο ε, για αυτή την ε, έκθεση. Αντικαθιστά τον κύριο Γκρέχ. Έχουμε τα συστήματα εγγύσεων των ε, ασφαλίσεων. Ο κύριος Κορέντε Κάμπος ε, θα παρουσιάσει την έκθεση αυτή εκ μέρους του κυρίου Γκρέχ. Σας ευχαριστώ εξ ονόματος του Λουί Γκρέχ. Θα προσπαθήσω να μην υπάρχουν ε, δίπλο επικαλύψεις ε, με θέματα της Επιτροπής ΕΚΟΝ και να ληφθούν μόνο υπόψη τα θέματα προστασίας καταναλωτών ιδιαίτερα. Το θέμα είναι ότι ο μηχανισμός ε, αποζημιώσεων για τις απώλειες ε, των καταναλωτών σε σχέση με ε, πτωχεύσεις ή χρεοκοπίες. Η ομάδα αυτή των καταναλωτών είναι από τις πιο ευάλωτες και σε σχέση και με την πρόσφατη κρίση, οικονομική κρίση, είδαμε ποιε είναι οι επιπτώσεις ε, για τους ε, καταναλωτές ε, και την εμπιστοσύνη όσον αφορά τον χρηματοοικονομικό τομέα. Πρέπει να διασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη σε σχέση με τους καταναλωτές για τις εγγυήσει των καταθέσεών τους. Δράση πρέπει να αναλυφθεί για να μπορέσουν να προστατευτούν αυτά τα συμφέροντα των καταναλωτών. Η αρχή είναι ότι πρέπει να μπορέσει να λειτουργήσει ένα επίπεδο ασφάλειας με ένα ε, σχέδιο εγγυήσεων των καταθέσεων. Και δυστυχώς σε σχέση με την προστασία των καταναλωτών, η ασφαλιστική αυτή συνιστόσα, το σκέλος ε, της, ασφα... της ασφάλειας ε, χωλαίνει. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι διαφορετικά συστήματα λειτουργούν σε διαφορετικά κράτη-μέλη και δημιουργούν άνισα επίπεδα προστασίας. Και αυτό παρεμποδίζει την λειτουργία διασυνοριακά της προστασίας ε, και την δημιουργία ενός ισότιμου πεδίου εμπλοκής. Ο εισηγητής θεωρεί ότι η εισαγωγή ε, συστημάτων ασφάλειας, εσφάλισης και εχέγγυων θα δώσει την δυνατότητα να ανακάμψει η εμπιστοσύνη των ε, καταναλωτών. Θεωρεί ότι ο εισηγητής ότι η πιο ρεαλιστική προσέγγιση αυτή τη στιγμή είναι η δημιουργία ενός νομικού, νομικά δεσμευτικού πλαισίου για αυτές τις εγγυήσεις που θα είναι επαρκής ε, ε, αντιστάθμιση ώστε να μπορέσουν να αντισταθμιστούν ε, οποιασδήποτε απώλειες. Δεν θα πρέπει ωστόσο να υπονομευθεί η προστασία που διασφαλίζεται από τα κράτη-μέλη ήδη σήμερα. Γι' αυτό το πλαίσιο της IGS θα πρέπει, όπως θεωρεί ο εισηγητής, να βασίζεται στο, στην αρχή της του ελάχιστου εναρμονισμού. Το μελλοντικό ε, σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί με τρόπο ώστε να μπορεί να συνάδει με τα συστήματα εποπτείας. Ο εισηγητής ε, εν τέλει αντιμετωπίζει θέματα ενημέρωσης και πληροφόρησης την ε, διαχείριση και διακυβέρνηση και αναφέρει ότι η πληροφόρηση και ενημέρωση πρέπει να είναι διαθέσιμη στους καταναλωτές σε περίπτωση προβλημάτων ε, σε σχέση με μια εταιρεία πιστεύει ότι μία ενιαία θηρίδα για όλες τις δυνατότητες αυτές ε, θα πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει, πράγμα το οποίο θα, αυξήσει την διαφάνεια και, την, ε, τα ειχέγγυα για την βάση του IGS και για ένα επαρκές πλαίσιο αντιστάθμισης θα πρέπει να συνοδεύεται από μια μεταβατική, επαρκή μεταβατική περίοδο και σε σχέση και με τις ε, ε, απαιτήσεις ε, για την διακυβέρνηση που θα πρέπει να είναι αποτελεσματική, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι το IGS θα διασφαλίζει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και θα διασφαλίζει αποτελεσματική εποπτεία και συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών εποπτείας και των ευρωπαϊκών αρχών εποπτείας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Uh, Σας ευχαριστώ <clears throat> και εγώ είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η έκθεση του κ. Γκρέκ που παρουσιάσατε. Η προστασία των καταναλωτών είναι πολύ σημαντική για την Επιτροπή μας. Θα ακούσουμε τώρα τις παρεμβάσεις των σκιωδών εισηγητών, Σβάμπ, Κρόιτσμαν, υποθέτω, θα δικαταστεί ο κ. Σμιτ. Κύριε Ρίουλε, Φόξ επίσης είναι παρόν. Ας ακούσουμε τώρα τους σκιώδη συγητές. Λίντε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κ. Μακρέζη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κ. Φάμπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πρώτα τον κύριο Κορέα Δεκάμπος. Ευχαριστώ βέβαια και τον ίδιο τον εισηγητή Λουί Γκρέκ με τον οποίο συναντηθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα για να συζητήσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά της, ομα... της έκθεσης ούτε στις μισές ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή χώρες μέλη ή και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου δεν υπάρχουν συστήματα εγγύσεων των ασφαλιστικών των, ασφαλίσεων και ποικίλουν και πολλοί και σε ό,τι αφορά το ποσόν και σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή. Γι' αυτό και η ομάδα μου και εγώ ως κοιόδη συγητής εκφράζουμε ικανοποίηση για την πρόθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει ενίο πλαίσιο για τα συστήματα αυτά με ελάχιστε προδιαγραφέ για όλε τι χώρε μέλη. Θεωρούμε ότι αυτό θα τονώσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στον κλάδο των ασφαλίσεων αλλά και την ίδια την ενιαία αγορά διότι θεσπίζουμε ίσους όρους ανταγωνισμού όλων των επιχειρήσεων, καθώς επίσης και διαφάνεια. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντάσσεται μετά από την ψήφιση της οδηγίας Solvency 2 σε μια σειρά μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν τον στόχο να αντιμετωπίσουν τις αδυσμενεί συνέπειες της παγκόσμιας κρίσης και μακροπρόθεσμα να επιτρέψουν στις ασφαλιστικές επιχείρησεις να σταθεροποιηθούν στην ε, νομισματική ένωση. Αλλά και να ολοκληρώσουν βέβαια την αγορά ασφαλίσεων. Καταρχήν, λοιπόν, συμφωνώ σε πολλά σημεία με την έκθεση του κύριου Λουίς Κρέσ, αλλά καλύτερα να έρθω να μιλήσω για τα ζητήματα εκείνα όπου ίσως θα καταθέσω τροπολογίες, διότι θεωρώ ότι χρειάζεται η έκθεση κάπου κάποιες βελτιώσεις. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό τέτοια συστήματα ασφαλίσεων όπως τα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να παρεμβαίνουν όταν δεν υπάρχουν πλέον άλλοι μηχανισμοί προστασίας, όπως για παράδειγμα οι ρυθμίσεις της οδηγίας Solvency 2. Διότι θεωρώ ότι σε ένα τομέα που μέχρι τώρα δεν έχουμε απολύτως καμία ρύθμιση, θα πρέπει πρώτα να απαιτήσουμε την εφαρμογή των ήδη φυσταμένων ρυθμίσεων και μετά να προχωρήσουμε πέραν αυτών. Δεύτερο, ένα άλλο θέμα που πρέπει να τεθεί είναι το, ένα ενδεχόμενο ασφαλιστικό όριο, δηλαδή να γνωρίζει ο καταναλωτής ποιον κίνδυνο αναλαμβάνει ο ίδιος κατά περίπτωση και ποιος κίνδυνος καλύπτεται από νομοθετική ρύθμιση. Θα πρέπει να είναι μια λύση που να εξασφαλίζει την εμπιστοσύνη του καταναλωτή προς την ασφαλιστική εταιρεία, αλλά ταυτόχρονα και ευνοϊκά ασφάλιστρα. Νομίζω ότι εδώ μπορούμε να συζητήσουμε ορισμένα πράγματα με τον κύριο Λουίς Κρέσ. Πάντως τον ευχαριστώ για τη συνεργασία του και ε, αναμένω με ενδιαφέρον την συνέχισή της. Ευχαριστώ κύριε Σφάπ. Εσείς κύριε Κρότσμαν. Στα αγγλικά σας ευχαριστώ. Εξ ονόματος του φίλου μου Όλε Σμιτ, ευχαριστώ τον κύριο Γκρέκ για την συνεργασία. Όλε Σμιτ θεωρεί ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η προστασία των καταναλωτών κυρίως για πολίτες οι οποίες έχουν διαμεθοριακές επενδύσεις και να έχουν ε, ίσο επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης όλες τις χώρες μέλη. Και βέβαια να εξασφαλιστεί και ο ανταγωνισμός σε ίσους όρους ε, στους ασφαλιστικούς κλάδους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και με εναρμόνιση των εθνικών ενόμων τάξεων στο θέμα αυτό. Να δημιουργηθεί μια ε, ισχυρότερη εννέα αγορά. Η ομάδα των φιλελευθέρων υποστηρίζει το μεγαλύτερο μέρος της εκθέσεως του κ. Γκρέσ και υποστηρίζει και στοιχεία όπως για παράδειγμα ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ελάχιστη εναρμόνιση και επίσης η αρχή της ε, χώρας μέλους της έδρας. Για περιπτώσεις πτωχεύσεων μέσα στον ασφαλιστικό κλάδο θα πρέπει να χρηματοδοτούνται εκ των υστέρων και όχι εκ των προτέρων τα συστήματα αυτά θα πρέπει να έχουν αμοιβαίο ασφαλιστικό χαρακτήρα και να μην είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο που τελικά να έχει την έννοια φόρου. Η χρηματοδότηση ex post θα καλύπτεται από τον καταναλωτή, αλλά χωρίς, γιατί στην περίπτωση αυτή θα καλύπτει τον καταναλωτή, χωρίς καμία πρόσθετη ωφέλεια για αυτόν. Τώρα, για τα άρθρα 4, 6 και 8, ο κύριος Σμιτ έχει ε, ορισμένες εμφορίες σχετικά με την κάλυψη σε ορισμένες δραστηριότητες που επεκτείνει το πεδίο των καλύψεων για να μπουν και σε περιπτώσεις αξιογράφων, αλλά ταυτόχρονα οι ασφαλιστικές εταιρείε σήμερα είναι ήδη υπεύθυνε για την συμπεριφορά των υπαλλήλων τους. Δεύτερο, ήδη οι διαμεσολαβητές έχουν, μεσολαβούντες δηλαδή, έχουν υποχρεώσει ήδη να είναι ασφαλιστικά καλυμμένοι. Και αυτό πρέπει να καλύπτει, όπως είπα, και τους ε, μεσάζοντες. Και τέλος, οι περιπτώσει απάτη υπάγονται στο ποινικό δίκαιο και δεν είναι θέμα να καλύπτονται εδώ. Στην παράγραφο 6 αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί, δεν προσφέρει καμία ωφέλεια στον καταναλωτή. Ο κ. Σμιτ είναι επιφυλακτικό διότι στην πράξη θα είναι αδύνατον οι, αρχέ εποπτεία να εξετάσουν περιπτώσεις πτωχεύσεων εάν ορισμένοι πελάτε απαιτούν χρηματικές αποζημιώσεις και σύμφωνα με την Σουηδική Εποπτική Αρχή των Ασφαλίσεων με την οποία διαβουλεύθηκε ο κύριος Σμιτ αυτό που κάνουν αυτοί είναι να προσπαθούν να πολλούν ολόκληρα ασφαλιστικά χορτοφυλάκια σε άλλες ασφαλιστικές ε, επιχειρήσεις σε περίπτωση πτωχεύσεως. Και αυτό είναι καλύτερα και για τον καταναλωτή. Το άρθρο 8 προκαλεί προβλήματα για μικρές αγορές όπου υπάρχουν δηλαδή λίγες μεγάλες επιχειρήσεις. Στις περιπτώσεις αυτές το ρόλο εγγυητού πρέπει να παίζει το κράτο, Εφόσον πτωχεύσει μία από τι μεγάλε αυτέ ασφαλιστικέ εταιρείε, οι μικρότερε ασφαλιστικέ εταιρείε δεν θα μπορούν να πληρώσουν τα ασφάλιστρα που θα απαιτεί το Ταμείο. Στι περιπτώσει αυτέ, μάλλον θα πρέπει να παρεμβαίνει το κράτο και να καλύπτει την ζημία. Αυτά λέει ο κ. Σμιτ, ο οποίο εκφράζει τη λύπη του για την απουσία του, αλλά θα συνεργαστεί με τον εισηγητή και θα δούμε πώς θα προχωρήσει η υπόθεση αυτή. Ευχαριστώ κύριε Κρότσμαν. Βεβαίως είναι σημαντική η γνώση του κυρίου Σμιτ και παρακαλώ να το μεταβιβάσετε σε ευχαριστίες μας. Τώρα ας μιλήσει ο κύριος Φόξ πριν από την κυρία Ρούλε διότι ECR τώρα και πράσινη, αφού η ECR απέκτησε, η συντηρητική δηλαδή απέκτησαν ένα μέρος παραπάνω προ δύο εβδομάδων, είναι ισοδύναμη σε αριθμό. Μάλιστα, ευχαριστώ. Γι' αυτό λέμε και εμείς του be 6 and sevens. Ορισμένες συντεχνίες δηλαδή είχαν ε, ισοδυναμία στην, ε, στο σίδι του Λονδίνου και γι' αυτό ε, μπορούσαν να λαμβάνουν το λόγο πότε η μία και πότε η άλλη πριν. Ευχαριστώ τον κύριο Γκρέσ που ασχολείται με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις αγορές ασφαλίσεων. Εμείς διαφέρουμε με την άποψη του κυρίου Γκρέσ. Εμείς υποστηρίζουμε μια ελάχιστη εναρμόνιση αλλά και την αρχή της ε, χώρας της έδρας. Να μην λησμονούμε ότι η ασφαλιστική αγορά είναι πολύ διαφορετική από την τραπεζική. Εάν πτωχεύσει μια ασφαλιστική εταιρεία, δεν θα συμβούν τα ίδια πράγματα όπως εάν πτωχεύσει μια τράπεζα. Δεν θα τρέξουν όλοι δηλαδή να ε, πάρουν τα χρήματα τους πίσω. Το ζήτημα είναι και πώς χρηματοδοτούνται οι ασφαλιστικές εταιρείε. Γι' αυτό πρέπει να συζητηθούν και τα επίπεδα χρηματοδοτήσεων πριν να επιβάλλουμε όρια ή επίπεδα μάλλον. Και όπως λέει και ο κύριος Κρότσμαν, δεν νομίζουμε ότι πρέπει να υπάρξει ένα ταμείο εξάντε. ante. Μπορεί να γίνει χρηματοδότηση ex post. Συμφωνούμε με την ομάδα των φιλελευθέρων επίσης ότι δεν θα πρέπει η κάλυψη αυτή να καλύπτει και περιπτώσεις απάτης, διότι τότε θα πρέπει οι καταναλωτές να στρέφονται κατά της επιχείρησης. Μόνο όπου ο ασφαλιστής επτόχευσε. Κύριε Πρόεδρε, εμείς συνεργαστήκαμε με τον κύριο Κρέσκο και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και στο μέλλον. Μάλιστα, σας ευχαριστώ κύριε Φόξ. Η κυρία Ρούλε ολοκληρώνει το γύρο αυτό της, ερωτήσεως, Θα είμαι σύντομη και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γκρέκα και να ευχαριστήσω τον κύριο Ντεκάμπος για την παρουσίαση των απόψεων του συντάκτη και της έκθεσης. Θέλω να πω ότι μου έκανα να προβληματιστώ κάποιες παρατηρήσεις και πρέπει να συζητήσουμε τους κοιόδης αυτά τα θέματα και το θέμα της ε, παραπλάνησης ή απάτης θα πρέπει να μπορεί να ε, ρυθμιστεί. Νομίζω όμως ότι αυτό δεν είναι υποχρεωτικό να ενταχθεί εδώ. Πρέπει όμως να συζητήσουμε αυτά τα πράγματα. Θέλω να δώσω συνέχεια σε κάτι το οποίο στην αρχή αναφέρθηκε και μετά αμελήθηκε. Ότι υπάρχει μεγάλος ε, κίνδυνος με την διαφάνεια των, της επικινδυνότητας και των επισφαλιών και είδαμε ότι το ίδιο το πρόβλημα υφίσταται ότι δεν υπήρχε σαφήνεια για τους ε, κινδύνους. Πώς δηλαδή θα μπορούσαν ε, να, έχουν επιπτώσεις όσον αφορά τα ε, έσοδα, τα, τα χρήματα των επενδυτών. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα εξετάσουμε περισσότερο νομίζω. Ευχαριστώ. Well, thank ευχαριστώ. Στην γενική γραμμή που παρακολουθούμε είναι η γραμμή που έχουμε θεσμοθετήσει σε αυτή την ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή όσον αφορά και την σαφήνεια των στοιχείων των πληροφοριακών στοιχείων για τους καταναλωτές, κάτι που θα έχει πολύ μεγάλη σημασία και είναι κάτι που θα ληφθεί υπόψη. Λοιπόν, με χαρά μπορώ να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει στη συνέχεια για το λευκό βιβλίο και ο κύριος ε, Μαρκέση θα είναι εκείνος ο οποίος ε, θα παρουσιάσει τις απόψεις αυτές. Παρακαλώ. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Κοινοβουλευτικής σα Επιτροπής για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε κάποια λίγα θέματα που πιστεύω ότι βρίσκονται στο επίκεντρο, στον πυρήνα των συζητήσεων, όχι μόνο σε αυτήν την Κοινοβουλευτική Επιτροπή, αλλά επίσης στην ε, Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το θέμα των κονδυλίων. Με χαρά άκουσα ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπάρχει εξ χρηματοδότηση για το IGS. Θα ήθελα να επαναλάβω όμως ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επ' αυτού. Αν όμως έχουμε μόνο εξ post χρηματοδότηση θα υπάρχουν διτά προβλήματα. Το ε, πρώτο είναι ο κίνδυνος, η επισφάλεια, επειδή δεν θα συνεισφέρει η ασφάλιση στα κονδύλια του Ταμείου. Αυτό ακριβώς ε, δεν θέλουμε να δημιουργηθεί ως κίνδυνος. Αν έχουμε από την άλλη πλευρά μόνο αποκλειστικά εξπόστ πιθανότατα καθώς ε, θα συσχετίζονται τα κονδύλια τα ασφαλιστικά, στο τέλος τέλος θα καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου θα ζητηθεί από τις επιχειρήσεις που θα βρίσκονται υποπίεση λόγω της κυκλικής εξέλιξης των πραγμάτων που συγκυριακά μπορεί να βαίνει ε, αρνητικά, να πληρώσουν ακριβώς τα χρήματα αυτά στην εσφαλμένη χρονική συγκυρία υπέρ της κυκλικής αυτής ε, ε, διαμόρφωσης των πραγμάτων η εξπός χρηματοδότηση. Γι' αυτό πιστεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η σωστή μορφή χρηματοδότησης είναι η εξάντε, εκ προημίου δηλαδή ε, προκαταβολική διασφάλιση των κονδυλίων στην ε, χρηματοδότηση. Και για να μην ε, υπερβάλλουμε κατά την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, θα ήθελα να αναφερθώ στο γεγονός ότι η μελέτη επιπτώσεων στο Λευκό Βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξειδικευμένα ρητά λαμβάνει υπόψη την κατάσταση σε σχέση με τους κινδύνους ε, τις επισφάλειας που δημιουργούνται σε σχέση με το Solvency 2, όταν αυτό θα έχει αρχίσει να λειτουργεί. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να προδικάζεται ή να αμελείται το γεγονός ότι είναι σημαντική η ε, χρηματοοικονομική σταθερότητα μέσα στο πλαίσιο του Solvency 2 ως τεκμήριο του πόσο καλό μπορεί να είναι ένα σύστημα. Δεν μπορεί να υπάρξει ένα μηδενικό επίπεδο κινδύνων. Θα υπάρχει πάντα κάποιος κίνδυνος και κάποια επισφάλεια και η δυνατότητα για κάποια απρόβλεπτα ε, γεγονότα οι ε, επόπτες, οι επιθεωρητές να μην μπορούν να προβλέψουν τα πάντα σε σχέση με μια ασφαλιστική εταιρεία. Γι' αυτό το IGS είναι σημαντικό για να διασφαλίσουμε ότι θα δημιουργηθεί εμπιστοσύνη από πλευράς των ε, καταναλωτών και επενδυτών που δεν θα μπορεί να σβήσει ή να εξαλειφθεί. Και το βρήκα ενδιαφέρον την αναφορά που έγινε σε σχέση με το πρόβλημα εκείνων των αγορών που η ασφαλιστική αγορά επικεντρώνεται σε αυτά τα πλαίσια. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί για μαγικές λύσεις. Πρέπει να καθορίσουμε, να καταλήξουμε στη σωστή ισορροπία μεταξύ προστασίας των καταναλωτών και όχι υπερβολικής συσσόρευσης κονδυλίων που θα απέβαινε αρνητική για τις επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα όταν υπάρχει ιδιαίτερο επίπεδο συμπίκνωσης που δημιουργεί μεγαλύτερες, ε, μεγαλύτερους κινδύνους. Όσο μεγαλύτερος ο όγκος, τόσο μεγαλύτερη κίνδυνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να λάβει υπόψη αυτά στη μελέτη επιπτώσεων από πλευρά τη. Και ιδιαίτερα έχουμε εισαγάγει την δυνατότητα υπολογισμών και στάθμισης από πλευράς IGS ανάλογα με το επίπεδο συμπίκνωσης, ε, επικέντρωσης που υπάρχει στις διάφορες αγορές. Αυτό δεν, δεν σημαίνει ότι οποτεδήποτε, σε οποιαδήποτε περίπτωση, οποιαδήποτε επισφάλεια, οποιοδήποτε μεγέθους μπορεί να απορροφηθεί από το IGS. Αλλά γίνεται προσπάθεια να ανταποκριθούμε σε αυτόν τον αυξημένο κίνδυνο όταν υπάρχει συμπίκνωση στην αγορά. Τούτων λεχθέντων θα έπρεπε να αναφέρουμε ότι δεν πρέπει μόνο αποκλειστικά να εξετάζεται το IGS σαν μόνη λύση να αποφευθούν ε, προβλήματα. Διότι σαφώς ε, αντιδρούν περισσότερο οι επιθεωρητές, οι επόπτες ε, στον μεγαλύτερο όγκο όταν ε, ε, σημειώνεται συμπίκνωση. Ιδιαίτερα θεωρώ πολύ σημαντικά τα μαθήματα τα οποία μπορούμε να συναγάγουμε από τέτοια προβλήματα όταν ζητείτε να υπάρξει ρευστοποίηση και να υπάρξει μετάβαση σε ένα άλλο ασφαλιστικό πλαίσιο. Θα πρέπει πάρα πολύ καλά να αξιολογήσουμε αυτή την κατάσταση. Διότι αυτό που είναι σημαντικό, όπως είπα, είναι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο, ώστε από κοινού με τους ε, επόπτες, τις εποπτικές αρχές να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Πρέπει να είναι ένας πρακτικός τρόπος λειτουργίας ε, και αντιμετώπισης των πραγμάτων για να είμαστε αποτελεσματικοί. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μας αρέσει αυτή η προσέγγιση της Κομισιόν μέσω της ε, Λευκή Βίβλου. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Καλό θα ήταν να συζητήσουμε στα πλαίσια του, της διαδικασίας του Εθνομοθετήν το χρονοδιάγραμμα. Και μετά ο κ. Κορέι Ντεκάμπος θα ξαναπάρει τον λόγο. Για την κατάθεση των τροπολογιών 24 Μαρτίου, θα εξετάσουμε τις τροπολογίες στις 12 Απριλίου, θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή στις 13 Απριλίου και θα ψηφίσουμε στην ε, Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων στις 2 Μαΐου. Ε, είναι αρκετά πιεσμένο το χρονοδιάγραμμα και θα ψηφίσουμε και στην Ολομέλεια του Ιουνίου. Νομίζω ότι ελέγχουμε το θέμα ε, και εφόσον το ελέγχουμε νομίζω θα καταφέρουμε να διεκπαιρεώσουμε τις τροπολογίες, την έκθεση, να κάνουμε τέλο όλη τη διαδικασία. Ο κ. Κορέα Ντεκάμπος θέλει να πει κάτι, να συνοψίσει. Θέλω να ευχαριστήσω απλώς τους συναδέλφους, λέει ο κ. Κορέντε Κάμπος. Σημείωσα τις παρατηρήσεις. Ε, επί της ουσίας δεν είμαι έτοιμος να απαντήσω. Όλα τα σχόλιά σας θα τα παραπέμψω στον συνάδελφο που είναι αρμόδιος, που είναι υπεύθυνος για την έκθεση, στον κύριο Λουίς Γκρέχ. Σας ευχαριστώ και τώρα περνάμε στο τελευταίο σημείο για σήμερα, που είναι η παρουσίαση από την Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς για το σύστημα αυτό ενημέρωσης για την εσωτερική αγορά. Ε, όπως ξέρετε, είναι μια σημαντική προσπάθεια, ένα σημαντικό σύστημα για να διευκολύνουμε τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Καλύπτει πολλά θέματα. Ε, χαίρομαι όταν έχετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μας παρουσιάζει διάφορα θέματα. Έχουμε και ένα αντίγραφο την έκθεση που θα μας παρουσιαστεί. Θα ήθελα τακτικά να έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ή μάλλον η κυρία Μαριάν ε, Γκράμερ, η οποία είναι υπεύθυνη, είναι τακτική στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα τώρα να μας κάνει την παρουσίασή της και συνεχεία να απαντήσει στις ερωτήσεις των ε, βουλευτών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για το πού βρισκόμαστε με αυτό το σύστημα ενημέρωσης για την εσωτερική αγορά και πού θέλουμε να φτάσουμε. Γιατί σας κάνω αυτή την παρουσίαση. Η Κομισιόν υιοθέτησε μία ανακοίνωση για την επέκταση και την ανάπτυξη αυτού του συστήματος ενημέρωσης. Υπάρχει και η ετήσια έκθεση με τα στοιχεία για το πώς λειτουργήσε αυτό το σύστημα το 2010. Επίσης, αυτή η παρουσίαση είναι σημαντική για να προετοιμάσει το έδαφος για ένα σχέδιο κανονισμού που θα σας υποβάλουμε ε, στις αργότερα, μέσα στο 2011. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω, τι είναι αυτό το σύστημα ενημέρωσης. Είναι καταρχάς μια εφαρμογή που βασίζεται στο ίντερνετ, δηλαδή δεν χρειάζεται κανένα ιδιαίτερο λογισμικό ή κανένα ιδιαίτερο εξοπλισμό. Είναι ένα εργαλείο που αναπτύξαμε με τα κράτη-μέλη, ε, ούτω ώστε να συνδέονται οι εθνικές αρχές σε όλα τα επίπεδα σε τοπικό ε, περιφερειακό και εθνικό. Δημιουργήθηκε αυτό το σύστημα για να καλύψουμε ένα μεγάλο χάσμα που υπάρχει από τις ε, εθνικές αρχές όταν ψάχνουν το σωστό ομόλογό τους. Έχουμε πάνω πάνω από 6.000 διαφορετικές αρχές σε όλα τα κρατη που είναι καταγεγραμμένες σε αυτό το σύστημα και είναι πολύ σημαντικό για τα κράτη-μέλη να έχουν ένα εργαλείο για να βρουν το σωστό συνομιλητή, το σωστό ομόλογο σε άλλο κρατός μέλος για να επικοινωνήσουν. Ε, το σύστημα αυτό επιτρέπει σε αυτές τις αρχές να ανταλλάσσουν πληροφορίες με ασφαλή τρόπο. Ε, είναι φιλικό ε, σε ό,τι αφορά την προστασία της βάσης δεδομένων. Έχουμε διάφορους κανόνες για την προστασία ενσωματωμένου στο σύστημα, ούτως ώστε η πληροφορία που έχει και προσωπικά δεδομένα συχνά να ανταλλάσσεται με ασφαλή τρόπο μεταξύ των διαφόρων αρχών και πολύ σημαντικό στοιχείο του συστήματος αυτού είναι ότι λειτουργεί σε όλες τις ε, ενωσιακές γλώσσες. Υπάρχουν ε, διάφορες ερωτήσεις και απαντήσεις που έχουν ήδη μεταφραστεί και που μπορεί να χρησιμοποιήσουν οι αρχές. Δηλαδή, αν παραδείγματο χάρη μια λιθουανική αρχή έχει μια ερώτηση προς μια πολωνική αρχή, ας πούμε, τότε οι λιθουανικές αρχές θα κάνουν κλικ στο, στο ερώτημα στα λιθουανικά το στέλνουν στις πολωνικές αρχές που το διαβάζουν στα πολωνικά, επιλέγουν την απάντηση στα πολωνικά, ε, το στέλνουν μέσω του συστήματος ε, και το διαβάζουν οι Λιθουανοί στα λιθουανικά. Είναι σημαντικό λοιπόν στοιχείο αυτό και καλύπτονται έτσι διάφορα χάσματα ε, και αυτό το χάσμα το γλωσσικό. Τώρα, διάφορα νούμερα. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή από το 2009, χρησιμοποιούμε αυτό το σύστημα ε, για τις επαγγελματικές δεξιότητες και το 2010 για την ε, οδηγία για τις υπηρεσίες. Για αυτούς τους δύο τομείς, όπως σας είπα, πάνω από 6.000 ε, φορείς και δημόσιες αρχές είναι καταγεγραμμένες. Κάποια κράτη-μέλη έχουν τόσο αποκεντρωμένη προσέγγιση που έχουν καταχωρήσει και όλες, όλες τις τοπικές αρχές, όλη την τοπική αυτοδιοίκηση δηλαδή. Από τις 6.000 αυτές αρχές υπάρχουν πάντο από 11.500 μεμονωμένοι χρήστες καταχωρημένοι στο σύστημα αυτό. Έχουμε 160 περίπου αιτήματα ενημέρωσης το μήνα, κατά μέσο όρο. Είναι σχετικά χαμηλό αυτό το νούμερο, αλλά αυξάνεται πολύ γοργά. Αν κοιτάξετε την ταχύτητα, 58% των αιτήσεων ε, απαντώνται μέσα σε δύο εβδομάδες. Πιστεύουμε ότι είναι αρκετά καλή ταχύτητα, αν λάβετε υπόψη σας ότι αυτές οι ανταλλαγές είναι μεταξύ ε, δημοσίων φορέων που δεν έχουν κοινή γλώσσα, δεν έχουν κοινέ διαδικασίε. Ε, το μόνο που έχουν κοινό είναι η χρήση αυτού του συστήματο, το AMI. Επίση, ε, θέλουμε να δούμε, μελετάμε δηλαδή για να δούμε την ανταπόκριση των χρηστών και αν θεωρούν ότι είναι φιλικό προ το χρήση και τι μπορούμε να κάνουμε για να το βελτιώσουμε αυτό. Το 92% των χρηστών μα απαντούν ότι το βρίσκουν εύκολο ε, ως προς τη χρήση το σύστημα αυτό. Τώρα κάποια νούμερα για ό,τι συμβαίνει με το σύστημα. Αυτά είναι οι στατιστικές για αιτήματα για τις επαγγελματικές δεξιότητες και προσόντα. Εδώ βλέπετε ότι ο μέσος όρος των αιτήσεων που, στέλνονται, που στέλνεται είναι περίπου 150 το μήνα. Φυσικά, οι στατιστικές συνοψίζουν διαφορετικά επίπεδα δραστηριότητα σε διάφορα κράτη-μέλη. Και αν κοιτάξουμε Ποιοι στέλνουν κυρίως ε, αιτήματα για πληροφορία ε, στον τομέα των επαγγελματικών προσόντων. Τότε το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία και η Ολλανδία στέλνουν τα περισσότερα αιτήματα για ενημέρωση. Αν δούμε ποιοι παραλαμβάνουν αυτά τα αιτήματα, βλέπουμε ότι η Ρουμανία, η Πολωνία και η Γερμανία είναι αυτοί που παραλαμβάνουν τα περισσότερα ερωτήματα ή αιτήματα, ας πούμε, για απάντηση. Τώρα, Ποια επαγγέλματα καλύπτουν αυτά τα, αυτές οι αιτήσει. Αυτή η γραφική παράσταση σας βλέπει ότι το 1 τρίτο των συνολικών ερωτημάτων αφορούν τους γιατρούς, που είναι πάρα πολύ έτσι, ευκίνητο επάγγελμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερο επάγγελμα είναι οι καθηγητές. Το 1 τρίτο επίσης τις πίτες και το άλλο τρίτο αν κοιτάξετε τουλάχιστον το MI, το σύστημα αυτό, είναι οι νοσοκόμες. Μετά καλύπτουμε και άλλα επαγγέλματα, οδιάτρους, ε, φαρμακοποιούς, ε, χειρουργούς, εκτινίατρους, αρχιτέκτονες, φυσιοθεραπευτές, λογιστές και ΜΕΣ. Έχουμε 35 επαγγέλματα που καλύπτονται και επεκτηνόμαστε για να καλύψουμε όλα τα επαγγέλματα που παρουσιάζουν μεγάλη κινητικότητα. Ένα άλλο νούμερο για το πόσο γρήγορα αυτά τα αιτήματα ε, προς ενημέρωση απαντώνται. Το 43% απαντάτε μέσα σε δύο εβδομάδες, όχι σε μία εβδομάδα. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι φτάνει το 59% και έτσι καλύπτουμε ένα 59% έχουμε τις απαντήσεις μέσα σε δύο εβδομάδες. Καλό αποτέλεσμα είναι αυτό. Αν κοιτάξετε τον δεύτερο τομέα που καλύπτεται από το σύστημα είναι ο τομέας των υπηρεσιών. Εδώ έχουμε άλλη εικόνα. Χρησιμοποιούμε αυτό το σύστημα εδώ και ένα χρόνο για τις υπηρεσίες και από ό,τι βλέπετε από τα νούμερα, έχουμε χαμηλότερα νούμερα εδώ από ότι για τις επαγγελματικές δεξιότητες. αυξάνονται όμως, ε, βλέπετε μια ανάπτυξη το Φεβρουάριο και ελπίζω αυτή η τάση να συνεχιστεί, αλλά ζητάμε από τις αρχές και τους εθνικούς συντονιστές ε, να μας πούν γιατί αναπτύσσεται αργά αυτό το σύστημα στον τομέα των υπηρεσιών. Ορισμένοι από τους λόγους που ανέφεραν ε, είναι ότι προσπαθούμε να πετύχουμε στον τομέα των υπηρεσιών το εξή. Να αλλάξουμε τις διοικητικέ πρακτικές. Οι αρχές εδώ και πολλά χρόνια είχαν ένα συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας και τώρα τους ζητάμε να λειτουργήσουν διαφορετικά. Να μην ζητάνε ας πούμε, πλήρη μετάφραση όλων των εγγράφων και να έρθουν σε επαφή μία αρχή, μία μόνο αρχή για να έρθουν, για να λάβουν ας πούμε, πληροφορίες, παρά να πούν «Α, όχι, δεν τους εμπιστεύομαι και δεν απαντάω». Επομένως, συζητάει αυτό το σύστημα απαιτεί μία αλλαγή της κουλτούρας της διοικητικής πρακτικής. Ορισμένες αρχές μας είπαν ότι δεν καταλαβαίνουν εύκολα ποιε είναι οι νέε υποχρεώσει υπό την οδηγία για τι υπηρεσίε πρέπει να υπάρξει μεγάλη κατάρτιση και μεγάλη αφύπνιση, αν θέλετε, μεγάλη συνειδητοποίηση για το τι είναι αυτό το σύστημα, τόσο ώστε να επιταχυνθεί η χρήση του συστήματο ενημέρωση. Δύο λόγια τώρα για την επέκταση και την ανάπτυξη του συστήματο ενημέρωση. Με βάση τη σημερινή χρήση για το τομέα των υπηρεσιών και των επαγγελματικών δεξιοτήτων, ε, βρίσκουμε το εργαλείο είναι πολύ αποτελεσματικό. Ε, χρήσιμο θα ήταν να επεκτείνουμε το εργαλείο και σε άλλου τομεί πολιτική, ε, το σύστημα είναι ένα γενικό εργαλείο. Δεν χρειάζεται δηλαδή να το χρησιμοποιήσουμε μόνο σε ένα τομέα και να περιοριστούμε. Μπορούμε να το προσαρμόσουμε εύκολα ε, για τις ανάγκες ε, μια άλλη πολιτική. Για να το αποδείξω αυτό, αποδείξει αυτό, στι 5 Μαρτίου το Συμβούλιο αποφάσισε να ξεκινήσει ένα πιλωτικό σχήμα για να το εφαρμόσει στον τομέα της ε, οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων βλέπουμε ότι χωρίς ε, περαιτέρω ανάπτυξη του λογισμικού, μπορεί να λειτουργήσει αυτό το σύστημα για να απαντήσουν, να στέλνουν ερωτήσεις οι αρχές και να λαμβάνουν απαντήσεις στον τομέα της απόσπασης εργαζομένων. Τέταρτος τομέας πολιτικής που θα προσθεθεί στο σύστημα, κυρίως χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί προσθέσατε μια αναφορά ε, στη νέα οδηγία για τα δικαιώματα των ασθενών, σε αυτό μια αναφορά σε αυτό το σύστημα, θα υπάρξει μια επέκταση λοιπόν ε, του συστήματος και στον τομέα αυτής της οδηγίας για τα δικαιώματα των ασθενών. Πέρυσι επίσης κοιτάξαμε διάφορες πολιτικές για να δούμε τι δυναμικό υπάρχει για να επεκτείνουμε προς αυτές τις πολιτικές το σύστημα. Βρήκαμε 25 διαφορετικές οδηγίες όπου θεωρητικά θα ήταν χρήσιμο να χρησιμοποιήσουμε το σύστημα αυτό αλλά θα πρέπει να το συζητήσουμε με τις εμπλεκόμενες αρχές και με τους ενδιαφερόμενους. Δύο από τους τομεί που έχουμε εντοπίσει και που μοιάζουν ε, πολλά υποσχόμενοι είναι τομέας του στοιχήματο και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ένας άλλος τομέας πολιτικής είναι ότι θα πρέπει να έχει διάφορες άλλες δυνατότητες λειτουργίας. Παραδείγματο χάρη για τι ε, διαδικασίε κοινοποίησεων. Σε πολλέ οδηγίε τα κράτη-μέλη έχουν υποχρέωση να κοινοποιούν του νέου εθνικού κανόνε ή τι εξαιρέσει και αυτό δεν γίνεται με συστηματικό τρόπο μέχρι στιγμή. Πιστεύουμε ότι μια και έχουμε τόσε πολλέ αρχέ που είναι καταχωρημένε στο σύστημα αυτό ενημέρωση. καλό θα ήταν να του δώσουμε και ένα εργαλείο για την διαδικασία κοινοποίηση. Να χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα δηλαδή για τι κοινοποίησει. Και τέλο, ένα άλλο τομέα επέκταση και ανάπτυξη του συστήματο είναι η διασύνδεσή του με τα υπάρχοντα συστήματα. Υπάρχουν πολλά συστήματα που λειτουργούν, παραδείγματο χάρη η βάση δεδομένων για τα επαγγελματικά προσόντα, που πιστεύουμε ότι καλό θα ήταν να συνδεθεί με το σύστημα αυτό ενημέρωση για την εσωτερική αγορά για να αποφύγουμε τι ε, επικαλύψει. Με δύο λόγια, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να αναπτύξουμε περαιτέρω το σύστημα αυτό, ε, ώστε ε, να είναι μια εργαλειοθήκη για τη διοικητική συνεργασία. Να δώσει στι αρχέ δηλαδή ε, εργαλεία για να ανταλλάσσουν πληροφορίε μεταξύ του, αλλά και μεταξύ των αρχών και τη Κομισιόν παραδείγματο χάρη για αυτέ τι ε, διαδικασίε κοινοποίηση. Τα ωφέλη από την χρήση του συστήματο είναι, είναι προφανή. Είναι πολύ πιο φθηνό να τον απτύξεις περαιτέρω αν δεν χρειάζεται να ξεκινήσει από το μηδέν. Επίση, ένα σύστημα που υπάρχει ήδη και δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε επιπλέον λειτουργίε, ε, λειτουργεί πολύ πιο γρήγορα, αλλά αν το δείτε και από τη σκοπιά του χρήστη, είναι πολύ πιο φιλικό για το χρήστη αν υπάρχουν πολλαπλά, πολλαπλές δυνατότητες που μπορούν να κάνουν ε, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν login σε διαφορετικά συστήματα, να, να θυμούνται ε, διαφορετικά, διαφορετικούς κωδικούς, διαφορετικά password. Είναι χρήσιμο ε, να έχουν ένα εργαλείο ε, για όλες αυτές τις δυνατότητες, για όλη αυτή την διοικητική συνεργασία. Επίσης, ε, είναι υπάρχει και ένα κοινό help desk, υπάρχει ένα μάθημα με πούμε, για τους ειδικού κτλ. Δεν χρειάζεται να το ξανακάνουμε. Επίσης, όσο όση περισσότερη διασύνδεση υπάρχει στο σύστημα, όσοι περισσότεροι είναι συνδεδεμένοι, τόσο καλύτερα λειτουργεί το σύστημα. Τελευταίο σχόλιο, σημαντικό για το σύστημα. Δεν υπάρχει κόστος για τους χρήστες. Είναι κεντρικό το σύστημα και χρηματοδοτείται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Τα κράτη-μέλη δεν χρειάζεται να συνεισφέρουν για την ανάπτυξη και συντήρηση του συστήματος αυτού. Επομένως, ε, δεν υπάρχει πρόβλημα οικονομικό. Το σύστημα αυτό δεν υπάρχει μόνο για τις διοικήσεις. Βοηθάει έμεσα και τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Ε, οδηγεί σε πιο γρήγορες αποκρίσεις, αντιδράσεις μάλλον από τις αρχές, γιατί βρίσκουν πιο εύκολα τις πληροφορίες. Επίσης, μειώνεται σημαντικά η ανάγκη για τη μετάφραση εγγράφων, γιατί τα κράτη-μέλη μπορούν να ζητήσουν απλώς από την αρχή στην άλλη, στην χώρα να τους πει «Α, ισχύει αυτό το έγγραφο», ε, παρά να χρειαστούν, ας πούμε, επικυρωμένο αντίγραφο της μετάφρασης. Τέλος, θα υπάρχουν λιγότερες αρνήσεις ε, και λιγότερες απορρίψεις μάλλον των αιτήσεων λόγω α, έλλειψης κατανόησης ας πούμε. Τα επόμενα βήματα. Θα πρέπει να εντατικοποιήσουμε την προσπάθεια κατάρτισης και συνειδητοποίησης ε, να χρησιμοποιήσουμε τη χρήση, να αυξήσουμε τη χρήση στον τομέα των υπηρεσιών επίσης. Ζητήσαμε επίσης μια μελέτη για την δομή του λογισμικού, τόσο ώστε να ξέρουμε ότι είναι βιώσιμο το σύστημα, ακόμα και όταν το επεκτείνουμε σε πολύ περισσότερες πολιτικές. Ε, μέχρι το 2012 επίσης θα πρέπει να έχουμε ένα σαφές διάγραμμα για την ανάπτυξη και επέκτασή του. Μέχρι στιγμής έχουμε το, εντοπίσει πολλούς τομείς, αλλά θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να δεσμευτούν ότι θέλουν πραγματικά να χρησιμοποιήσουν το σύστημα και θα το χρησιμοποιήσουν, ούτω ώστε να αναπτύξουμε τις νέες λειτουργικότητες που χρειάζεται. Και τέλος, θα, θα υποβάλουμε μία πρόταση για ένα κανονισμό του συστήματος προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο τον Ιούνιο. Ο κανονισμός αυτός θα παγιοποιήσει και θα κωδικοποιήσει τους κανόνες για την προστασία της βάσης δεδομένων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε αποφάσεις και συστάσεις της Κομισιόν. Ε, ο, επόπτης για την προστασία των, της βάσης δεδομένων είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα εργαλείο συναπόφασης που θα προστατεύει αυτούς τους κανόνες και τώρα θα το έχουμε αυτό το εργαλείο, τον κανονισμό. Πέρα από, το, από τους κανόνες προστασίας, θα πρέπει να δούμε και το ρόλο και τις ευθύνες των διαφόρων φορέων και θα πρέπει να έχουμε ένα ευέλικτο εργαλείο που θα μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο ε, και σε άλλες πολιτικές, αλλά με εύκολο τρόπο. Αυτά είναι λοιπόν ήδη σε φάση εξέλιξης. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες έχουμε μια ιστοσελίδα με πολλά έγγραφα. Στην ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε και την ετήσια έκθεση αλλά έχετε λάβει μόλις και το αντίτυπο, στην ε, ανακοίνωση της Κομισιόν για την επέκταση και ανάπτυξη του ε, συστήματος ενημέρωσης θα βρείτε κριτήρια, ε, κατευθυντήριε γραμμές για την στρατηγική επέκτασή του και αν ενδιαφέρεστε πραγματικά θα μπορούσατε να παραστείτε σε μία ενημερωτική έτσι σύνοδο για τους βουλευτές και τους βοηθούς τους κάποια στιγμή το Μάιο ή Ιούνιο. Αν ενδιαφέρεστε για να μάθετε περισσότερα για το πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα ενημέρωσης για την εσωτερική αγορά. Αυτά λοιπόν από μένα, αλλά φυσικά μπορώ να απαντήσω σε οποιασδήποτε ερωτήσεις έχετε. Σας ευχαριστώ Μαριάν για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Και ευχαριστώ που μας ε, συντρέχετε έτσι για την αναθεώρηση για την μελλοντική στρατηγική που αυξάνει η σημασία του θέματος ιδίως με, την νομοθεσία της ενιαίας αγοράς που έχουμε συζητήσει με ορισμένες ε, χώρες μέλη και τα νομοθετήματα αυτά είναι σημαντικά εργαλεία για μας και ορισμένοι από τους τομείς όπου σκοπεύετε να επεκτείνεται το IMI σε αυτούς θα σας υποστηρίξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μαζημένοι θα σα υποστηρίξει παρούσα επιτροπή. Μας μένει λίγος χρόνος, αν θέλετε να θέσετε ερωτήσει. Ο κ. Φαμπ έχει σηκώσει το χέρι, του. Μετά ο κ. Κάμπος, άλλο κανείς, κ. Ριούλε. Α αρχίσουμε με τον κύριο Σφαμπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα, βεβαίω θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το σύστημα ενημέρωση για την έννοια αγορά ήδη έχει προχωρήσει, αποτελεί ένα πολύτιμο μηχανισμό για αμοιβαία ενημέρωση των χωρών μελών και για την υπέρβαση των γλωσσικών προβλημάτων, του γλωσσικού φραγμού δηλαδή, που συχνά και μόνο για το λόγο αυτό δεν είναι σε θέση να συνεργάζονται οι χώρες μέλη. Άρα βοηθεί πολύ εδώ. Αυτό που βρίσκω σωστό είναι ότι προτίθεστε να περιλάβετε και κανονισμό για την προστασία των δεδομένων που είναι και συχνά και δεδομένα που άπτονται της εθνικής κυριαρχίας. Εξετάζω τα όσα περιγράφεται. Όντως η Γερμανία είναι ο πρωταθλητής σε ό,τι αφορά τους φορείς που έχουν εγγραφεί στο IMI. Υπάρχουν και μικρές χώρες με πολλούς φορείς που έχουν εγγραφεί. Νομίζω η Εστονία, η Εστονία έχει εγγράψει πολλές κοινοτικέ και άλλε αρχές, εμένα θα με ενδιέφερε να μου εντοπίσετε πού είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα. Το σύστημα είναι νέο. Οι χώρες μέλη βέβαια θα έχουν και διαφορετικές ερωτήσεις να, να θέτουν στο σύστημα. Ποιε είναι, πού είναι, εντοπίζουν τα προβλήματα. Για παράδειγμα μιλήσατε για τον κλάδο των γιατρών. μήπω μπορείτε να εντοπίσετε λίγο πού βρίσκονται τα προβλήματα τα οποία του τους απασχολούν. και ο κύριος Άτσμαν είναι ε, μπορούμε να δούμε και το θέμα και, και η κυρία Ράπτη. Βλέπω ότι είναι 65 οργανώσεις από την Ελλάδα που έχουν εγγραφεί επαγγελματικού χαρακτήρα. Ε, εσείς κύριε καθηγητάτε Κάμπος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω για αυτή την παρουσίαση που θεωρώ ότι είναι σαφέστατη. Αλλά επίσης έχει και μια ολόκληρη πραγματικότητα που παρουσιάζει που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Οι αμφιβολίες που έχω είναι δύο ή τρεις. Πρώτα απ' όλα η έννοια του National Authorities, εθνικών αρχών at all levels, σε όλα τα επίπεδα. Γνωρίζουμε ότι μπορούν να συμπεριλαμβάνουν επιχειρηματίες επίσης και αναφέρθηκε και στην παρουσίαση. Υποθέτω επίσης ότι μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και συνδικάτα, έτσι δεν είναι. Κατά κάποιο τρόπο Υπάρχει αυτό στο ε, σχέδιο του IMI ένα απόλυτο άνοιγμα για τους απλούς πολίτες ή δεν υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα. Υπάρχει ένας περιορισμός μήπως, ας το πω έτσι, και επιτρέπεται μόνο θεσμικά όργανα να μπορούν να εντάσσονται. Δεύτερο ερώτημα, συσχετίζεται με τον χαρακτήρα ενεργητικού χαρακτήρα ή ενημερωτικού χαρακτήρα φυσικά θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, πάρα πολύ σπουδαία ε, παρέμβαση αυτή η παροχή πληροφοριών. Όμως το πιο ενδιαφέρον θα ήταν και ε, από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μας δώσει ένα παράδειγμα της μεταρρύθμισης της proactive ενεργητικής ε, μεταρρύθμισης όπου μία αρχή θα μπορούσε άμεσα να έρχεται σε επαφή με την αρχή άλλου κράτους μέλους. Αυτό προβλέπεται μέσα στα σχέδια αυτά για το IMI. Είναι απλώς κάτι που θα επικεντρώνεται στην παθητική ενημερωτική ας το πω συνιστόσα στο ενημερωτικό σκέλος. Αυτά ήθελα να πω και θέλω να συγχαρώ για την επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας. Ευχαριστώ. Um, any, other colleagues? Τότε λίγα σχόλια δικά μου. Αναφερθήκατε στη σημασία των γλωσσών και των μεταφράσεων και υπάρχει και ένα σημείωμα σχετικά με αλλαγές στο σύστημα μεταφράσεων. Από, από τις οποίες εξαρτάται το ε, μεταφραστικό σύστημα του IMI. Με ποιον τρόπο το αντιμετωπίζετε. Δεύτερο, σημαντικό ήταν να τεθεί το θέμα της εκπαίδευσης και της πρόθεσης της χρήσης του συστήματος στις χώρες μέλη. Γνωρίζω ότι έχετε συναντήσει συνεργασία κλπ. Αλλά μπορείτε να κάνετε και άλλα πράγματα στον τομέα αυτό με άλλα επιγραμμικά εργαλεία που να επιτρέψουν την ενθάρρυνση των χωρών μελών ώστε να κάνουν περισσότερη χρήση του συστήματος. Και δεν είναι μόνο αξιωματούχοι τα πρόσφατα που το χρησιμοποιούν, αλλά και επιχειρήσεις και πολίτες εφόσον αντιληφθούν ότι έχουν τη δυνατότητα έτσι να αντλούν με ταχύτητα πληροφορίες και μπορούν βέβαια να έρθουν σε επαφή πρώτα με το σύστημα Solvit το οποίο με κάποιο τρόπο θα διασυνδέεται με το IMI. Σας ευχαριστώ. Αρχίζω με την ερώτηση του κ. Σφάπ που εντοπίζονται επί του παρόντος τα προβλήματα να αποσαφηνίσουμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο των πληροφοριών που ανταλλάσσεται στο σύστημα. Έχουμε στατιστικές μόνο ποιε συναλλαγές υπάρχουν σε ποιους τομείς. Ο λόγος είναι ότι οι συναλλαγές πληροφοριών αφορούν ατομικές περιπτώσεις και προσωπικά δεδομένα και όπως επεξήγησα στην αρχή μέσα στο σύστημα διασφαλίζουμε ότι μόνο εκείνοι οι οποίοι έχουν κάποιο συμφέρον, ένομο συμφέρον έχουν πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να επισημάνουμε ποια είναι η, ε, το όφελος όσον αφορά την ταχύτητα επαφών αλλά όχι το περιεχόμενο σε σχέση με τα προβλήματα τα οποία ταυτοποιήσαμε σε σχέση με τον κατάλογο των αρχών που είναι πραγματικά εντυπωσιακός υπάρχουν κάποιες χώρες όπου θα ανέμενε κανείς υψηλότερο αριθμό καταχώρησης όπου στην Ιταλία για παράδειγμα έχουμε 30 που έχουν καταχωρηθεί. Μπορεί να φαίνεται ότι επαρκεί, αλλά στην πρακτική εφαρμογή δεν επαρκεί, διότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία να διασφαλιστεί ότι όλε οι αρχέ που πρέπει να καταχωρηθούν σε περιφερειακό επίπεδο πράγματι καταχωρούνται. Είναι ένα θέμα στο οποίο συνεχίζουμε να προτρέπουμε τι Ιταλικέ αρχέ και να τι ενθαρρύνουμε, να τι πιέζουμε να ε, αυξήσουν τι ε, καταχωρήσει σε σχέση με την δυνατότητα καταγραφής τους, διότι αν δεν καταχωρούνται δεν μπορεί να ικανοποιηθεί η ανάγκη αυτή που υπάρχει στο σύστημα. Πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν ότι όλες οι αρχές θα έχουν ένα ρόλο να διαδραματίσουν σε αυτό το ε, επίπεδο. Αυτό με φέρνει στην παρατήρηση, παρατηρήσεις και ερωτήσεις του κυρίου Κορέα ε, Ντεκάμπος επιχειρηματίες και πολίτες δεν μπορούν να καταχωρηθούν στο σύστημα. Το IMI είναι ένα εργαλείο για επικοινωνία μεταξύ διοικητικών αρχών και θεσμών. Όμως σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχουν εμπορικά επιμελητήρια για παράδειγμα που έχουν κάποιο ρόλο να διαδραματίσουν όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας περί υπηρεσιών. Παράδειγμα για την καταχώρηση ε, τέτοιων επιχειρήσεων. Σε τέτοιες περιπτώσεις τα ε, εμπορικά επιμελητήρια καταχωρούνται και είναι χρήστες του IMI. Το IMI δεν είναι ανοιχτό σε απλούς πολίτες ως σύστημα. Αν διαβάσετε όμως την ανακοίνωση για την ε, δομή και ανάπτυξή του, εξετάζουμε την προοπτική να αναπτυχθεί ένα μέσο, ένα εργαλείο, να διασφαλίσει ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν τέτοια στοιχεία άμεσα στις αρχές, άμεσα μέσω IMI. Θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη για κάποιους τομείς πολιτικών να γίνεται αυτό για κάποια πεδία. Ο κύριος ε, Δεκάμπ ρώτησε αν οι ανταλλαγές αυτές είναι ενημερωτικές ή όχι. Όχι, δεν είναι ενημερωτικού χαρακτήρα. Οι αρχές ζητούν πληροφορίες όταν χρειάζονται αυτές τις πληροφορίες για μια συγκεκριμένη περίπτωση ή ανάγκη ως μέρο μήμα ενός, ε, του εποπτικού τους ρόλου ε, που έχουν να διαδραματίσουν, έχουν να διαμορφώσουν για παράδειγμα έλεγχο μιας ε, άδεια ε, λειτουργίας ε, εταιρεία που από την Πολωνία πολλούσε τα εμπορεύματά της στην Τσεχία ισχυρίστηκε ότι είχε μια διοδότηση ε, να ε, πολύ αυτά τα εμπορεύματα στην ε, Τσεχία όμως σε σχέση με τον έλεγχο που έγινε δεν πιστοποιήθηκε αυτό. Ήρθαμε σε επαφή με, τους, με την αρμόδια αρχή και απάντησαν ότι πράγματι ήταν μια πιστοποιημένη άδεια αυτή την οποία είχε. Αυτό δείχνει με υπό ποια μορφή μπορεί ο ρόλος ε, ε, υπό το πλαίσιο αυτής της ε, οδηγίας να υλοποιηθεί μεταξύ επικοινωνίας αρχών. Μια υποσημείωση τώρα σε σχέση με το σύστημα μετάφρασης στο IMI. Είναι ατυχές θα έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το μηχανικό σύστημα μετάφρασης που χρησιμοποιείται για την μετάφραση κειμένων έπρεπε να μην λειτουργήσει από το Δεκέμβριο πέρσι, να μην λειτουργεί λόγω νομολογίας ε, του δικαστηρίου, λόγω επίμαχων θεμάτων για τα πνευματικά δικαιώματα αυτής της ε, μηχανικής αυτόματης μετάφρασης. Τώρα έχουμε feedback, έχουμε παρατηρήσει από τους χρήστες ότι τους λείπει αυτό το μέσο, αυτό το εργαλείο και πρέπει να τεθεί πάλι στο διαδίκτυο διαθέσιμο όσο το δυνατόν πιο γοργά. Και εδώ έχουμε το πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να υποκατασταθεί αυτό και σε σχέση με το ε, Google για παράδειγμα όταν αφορώνται προσωπικά δεδομένα εργαζόμαστε πάρα πολύ στενά ε, με την ε, υπηρεσία για τις μεταφράσεις όσον αφορά το αυτόματο μηχανικό σύστημα μεταφράσεων και μας πρόσφεραν η δοκιμαστική μορφή αυτού του συστήματος να μπορέσει ίσως να αρχίσει να λειτουργεί τον Σεπτέμβριο του 2011. Δυστυχώς μέχρι τότε δεν θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται το μηχανικό το αυτόματο σύστημα μετάφρασης της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πράγμα που δεν σημαίνει ότι όλα αυτά έχουν εξαλειφθεί, έχουν εξαφανιστεί από το IMI, διότι έχουμε και προκαθορισμένα πρότυπα ερωτήσεων-απαντήσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως στοιχεία Τώρα για την κατάρτιση και την ε, προαγωγή, για την εκπαίδευση και προαγωγή προχωρούμε μεταξύ των κρατών μελών και τους ε, εμπλεκόμενους να δούμε γιατί υπάρχει τέτοια βραδία διάδοση του IMI και εφόσον θα έχουμε τα στοιχεία που θα εξηγούν αυτή την κατάσταση θα ε, δούμε ξανά το τι πρέπει να γίνει σε σχέση με την εκπαίδευση και την προαγωγή, την πρόθεση του συστήματος για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Επίσης ε, την δυνατότητα να μπορέσουμε να ε, καταλήξουμε σε ένα πολύ ευρύτερο ε, ε, κοινό, σε πολύ πιο πολυάριθμο κοινό που θα ενδιαφερθεί. Πρέπει να βρούμε τη σωστή μορφή προτύπου για την προαγωγή και την εκπαίδευση. Πρέπει όμως πρώτα να εντοπίσουμε τα πραγματικά προβλήματα και μετά να ακολουθηθεί από ένα πρόβλημα κατάρτισης, εκπαίδευσης που θα προσαρμόζεται στις ανάγκες για να επιληθούν αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ αν δεν υπάρχουν... Ναι, μια τελευταία ερώτηση από εσάς παρακαλώ. Ε, μικρόφωνο. Ε, ήθελα να ρωτήσω... Κυρία Ράπτη παρακαλώ. Ε, στο δίκτυο αυτό μπορούν να εγγράφονται συνδικαλιστικές οργανώσεις. Νομίζω ετέθη το ερώτημα αυτό. Τι εννοώ, για παράδειγμα, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών, που είναι το όργανο που εκφράζει τις βιομηχανίες ή η ΑΔΕΔΗ. Ε, μιλάω για την πραγματικότητα της Ελλάδας, αλλά μπορεί προφανώς να συμβαίνει και σε άλλα κράτη. Ε, η ΑΔΕΔΗ που είναι το όργανο που εκφράζει το συνδικαλιστικό όργανο των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι ε, δημόσιοι υπάλληλοι αποτελούν μέρος της διοίκησης, μέλη της διοίκησης που ζητούν πληροφορίες. Αυτοί όλοι μπορούν να είναι μέσα στο δίκτυο ή όχι. Um, Ευχαριστώ κύριε Ράπτη. Παρακαλώ. Οι χώρες μέλη, οι χώρες μέλη θα αποφασίσουν ποιον θα εγγράψουν, ποιον θα καταχωρήσουν ως αρμόδιο στο σύστημα. Καμία αρχή δεν αποκλείεται. Εάν μια χώρα μέλος θεωρήσει ότι ένα συνδικάτο έχει ένα ρόλο να παίξει, για παράδειγμα για την εφαρμογή της ε, οδηγίας περί μπορεί να αποφασίσει η χώρα μέλος να καταχωρήσει αυτόν τον φορέα, έστω και αν είναι συνδικάτο. Υπάρχει λοιπόν πλήρης ευκαμψία από πλευράς μας υπέρ των χωρών μελών να αποφασίζουν. Αυτό βέβαια θα έχει σχέση αν αρχίσει να μπαίνει θέμα και απόσπαση εργαζομένων. Σας ευχαριστώ πολύ πάντως, καθώς και την ομάδα σας και επιθυμώ, ελπίζω ακόμη να μας παρακολουθούν όσοι εργάζονται για το σύστημα IMI στις χώρες μέλη. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι υποστηρίζουμε την προσπάθεια. Αναμένουμε με ενδιαφέρον λοιπόν την περαιτέρω συνεργασία αλλά και την διαβίβαση της επίσημης νομοθετικής σας προτάσεως αργότερα μέσα στο έτος και οι συντονιστές θα εξετάσουν να δουν εάν μπορούν την κοινοποίησή σας να την περιλάβουμε σε κάποια από τις πρωτοβουλίες μας για την ενιαία αγορά. Βεβαίως εμείς έχουμε διαρκώς ιδέες για το πώς μπορούμε να συμβάλλουμε, να συνεισφέρουμε. Έχουμε και τα βαθμολόγια που εξετάζουμε για την ώρα, αλλά μπορούμε ίσως να τα συνδυάσουμε με την έκθεσή σας. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και πάλι. Έχω τώρα λίγες ανακοινώσεις πριν κηρύξω τη λήξη της σας. Ξαναβρισκόμαστε αύριο το πρωί στις 9 εδώ. Μία μικρή αλλαγή στην ημερήσια διάταξη της αύριο. Το πρώτο θέμα θα είναι η έκθεση Ρόιτεβα για το Deposit Guarantee Schemes στις 9. Μετά θα ακολουθήσει η έκθεση του κυρίου Παντζέρη και του, μετά του κυρίου Σαλβίνη στις 10 και 4 θα ψηφίσουμε. Μετά θα έρθει ο Αντιπρόεδρος Επιτροπής κ. Σταγιάννη στις 11.30 να μιλήσει για το μελλοντικό πρόγραμμα εργασιών του και θέλει να μας θέσει υπόψη ορισμένα σημαντικά θέματα, μεταξύ των οποίων και την τυποποίηση. Μετά θα ακολουθήσουν 3 έως 4.30 συντονιστές και 4.30 έως 6.30 σημαντική ακρόαση που θα διευθύνει ο κ. Βαντεκάμπ εισηγητή για, τη νέα, για τους κανονισμούς εγκρίσεως δικύκλων και τρικύκλων οχημάτων. Και θα έχουμε και ε, να μας παρακολουθούν και ειδικευμένος τύπος ε, ε, που ασχολείται με τα οχήματα αυτά και βεβαίως θα είναι σημαντικό να τους δείξουμε πόσο πολύ μας ενδιαφέρει το θέμα. Σας ευχαριστώ όλες και όλους. Ευχαριστούμε και τους, ε, τα πρόσωπα που μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο και θα σας αναμείνω όλους αύριο το πρωί.